Ονομάζομαι Τσέσο Σεκέρσκι και ως πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας θα έχω τη χαρά να προεδρεύσω στη σημερινή αυτή συνάντηση. Να με συμπαθάτε για την κάπως απότομη έναρξη, αλλά σκέφτηκα να ξεκινήσουμε όσο πιο νωρίς γίνεται για να έχουμε περισσότερο χρόνο για τη συζήτηση. Με, με ιδιαίτερη χαρά θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην ε, συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια και κυρίως ε, με εθνικούς βουλευτές που ασχολούνται κυρίως με γεωργικά ζητήματα, τρόφιμα και αγροτική ανάπτυξη. Σας ε, καλωσορίζω θερμότατα σε αυτή την κοινή μας συνεδρίαση. Σας ζητώ εκ των προτέρων συγγνώμη για κάποια ταλαιπωρία ενδεχομένω που υποστήκατε. Ελπίζω να μην ήταν πολύ σημαντική. Όπως ξέρετε, το θέμα της σημερινής συζήτησης ε, είναι τα τρόφιμα, το μέλλον το τρό... της γεωργίας και των τροφίμων. Δεν ε, θα επεκταθώ. Γνωρίζουμε το αντικείμενο της συνάντησης. Έχουμε τις τελευταίες εξελίξεις, την ανακοίνωση του, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, του Νοεμβρίου Επίσης αναμένουμε ε, στα ε, αυτό το τέλη Νοεμβρίου. Αναμένουμε στα τέλη του Μαΐου την, ε, την πρόταση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και το νομοθετικό πακέτο για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ μετά το 2020. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στη σημερινή μας συνάντηση και θα ήθελα εκ μέρους όλων μας να καλωσορίσω, να καλωσορίσω τον Φιλ ε, Χόγκαν, τον αρμόδιο επίτροπο για τα θέματα που μας ενδιαφέρουν. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έχει την καλοσύνη να έρθει εδώ ο Επίτροπος. Και έχουμε εδώ και τον κύριο Ρούμεν Ποροτζάνοφ, τον Βούλγαρο Υπουργό Γεωργίας, Τροφίμων και Δασοκομείας, που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου αυτή τη στιγμή. Και είναι και ο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλίας. Επίσης ε, βρίσκεται εδώ και ο κύριος Γιώζεφ Πλάνκ, Γενικός Γραμματέας ε, στο Αυστριακό Υπουργείο Βιωσιμότητας και Τουρισμού. Χαιρόμαστε ιδιαίτερος ε, για την παρουσία και του Αυστριακού εκπρόσωπου, γιατί η Αυστρία θα αναλάβει την Προεδρία αμέσως μετά τη Βουλγαρία, στο δεύτερο εξάμεινο του 2018. Και στη συνέχεια θα έχουμε συζήτηση με δύο πάνελ ε, θα μας μιλήσει στο πρώτο πάνελ ο κ. Παντέρινγκ, ε, που είναι πρόεδρος της ε, κοινή Επιτροπής Γεωργίας Τροφίμων και Θάλασσας από την Ιρλανδία. Θα μας μιλήσει ο κ. Χέρμπερ Ντόρφμαν, Ιταλός βουλευτής, που είναι ο εισηγητής μας για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η κυρία Αγγιλέρα, που είναι αντιπρόεδρος Επιτροπής Γεωργίας. Επίσης, θα έχουμε και τον Γενικό Διευθυντή της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, τον κύριο Γέζη Πλέβα, που θα μας μιλήσει για τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά νομίζω ότι οι καλεσμένοι μας θα σας ενημερώσουν πολύ καλύτερα από μένα. Γι' αυτό δεν θα επεκταθώ άλλο. Τώρα, ως προς τα διαδικαστικά, έχετε δύο έντυπα με διαφορετικά χρώματα για να ζητάτε το λόγο για το πρώτο ή το δεύτερο πάνελ. Παρακαλώ συμπληρώστε τα. Δώστε τα στους κλητήρες και η γραμματεία θα προσπαθήσει να καταρτήσει κατάλογο αγοριτών όσο πιο ευρύ γίνεται, ώστε να συμμετέχουν οι πρόσωποι όλων των χωρών, ε, ευρωβουλευτές και όσοι επιθυμούν να λάβουν το λόγο. Ο χρόνος ε, είναι πολύτιμος Γι' αυτό θα διακόψω εδώ και θα περάσουμε στον πρώτο καλεσμένο μας, την πρώτη παρουσίαση που θα γίνει από τον Επίτροπο Φιλ Χόγκαν και τον Υπουργό Ποροτζάνοφ από τη Βουλγαρία. Περιμένουμε με ανυπομονησία τις ομιλίες σας για να κατατοπιστούμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γεωργία και τις λύσεις που προτείνουμε. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον Επίτροπο Φιλ Χόγκαν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, αγαπητοί προσκεκλημένοι. Κυρίε και κύριοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο τη Επιτροπή Γεωργία, τον κύριο Σερκεύσκη, για την ε, πρόσκληση να συμμετάσχω στη σημερινή ε, διακοινοβουλευτική ε, διάσκεψη. Είναι πολύ σημαντική η συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια και αποτελεί προτεραιότητα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκτιμάται ότι τα μέλη αυτού του σώματος, δηλαδή των Εθνικών Κοινοβουλίων, έχουν, ε, συγγνώμη, του Κολεγίου των Επιτρόπων έχουν κάνει πάνω από 470 επισκέψεις σε Εθνικά Κοινοβούλια στα 28 κράτη-μέλη. Ε, προσωπικά έχω επισκεφθεί πάνω από 20 Εθνικά Κοινοβούλια. Την προηγούμενη εβδομάδα συμμετείχα στη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με την συνεργασία ακριβώ με τα εθνικά κοινοβούλια, του μηχανισμού που έχουμε στη διάθεσή μα για αυτό και πώ μπορούν να βελτιωθούν. Και στην ομιλία μου είπα ότι τα εθνικά κοινοβόλια παίζουν και θα συνεχίζουν να διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έρχεται κοντά στους πολίτες έτσι ώστε να ασκείται έλεγχος από τους πολίτες στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ε, και τις ε, διεργασίες που γίνονται σε αυτά. Και θα έλεγα ότι η σημερινή διακοινοβουλευτική συνάντηση μας δίνει μια πολύ καλή ευκαιρία να το κάνουμε αυτό στην πράξη, γιατί έχετε τη δυνατότητα να συζητήσετε με τους συναδέλφους σας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλοι μαζί να δώσετε ε, προτάσεις και παρατηρήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς εκείνη προετοιμάζει τις νομοθετικές της προτάσεις για το μέλλον της Γεωργίας μετά το 2020. Γνωρίζετε ως ε, αυτή τη ε, στιγμή έχουμε την ανακοίνωση του Νοεμβρίου για το μέλλον της, ε, της ΚΑΠ και έχουμε επίσης και την πολύ καλή συνεργασία με τον φίλο μου, τον κύριο Ρούμεν νόφ, υπουργό Γεωργίας της Βουλγαρίας που έχει αυτή τη στιγμή την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα ήθελα επίσης να εξάρω τον ρόλο των εισηγητών και των σκιωδών εισηγητών που έχουν προετοιμάσει τις διάφορες νομοδοτήσεις που μας υποβάλλει η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γνωρίζω ότι τον επόμενο μήνα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα υπάρξει και ψήφισμα σε σχέση με την ανακοίνωση της Επιτροπής που σας ανέφερα. Τους επόμενους δύο μήνες θα ε, έχουμε πολλά γεγονότα σε σχέση με το μέλλον της γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα, την επόμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή τον γενικό προπολογισμό μετά το 2020. Δεν πρέπει να έχουμε αυτά αυταπάτες. Όταν έχουμε το Brexit, όταν έχουμε την αποχώρηση ε, ενός, μιας χώρας που εισφέρει, ε, θα είναι περιορισμένοι οι πόροι. Όμως, θα πρέπει να συζητηθεί και τελικά είναι στα χέρια των ηγετών των κρατών μελών να δούμε αν θα επιθυμούν και αν θα αποφασίσουν τελικά να αυξήσουν τις συνεισφορές τους. Βεβαίως τον, όλο, όλο τον επόμενο χρόνο θα έχουμε μια ολόκληρη διαδικασία για τη συζήτηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Εσείς ως μέλη των αρμοδίων επιτροπών στα Εθνικά Κοινοβούλια, των αρμοδίων για τη Γεωργία, ε, είμαι σίγουρος ότι συμφωνείτε μαζί μου. Ότι πρέπει να έχουμε μια κοινή αγροτική πολιτική η οποία να έχει ουσιαστικούς όρους, η οποία να είναι σωστά χρηματοδοτημένη και η οποία να συνεισφέρει και στη Γεωργία και στην, στην ε, βελτίωση των συνθήκων στις αγροτικές περιοχές, καθώς επίσης και τους περιβαλλοντικούς μας στόχους, όπως για παράδειγμα η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ε, ε, εγώ εκπροσωπούσα μια αγροτική περιοχή στο, στο Ιρλανδικό Κοινοβούλιο εδώ και 27 χρόνια και γνωρίζω ότι η ΚΑΠΑ από το 1962 έχει αποδείξει την αξία της, έχει ε, αντέξει στο χρόνο και είναι πολύ σημαντική και συνεχίζει να είναι πολύ σημαντική για ε, εκατομμύρια πολίτες στην Ευρώπη. Όταν λοιπόν ως βουλευτές απαιτούμε μια ισχυρή ΚΑΠ, μπορείτε και σας ζητώ να απευθυνθείτε στις εθνικές σας κυβερνήσεις και να επισημάνετε Σπάνια βλέπω τη συνάδελφο Σόιχλ να χειροκροτεί τις ομιλίες μου. Χαίρομαι γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι αμφισβητούν τη σημασία της ΚΑΠ και η απάντησή μου σε αυτούς είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε το χρέος μας να υποστηρίζουμε τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους. Αποτελεί εξάλλου και στοιχείο των ε, συνθήκων ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτός ο στόχος παραμένει επίκαιρος όσο, όσο ποτέ. Και αυτό θα φανεί και στις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα υπενθυμίσω κάτι που αναφέρεται στην ανακοίνωση της σχετική της Επιτροπής. Είναι ξεκάθαρο για μας ότι παραμένει θεμελιώδους σημασίας η υποστήριξη του αγροτικού εισοδήματος. Γνωρίζουμε ότι οι άμεσες πληρωμές μόνο εν μέρη λύνουν το πρόβλημα, μόνο εν μέρη καλύπτουν το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στο αγροτικό εισόδημα και το εισόδημα σε άλλες περιοχές σε άλλους τομείς της οικονομίας ε, και πρέπει να παρέμβουμε και επίσης προς την κατεύθυνση της αγροτικής ε, ανάπτυξης. Γιατί η ανάπτυξη της περιφέρειας έχει μεγάλη σημασία κοινωνική για την κοινωνική συνοχή και για αυτόν τον λόγο λοιπόν οι άμεσες πληρωμέ θα παραμείνουν μια, ένα σημαντικό στοιχείο της νέας ΚΑΠ σύμφωνα με βέβαια τι τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συνθήκες. Ε, αυτό δεν το κάνουμε μόνο για να βοηθήσουμε τους αγρότες, αλλά για να βοηθήσουμε την κοινωνία συνολικά. Οι αγρότες είναι πρώτα απ' όλα εκείνοι που παράγουν την τροφή μας και θέλουμε αυτή να είναι υψηλής ποιότητας, αλλά επίσης βρίσκονται στην ύπεθρο και άρα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προστασίας του περιβάλλοντος ε, και είναι οι πρώτοι που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή. Ε, στην προσπάθεια μας αυτή να προστατεύσουμε το εισόδημα το αγροτικό. Χαίρομαι που διαπιστώνω ότι έχω την υποστήριξη και του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου αλλά και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γνωρίζω από τους Υπουργούς, από τον Υπουργό Αποσδόροφ. Γνωρίζω επίσης ότι το ζήτημα αυτό σας απασχολεί ουσιαστικά και είναι στην καρδιά σας και για πολλούς από εσά στα Εθνικά Κοινοβούλια. Και θα τη χρειαστώ αυτή είναι η βοήθειά σας γιατί θα είναι δύσκολες οι συζητήσει για τον προϋπολογισμό τις επόμενες εβδομάδες και μήνες μετά από τη γενική πρόταση πλαίσιο για το πολιτές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο, η Επιτροπή θα παρουσιάσει ε, το, στις αρχές ε, Ιουνίου τις τομεακές προτάσεις. Και θα ξεκινήσει η σχετική συζήτηση. Το, αυτό που μπορώ ήδη βέβαια να σας πω είναι ότι η τομεακή πρόταση για την αγροτική οικονομία, για την, για την ΚΑΠ, θα είναι πλήρως συμβατή με την ανακοίνωση που κάναμε ως Επιτροπή τον Νοέμβριο. Θέλουμε να καταλήξουμε σε μια λύση δηλαδή η οποία θα γίνει ε, ευρέως αποδεκτή και θα υποστηριχθεί. Ε, αντιλαμβάνομαι ότι αυξάνεται η υποστήριξη σε αυτή την προσέγγιση ε, και είχαμε τη δυνατότητα τις, τους μήνες που ακολούθησαν μετά την ανακοίνωση να εξηγήσουμε καλύτερα και ποιες είναι οι επιδιώξεις μας και η προτεραιότητάς μας ως Επιτροπή γιατί σε μια ανακοίνωση μας έχουμε και τον περιορισμό του, του, της έκτασης για την Επιτροπή συνεχίζει να είναι πολύ σημαντική ε, η αρχή της επικουρικότητας και αυτό σημαίνει ότι οι περιφέρειες θα πρέπει να συνεχίσουν να αναλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερη ε, ευθύνη. Ε, με άλλα λόγια, οι αποφάσεις να λαμβάνονται πιο κοντά στον πολίτη. Αυτό είναι γενικό ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι έχουμε απεμπολίσει τον ουσιαστικό ρόλο που πάντα έπαιζε και θα παίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην κοινή αγροτική πολιτική. Η κοινή αγροτική πολιτική θα συνεχίσει να βρίσκεται στο ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό που θα χρειαστεί θα είναι μεγαλύτερη ευηλιξία στην εφαρμογή τη στο επίπεδο των κρατών μελών. Γιατί γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε σε 28 κρατημέλη να εφαρμόσουμε το ίδιο μοντέλο. Ε, είναι κάτι πολύ διαφορετικό η κατάσταση ε, για του Έλληνε αγρότε στον Νότο με του Φινλανδού αγρότε στο Βορρά. Θα έχουν μια διαφορετική προσέγγιση, μια διαφορετική νοοτροπία, διαφορετικέ επίση μεθόδου για να επιτύχουν παρόμοιου στόχους. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε και να το λάβουμε υπόψη μα. Έτσι ερχόμαστε στα εθνικά στρατηγικά σχέδια για την κοινή αγροτική πολιτική που εσείς στα κράτη-μέλη θα καταρτήσετε, η Βουλή, το Εθνικό Κοινοβούλιο κάθε χώρα θα παίξει ρόλο σε αυτή την κατάρτιση ε, συνεργαζόμενοι και ασκώντας έλεγχο κοινοβουλευτικό στον ε, αρμόδιο υπουργό της χώρας σας πριν η κυβέρνηση της χώρας σας υποβάλει το σχετικό στρατηγικό σχέδιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν ε, θα αξιολογεί αυτά τα σχέδια με βάση τους γενικούς στόχους που έχουμε θέσει στο ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να υπάρχει μια γενικότερη συνεκτικότητα. Ε, σε κάποιες χώρες έχουν υπάρξει ανησυχίε σε σχέση με αυτά τα στρατηγικά σχέδια. Όσες, εκπρόσωποι των πολιτών γνωρίζετε ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να μην καθυστερήσουν οι άμεσες πληρωμές στους αγρότες εξαιτίας μιας κάποιας καθυστέρησης της ΚΑΠ. Ένας τρόπος είναι αυτή η χάραξη πολιτικής μέσω αυτού του συστήματος που σας περιέγραψα. Θα δώσουμε τη δυνατότητα μέσω αυτών των στρατηγικών σχεδίων των κρατών μελών να μην υπάρξει ε, διακοπή στις ε, πληρωμές των αγροτών ακόμα και αν ε, στο πλαίσιο της συζήτησης με την Επιτροπή συζητώνται κάποια άλλα θέματα κάποια στιγμή. Πιστεύω ότι μπορούμε να είστε υπερήφανοι για το ρόλο που έχει δραματίσει η κοινή γεωργική πολιτική το τελευταίο, τα τελευταία 50 χρόνια, γιατί εξασφάλισε και ε, πιστιστική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά πέραν αυτό και για την ανάπτυξη και την αποδοχή του ευρωπαϊκού εγχειρήματο χάρη στην ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική. Είναι η επιτυχία της, ε, μια επιτυχία που οφείλεται πάνω απ' όλα στους γεωργούς και σημαίνει ότι μπορεί να προσαρμόζεται και στις ε, νέες προκλήσεις. Ωστόσο, εξαρτάται αυτή η επιτυχία και από μια καλά λειτουργούσα ιστορική αγορά για τη γεωργία. Και πρέπει να την προστατεύσουμε αυτή την ιστορική αγορά. Και ο κύριο Ντόρφμαν, ο εισηγητή στην έκθεσή του, πολύ εύγλωτα επεσήμανε αυτέ τι αρχέ τον είπε ότι η ακαιρεότητα τη εσωτερική αγορά και μια εσωτερική, πραγματική εσωτερική κοινή πολιτική πρέπει να είναι κύριε προτεραιότητά μα. Αυτό θέλω να υπογραμμίσω και εγώ με μια νέα προσέγγιση μεν ω προ την υλοποίηση τη πολιτική, δεν αλλάζει ο θεμελιωδό κοινό χαρακτήρα τη κοινή γεωργική πολιτική και πρέπει να συνεχίσει αυτή να είναι μια πολιτική που θα αντιμετωπίζει μια σειρά από ζητήματα, από κοινού στόχου που θα προσμετρώνται με αναφορά σε ένα ευρύτερο σύνολο κοινών δικτών που θα υπάγονται σε ένα κοινό σύστημα έγκριση με τον έλεγχο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την ακαιρεότητα λοιπόν τη ιστορική αγορά και την εξασφάλιση ενό ότιμου πεδίου ανταγωνισμού και λειτουργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρε, ξέρω ότι έχω καθυστερήσει αρκετά στον χρόνο μου, θα επιταχύνω λοιπόν ε, την ομιλία μου έχουν ε, θεωρηθεί για πολύ καιρό δυστυχώς οι γεωργοί κομμάτι ενός περιβαλλοντικού προβλήματος ενώ θα έπρεπε να θεωρηθούν περισσότερο ως κομμάτι της λύσης του προβλήματος αυτού. Για να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις, ε, τα αποτελέσματα της οικολογικοποίησης που δεν έχει φέρει τους αναμενόμενους καρπούς. Θα ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη λοιπόν για άλλη μια φορά να μας υποβάλουν προτάσεις ε, για το εθνικό πάντα σχέδιο που θα δώσουν απαντήσεις στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Και έτσι θα έχουμε και λιγότερη γραφειοκρατία και καλύτερη στόχευση στο τοπικό επίπεδο των στόχων και πιο αποτελεσματική υλοποίηση, ταχεία υλοποίηση, ενσωμάτωση των μέσων που είναι διαθέσιμα στις ε, εφαρμογές. Ξέρω ότι έχετε συχνά επικοινωνία με τους νέους και ότι γνωρίζετε ότι πολλοί από αυτούς ενδιαφέρονται ή σκέφτονται τουλάχιστον να ξεκινήσουν μια γεωργική δραστηριότητα. Ταυτόχρονα φαντάζομαι θα γνωρίζετε και πόσο οι δυσφορία αισθάνονται γιατί είναι πολλοί αυτού ε, Έχοντα υπόψη αυτή τη δυσφορία, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διατεθειμένη να αναλάβει το δικό τη κομμάτι τη ευθύνη και, και τι θεωρούμε ότι είναι μια ευθύνη κοινή με τα κράτη-μέλη, να διευκολύνει με μέτρα και μέσα ε, όπου έχει την αρμοδιότητα αυτή τη δραστηριότητα. Έτσι λοιπόν ε, στηρίζομαι και στη δική σας την υποστήριξη για τα νέα μας σχέδια. Έχουμε να κάνουμε με μια πρωτοβουλία για το έξυπνο χωριό το οποίο η οποία ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο. Ένα πολύ ενδιαφέρον έργο, ένα συναρπαστικό έργο που σημαίνει ότι δίνονται πρακτικές λύσεις σε χωριά στην ε, Ήπεθρο για την εξασφάλιση καλύτερων και νέων ευκαιριών και είδαμε ότι ήδη στη Σλοβενία ξεκίνησε ένα πιλωτικό σχέδιο για την ανάπτυξη έξυπνων οικολογικών και κοινωνικών χωριών όπου μπορούν να βελτιώσουν χάρη στο έργο αυτό οι τοπικές κοινότητες τις συνθήκες τους. Θέλω να ευχαριστήσω τους, ευ... τον Ευρωβουλευτή, τους Ευρωβουλευτές Μπόκοβιτς και Σιάννη, οι οποίοι με την, με τον ενθουσιώδη, με την ενθουσιώδη υποστήριξή τους εξασφάλισαν 3,3 εκατομμύρια για μια προπαρασκευαστική δράση που θα ξεκινήσει από το 2019. Ε, αυτή τη στιγμή δίνουμε υποστήριξη σε 10 έξυπνα χαρτιά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσεί ω εθνικοί βουλευτέ πρέπει να βοηθήσετε ώστε να μην μείνει κανένα κράτο μέλο ε, αποκλεισμένο από αυτό το τεράστιο δυναμικό. Δεν θέλω να ολοκληρώσω επαναλαμβάνοντα ότι η ελπίδα μα είναι να εξασφαλίσουμε τα μέγιστα δυνατά ε, αποτελέσματα για τους ε, πολύ καλούς στόχους που έχουμε ορίσει για τους γεωργούς και τον παραγωγό των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολιτική είναι μια κοινή γεωργική πολιτική για όλο το μέλλον, για όλους τους λαούς της Ευρώπης, για ολόκληρη την Ευρώπη, για όλους τους Ευρωπαίους, για να έχουμε μια καλή πολιτική γεωργίας, πολιτική τροφίμων. Πιστεύω ότι τους επόμενους μήνες θα έχουμε καλά αποτελέσματα προς όφελος όλων των πολιτών της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Πίτροπε. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον Βούλγαρο Υπουργό Ποροτζάνοφ για 10 λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, συντονιστές των πολιτικών ομάδων, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ και αξιότιμοι βουλευτέ από τα Εθνικά Κοινοβούλια, κύριε Επιτροπέ, κυρίες και κύριοι. Θα είμαι πολύ σύντομος, θα χρειαστεί καν να εξαντλήσω το δεκάλεπτο, γιατί ο Επίτροπος ε, μίλησε διεξοδικά για τις προσπάθειες που γίνονται και όλα όσα μας ανέφερε είναι αντικείμενο συζήτησης και στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας φέτος. Η Βουλγαρική Προεδρία τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο διοργάνωσε συζητήσεις γύρω από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας. Μίλησαμε για τις προτεραιότητες, ε, τις άμεσες ενισχύσεις, ε, ε, τον εξορθολογισμό της σύγκλησης, την επικουρικότητα και πολλούς άλλους τομείς, τις πράσινες οικολογικές πληρωμές και ούτω καθεξής. Οι συνεδριάσεις αυτές ήταν δημόσιες και μάλιστα παρακολουθήθηκαν από ευρύ κοινό, όχι μόνο από γεωργούς, αλλά και γενικώ από την κοινή γνώμη. Γιατί η γεωργική πολιτική δεν περιορίζεται μόνο στη γεωργία. Και μάλιστα με την ολοκλήρωση τη συζήτηση τον Μάρτιο καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα, κάτι που δεν ήταν διόλου εύκολο. Τελικά τα συμπεράσματα αυτά εγκρίθηκαν από 23 χώρες μέλη και 5 χώρες διαφώνησαν με ένα μόνο σημείο αυτών των συμπερασμάτων. το θέμα της σύγκλησης ε, ή της εναρμόνισης των επιπέδων στραματικής ενίσχυσης. Αυτά τα συμπεράσματα είναι γνωστά σε όλους και είναι αναμφίβολο ότι το μήνυμα του Συμβουλίου Υπουργών θα βοηθήσει και τον Επίτροπο Χόγκαν και τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας κατά την προετοιμασία του νέου νομοθετικού πακέτου για την μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής μετά το 2020. Όλοι περιμένουμε με ανυπομονησία αυτό το πακέτο και τον Ιούνιο το Συμβούλιο Υπουργών θα ξεκινήσει τη συζήτηση επί των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και μάλιστα το σχέδιο έκθεσης που εκπονεί η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πλησιάζει τη συζητήσει στο Συμβούλιο. Και συμβαδίζει με αυτά που είπαμε εκεί. Σε κάθε συνάντηση έχουμε διαβούλευση και με την Κόπα Κοζέκα, τη μεγαλύτερη οργάνωση αγροτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα συμπεράσματά μας λαμβάνουμε υπόψη και τις δικές τους θέσεις. Πάντως όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα ξεκάθαρο όραμα για τη νέα κοινή γεωργική πολιτική. Γι' αυτό και θα πρέπει να συνεχίσουμε τις αργότερες προσπάθειες και εμείς, η Βουλγαρική Προεδρία, αλλά και η επόμενη Προεδρία, η Αυστριακή, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για την απλούστευση της κοινή γεωργικής πολιτικής και για τη συγκεκριμενοποίηση πολλών θεμάτων που τώρα είναι κάπως γενικά, αλλά στην πορεία θα συγκεκριμενοποιηθούν. Και ευελπιστώ ότι θα φέρουμε σε αίσιο πέρας και τη δική μας Προεδρία και η Αυστριακή Προεδρία θα συνεχίσει την δική της θετική προσπάθεια και ελπίζω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας στηρίξει. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται να εγκρίνει την, το νέο νομοθετικό πακέτο κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας και να εξασφαλίσει ένα σταθερό μέλλον για τους Γεωργούς. Περιμένουμε επίσης ε, με αδημονία την πρόταση για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, και ξέρω ότι ο Φιλ Χόγκαν θα κάνει ό,τι μπορεί, θα βάλει τα δυνατά του για να διασφαλίσει ένα καλό γεωρικό προϋπολογισμό μέσα στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Πάντως το κοινό μας μήνυμα είναι να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση στην κοινή γεωρική πολιτική για να μπορέσει να εφαρμοστεί και κατάλληλα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και προσβλέπω σε πολύ επικοδομητική καρποφόρα συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής σα και τους Εθνικούς Βουλευτές. Θα ήθελα και εγώ να σα ευχαριστήσω κύριε Υπουργέ. Και τώρα θα ε, ζητούσα από τον κύριο Σιμών να έρθει να λάβει θέση στο Προεδρείο για να συντονίσει το πρώτο πάνελ. Το πρώτο πάνελ λοιπόν θα συντονιστεί από τον κύριο Σάιμον που έχει και πέντε λεπτά στη διάθεσή του για να κάνει την εισαγωγή και μετά θα ακούσουμε τον κύριο Ντόρφαν που είναι ο εισηγητής της έκθεσης για την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κατόπιν θα μιλήσει ο κύριος Πλάνκ, ο Γενικός Γραμματέας του Αυστριακού Υπουργείου Βιωσιμότητας και Τουρισμού Ο κύριο Σάμαν έχει το λόγο. Πέντε λεπτά για εσά και μετά οι δύο καλεσμένοι του πρώτου πάνελ. Καλημέρα σας. Τώρα που κάθισα θα ήθελα εν συντομία να σας κάνω μια επισκόπηση που το πολιτικό του σκέλος το παρουσίασαν ο Επίτροπος και ο Βουλγαρός Υπουργό και θα σας αναφέρω και το χρονοδιάγραμμα. Στις 2 Μαΐου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει το σχέδιο πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου που φυσικά θα πρέπει να λάβει υπόψη το χρηματοδοτικό κενό των 12 δισεκατομμυρίων στον ενωσιακό προπολογισμό. Το χρηματοδοτικό κενό που δημιουργείται από την αποχώρηση τη Μεγάλη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να λάβει υπόψη και τι νέε προτεραιότητε, την ασφάλεια, τη μετανάστευση και την άμυνα. Με βάση τι νέε αδιακρίσει που κυκλοφορούν στι Βρυξέλλε, ε, ε, τι φήμε, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προτείνει την επόμενη εβδομάδα μείωση κατά 6% των γεωργικών δαπανών καθώς και των κονδυλίων της συνοχής και των διαρθρωτικών ταμείων. Στην δημοσιονομική συζήτηση λοιπόν που θα γίνει, ο Επίτροπος ε, Φιλ Χόγκαν δήλωσε πρόσφατα στις 20 Απριλίου ότι θέλει να προστατεύσει τους μικρούς γεωργούς και αυτή είναι η βασική του προτεραιότητα στις δημοσιονομικές διαπραγματεύσεις. Εν συνεχεία, σε ό,τι αφορά την γενική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον των τροφίμων και της ε, γεωργίας ε, της 29ης ε, παρελθόντος Νοεμβρίου. Εκεί αναφέρεται στην επικουρικότητα, ώστε στη θεωρία τουλάχιστον να πλουστευτεί η ΚΑΠ. Επικουρικότητα σημαίνει ότι ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων θα ενισχυθεί. Και αυτό θα είναι το αντικείμενο του δεύτερου πάνελ της συζήτησης. Δεύτερον, η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτείνει μια νέα οικολογική αρχιτεκτονική. Δηλαδή μια νέα υποχρεωτική αιρεσιμότητα που θα απορροφά το, τις τωρινές προτάσεις της οικολογικοποίησης και θα περιλαμβάνει και ένα επιπλέον στρώμα που θα είναι προαιρετικό για τα κράτη-μέλη, ένα επιπλέον εκούσιο επίπεδο που θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη που θέλουν να είναι πιο φιλόδοξα να το κάνουν. Και μάλιστα η ανακοίνωση αυτή έχει γίνει δεκτή από το Συμβούλιο. Και την Παρασκευή, την επόμενη Παρασκευή, ε, θα υποβληθεί στους Προέδρους ε, Επαγγελματικών Οργανώσεων και Γεωργικών Συνεταιρισμών της Ευρώπης, την ΚΟΠΑ ΚΟΖΕΚΑ, που θα δηλώσουν ότι η ανακοίνωση είναι καλή βάση για τη συζήτηση υπό δύο προϋποθέσεις. Ότι δηλαδή δεν θα οδηγήσει σε κατακαιρματισμό της εφαρμογής της κοινή γεωργικής πολιτικής, πρώτον, και δεύτερον, θα οδηγεί σε πραγματική απλοποίηση της ΚΑΠ για τους γεωργούς, κάτι που δεν είναι δεδομένο. Δεύτερον, το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο έχει δεχτεί γενικώ θετικά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιορίζεται στην απαρίθμηση κάποιων γενικών αρχών, αλλά και στο Συμβούλιο κάποιοι υπουργοί εξέφρασαν την ε, ανησυχία τους για το πιθανό κατατεμαχισμό της εφαρμογής της κοινή γεωρικής πολιτικής και την πιθανή στρέβλωση ανταγωνισμού που κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει. Και δεύτερον, ένα πολιτικό θέμα. Η εξίσωση των θερματικών ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών είναι ένα καθόδε ζήτημα. Η σύγκληση των ενισχύσεων. Βέβαια αυτό δεν είναι τόσο αρμοδιότητα των Υπουργών Γεωργίας, αλλά περισσότερο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, γιατί αυτοί θα προσδιορίσουν τα εθνικά κονδύλια για την κοινή γεωργική πολιτική ένα θέτο χρόνο. Τέλος, η έκθεση του κύριου Ντόρφμαν, που αφορά την ανακοίνωση του Νοεμβρίου και που θα εγκριθεί στην Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συνεδρίαση της 16ης και 17ης Μαΐου. Επίσης, 29 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει τις ε, κλαδικές της νομοθετικές προτάσεις ε, στο επόμενο ΠΔΕΛΤΑΠΗ για την κοινή γεωργική πολιτική. Θα υποβάλει τρεις προτάσεις. Η πιο ε, γενική θα αφορά τις λεπτομέρειες των ε, ενισχύσεων της ΚΑΠ, το σχέδιο στήριξης ε, ΚΑΠ, που θα πρέπει να εκπονείται από κάθε κράτος μέλος στα πλαίσια αυτής της επικουρικότητας. Το σχέδιο στήριξης των μέτρων της ΚΑΠ. Δεύτερον, με βάση αυτά που κυκλοφορούν, είναι ότι η γεωργικές υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί το κείμενο αυτό συστάται γενικά τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να προβλέψουν ε, ε, για τους μικρούς ε, καλλιεργητές ένα ανώτατο όριο των ενισχύσεων αναεκμετάλλευση. 60.000 ευρώ αναεκμετάλλευση είναι το ποσό που φημολογείται ότι θα εγκριθεί, ανάλογα με τον αριθμό θέσεων στην κάθε γεωργική εκμετάλλευση. Και το το, θέμα, το διαβόητο θέμα των αντισταθμιστικών πληρωμών για το πρώτο, αναπρώτο εκτάριο, που θα είναι υποχρεωτικέ. Δεύτερος κανονισμός, πολύ σημαντικό κανονισμός, που είναι ο οριζόντιος κανονισμός. Και τέλος, η παρουσίαση που θα κάνει ο επίτροπο Χόγκαν τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, για αυτό το τελευταίο σημείο. Κάτι που έχει γίνει και είναι πολύ σημαντικό, είναι ο κανονισμός Omnibus που με μεγάλη δυσκολία εγκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις οργανώσεις παραγωγών και την εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού. Και μια πρόσφατη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές στην ε, αλυσίδα τροφίμων. Και μέχρι το τέλειο του έτου, το έτους περιμένουμε τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαφάνεια στην τροφική αλυσίδα, ε, συμπεριλαμβανομένης και της διαφάνειας των τιμών αυτά και τώρα θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Ντόρφμαν που είναι ο εισηγητής της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, επί της ανακοίνωσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας. Κύριε Ντόρφμαν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι των Αθηνικών Κοινοβουλίων. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Όπως ε, ήδη υπόθηκε, έχω αναλάβει ως εισηγητής να εκπονήσω έκθεση εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ε, ανακοίνωση, έκθεση πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας ε, της Επιτροπής. Να σας εξηγήσω λοιπόν με λίγα λόγια ποια είναι τα κύρια σημεία της έκθεσής μου και που θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση για τις πολιτικές αποφάσεις εδώ στο Κοινοβούλιο. Σημείο αφετηρίας, το επεσήμανε και ο Επίτροπος Χόγκαν, είναι το οικονομικό. Εάν δεν έχουμε τον απαραίτητο προϋπολογισμό στη διάθεσή μας, για μια πολύ σημαντική πολιτική που καλύπτει μεγάλο κομμάτι του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, λογικό είναι να μην είναι εφικτή η υλοποίηση αυτής της πολιτικής. Και εδώ ακριβώς ε, έγινε και η επισήμανση ότι με τον προϋπολογισμό, τον νέο, προπολογισμό προϋπολογισμό έχουμε εκρεμεί δύο ζητήματα. Το ένα είναι το Brexit και το άλλο είναι οι νέε αρμοδιότητες. Και εδώ λοιπόν ε, με τους ε, συνεισηγητές στα θέματα αυτά έχουμε συζητήσει την δυνατότητα να διατηρήσουμε στα επίπεδα που είχαμε μέχρι τώρα την χρηματοδότηση για τον προϋπολογισμό της Γεωργίας, γιατί θεωρούμε ότι δεν πρέπει η Γεωργία να πληρώσει το κόστος του Brexit. Περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα και από τον Επίτροπο Έτιγκερ τις σχετικές ε, τοποθετήσεις. Πάντως, το κενό που προξενείται από το Brexit είναι αρκετά σημαντικό κομμάτι και δεν θα πρέπει να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό. Απευθύνω έκκληση σας, Επίτροπε Χόγκεν, εδώ να, αλλά και σε εσά αγαπητοί συναδελφοί, να ασκήσετε τι απαιτούμενε ε, πιέσει προ τα κράτη-μέλη, ώστε να μην καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου η Γεωργία θα υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα ε, στον προπολογισμό. Ένα άλλο θέμα είναι ότι το Brexit συνιστά και κίνδυνο για τη Γεωργία. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με μια προσπάθεια για την ολοκλήρωση μιας εσωτερικής αγοράς. Η γεωργία κινδυνεύει να πληγεί λοιπόν ως τομέας από την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την δυνατότητα εξαγωγών γεωργικών προϊόντων η κυκλοφορία καλύτερα γεωργικών προϊόντων από τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Ηνωμένο Βασίλειο, βόηο, κρέας, γάλα, ε, οπορολαχανικά. Είναι τεράστιες οι ποσότητες και μπορεί η Έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση να οδηγεί σε τεράστια προβλήματα. Έτσι λοιπόν πρέπει να κοιτάξουμε και να μην είναι ο προϋπολογισμός πολύ πιο ε, μικρός για τη γεωργία, αλλά και ταυτόχρονα να μην υποστεί το ε, αντίκτυπο του Brexit η αγορά των γεωργικών προϊόντων. Σε τρία κομμάτια λοιπόν είναι διαρθρωμένη η έκθεσή μου, τα περιέγραψε και ο κύριος ε, Σάιμον, το πώς δηλαδή αναμένεται να εξελιχθεί η νομοθετική δραστηριότητα, αφενός με από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις προτάσεις, το New Delivery Model όπως ονοφέρεται, το ε, κομμάτι που αφορά τον πρώτο και δεύτερο πυλώνα που είναι και το σημαντικό βεβαίως ο πυρήνας της Ένωσης, της ε, πολιτικής για τη γεωργική πολιτική και βέβαια το τρίτο κομμάτι που αφορά τα υπόλοιπα περί την ε, κοινή γεωργική πολιτική ζητήματα. Νέες σχέσεις λοιπόν μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών. Έτσι θα μπορούσαμε να περιγράψουμε τη νέα κατάσταση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών και περιφερειών αυτών. Το είπε και ο Επίτροπος Χόγκαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προτείνει ε, μια σειρά από μια πολιτική δηλαδή η οποία θα στηρίζεται σε δείκτες με τακτική επαλήθευση του σεβασμού τους, πάνω στους οποίους δείκτες θα στηρίζεται η κοινή γεωρική πολιτική. Εγώ δεν τάσομαι επί της αρχής κατά μια τέτοιας προσέγγισης, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε πώς αυτή η κοινή γεωρική πολιτική που ήδη είναι αρκετά περίπλοκη δεν θα καταστεί ακόμη πιο ε, περιπλοκή με ένα τέτοιο σύστημα και πώς βεβαίως θα εξασφαλιστεί ένα πεδίο ε, δραστηριότητας, ένα ε, κομμάτι διακριτικής ευχέρειας στη διάθεση των κρατών μελών. Ωστόσο υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις που δεν μπορούμε να παραμελήσουμε. Ασφαλώς η σημαντικότερη προϋπόθεση ή όρος θα ήταν η πολιτική να παραμείνει κοινή γεωργική πολιτική. Γνήσια κοινή γεωργική πολιτική, γιατί μόνο τότε μπορεί να έχει νόημα. Μέσα σε μια κοινή αγορά και μέσα από μια κοινή ε, αγορά μπορούμε να έχουμε την υλοποίηση μιας κοινή γεωργικής πολιτικής. Και γι' αυτό όπου είναι να γίνει παρέμβαση στην αγορά, ε, δηλαδή οπουδήποτε ε, προσεγγίζει και αγγίζει την κοινή αγορά ή κοινή γεωρική πολιτική, πρέπει να έχουμε αυτή την προσέγγιση πάντα. Μελλοντικά μοντέλα της κοινή γεωρικής πολιτικής θα πρέπει να οδηγούν σε όσο το δυνατόν λιγότερες στρεβλώσεις της αγοράς. Ταυτόχρονα θα μπορούσα να δεχθώ και μια ιδέα, μια γενική ιδέα, ε, μιας πολιτικής που θα αναλάμβαναν να οργανώσουν προς τώρα τα εθνικά, ε, τα κρατη δηλαδή, σε εθνικό επίπεδο, με τα εθνικά στρατηγικά σχέδια και βέβαια μαζί με τις περιφέρειές τους, καθώς έχουμε και πολλά που ε, έχουν ε, μια κρατική οργάνωση με σαφείς αρμοδιότητες για τις περιφερειακές αρχές και άρα εδώ περνάμε στο δεύτερο πυλώνα, τα σχέδια ανάπτυξης της υπαίθρου και εδώ δεν είναι σαφέ για μένα ακόμα αυτέ οι περιφερειακέ αρμοδιότητε πώ μπορούν να συγκεραστούν με την αρμοδιότητα του κεντρικού κράτου. Γιατί θα υπάρχουν αποκλειστικέ αρμοδιότητε των περιφερειών, αλλά ταυτόχρονα αυτές θα πρέπει να υλοποιούν τις, τα εθνικά στρατηγικά σχέδια τα οποία θα έχουν χαράξει οι κεντρικές Είπε ο επίτροπο Χόγκαν ότι θα υπάρχει και ένα στάδιο έγκριση, μάλλον μια σταδιακή έγκριση του σχεδίου, του στρατηγικού σχεδίου και ίσως εκεί θα μπορούσαν να επιληθούν ζητήματα σχετικά με τις αρμοδιότητες των περιφερειών. Γιατί οπωσδήποτε δεν είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει στόχο να περικόψει, να περιστείλει τις αρμοδιότητες των περιφερειών. Και πάντως θα μπορεί να το κάνει αυτό γιατί είναι ζητήματα σταγματικής τάξης για ορισμένα κράτη-μέλη αρμοδιότητες των περιφερειών. Αυτά λοιπόν για το πρώτο κομμάτι, πρώτο-δεύτερο πυλώνα. Ε, πάνω απ' όλα πρέπει να μας απασχολήσει το ποιος είναι ο στόχος της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ποιος είναι ο βασικός στόχος. Βασικός στόχος της κοινή γεωργικής πολιτικής, πιστεύω, είναι η διαφύλαξη αυτού του ευρωπαϊκού μοντέλου της γεωργίας. Η, αγροτική οικογένεια, η αγροτική οικογενειακή επιχείρηση που είναι ευρέως δεδομένη στην Ευρώπη, που δραστηριοποιείται ακόμα και σε λιγότερο ευνοϊκέ συνθήκες, που έχει ένα σύστημα παραγωγής, ε, μία μέθοδο παραγωγής σε μεγάλο βαθμό ε, αηφόρο. Και έτσι, εάν θέλουμε πράγματι να υποστηρίξουμε αυτό το στόχο, πρέπει να ξανασκεφτούμε τη διαμόρφωση του πρώτου πυλώνα. Και εδώ θα επισημάνω δύο-τρία σημεία. Πρώτο σημείο λοιπόν, πρώτο ερώτημα. Υπολογισμός των απαιτήσεων σε πληρωμές και δι το σύστημα των πληρωμών στον πρώτο πυλώνα. Εδώ θα πρέπει να σχεδιάσουμε μια πολιτική η οποία από το 2020 και μετά θα ισχύσει, θα λειτουργήσει, θα φτάσει μέχρι το 2027. Μια νέα πολιτική όπου ο υπολογισμός της πρημοδότησης θα είναι ε, στηριγμένος σε ιστορικά δεδομένα για την επιχείρηση αλλά δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν το 2027 να εξακολουθούμε να πληρώνουμε ενισχύσεις ε, που έχουν υπολογιστεί, που έχουν στηριχθεί σε μια ιστορική ε, αναφορά, σε μια ιστορική περίοδο αναφοράς, 27 χρόνια πριν. Άρα πρέπει να βρούμε ένα νέο σύστημα, νέα συστήματα. Και νομίζω ότι πολλά κράτη-μέλη, πάντως αρκετά, έχουν βρει επιτυχείς λύσεις στο θέμα αυτό. Δεν μπορούμε βεβαίως να μιλήσουμε για καταποκοπήν ε, ποσά αλλά ε, πρέπει να βρούμε ένα σύστημα πρακτικό, ένα σύστημα το οποίο θα δίνει την ενίσχυση, θα καταβάλει ποσά σε αυτόν που πράγματι έχει ανάγκη και απέτηση και όχι σε αυτόν που δεν έχει καμία σχέση με τη γεωργική δραστηριότητα. Στα κράτη στα οποία υπάρχει ακόμη το σύστημα των ιστορικών αναφορών υπάρχουν ε, πολλοί δικαιούχοι χάρη σε αυτές τις ιστορικές αναφορές που δεν δραστηριοποιούνται πλέον εντατικά στη γεωργία. Και άρα δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να είναι ο στόχος ή το νόημα μιας ε, τέτοιας ε, κοινή γεωργικής πολιτικής. Εδώ έρχεται και το ζήτημα της ε, υποστήριξης των νέων γεωργών. Υπάρχουν αρκετοί νέοι που θέλουν να ξεκινήσουν γεωργική δραστηριότητα, αλλά δεν έχουν ε, δυνατότητα να διεκδικήσουν ενισχύσεις. Και άρα έχουν μειονέκτημα ανταγωνιστικό. Ένα πιο ενιαίο λοιπόν σύστημα θα πρέπει να αναζητήσουμε. Ένα σύστημα το οποίο θα μπορούσε να οδηγηθεί σε, μια, σε ένα σύστημα απλού υπολογισμού με τις αντισταθμιστικές πληρωμές, το, η περιβαλλοντική ενίσχυση ή κάτι άλλο το οποίο δεν είναι πλέον οι ιστορικές ε, αναφορές. Η εξωτερική σύγκληση επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία στη συζήτηση αυτή. Πρέπει όσο το δυνατόν να είναι δίκαιη η κατανομή των κονδυλίων, χωρίς αυτό να σημαίνει η λέξη δίκαιη, η κατανομή δεν σημαίνει πρέπει να είναι ισόποσες οι ενισχύσεις σε όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν διαφορετικές οικονομικές συνθήκες σε διάφορα κράτη-μέλη διαφορετικές εισοδηματικές συνθήκε. Κόστο παραγωγή διαφορετικό στη γεωργία. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να εκφραστεί μέσα σε μια σταδιακή διαμόρφωση των, του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα στην κοινή γεωργική πολιτική. Στι συνδεδεμένε πληρωμε πληρωμές. Ξέρω ότι ορισμένα κράτη-μέλη έχουν ε, ζητήσει περισσότερες συνδεδεμένες πληρωμές. Εγώ νομίζω ότι μέχρι τώρα αυτές όπως έχουν αρκούν για να καλύψουν κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Σημαντικό είναι οι συνδεδεμένες πληρωμές να μην οδηγούν σε στρεβλώσεις της αγοράς. Και ένα ζήτημα που πρέπει να συστήσουμε ακόμη σήμερα είναι η σταδιακή μείωση του κάπινγκ, του ανώτατου επίπεδου. Εδώ νομίζω ότι πρέπει Έντοιμα ε, να πούμε ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν μικρότερο κόστος λειτουργίας από τις μικρότερες και άρα αυτή η σταδιακή, μείωση ε, μπορεί να εισαχθεί χωρίς να επιβαρύνει την γεωργική παραγωγή, γιατί είναι χαμηλότερο το κόστος της. Είναι κάτι το οποίο έχουμε συστήσει και θα, θα ξανασυστήσουμε τις επόμενες ημέρες εδώ στο Κοινοβούλιο. Ένα υποχρεωτικό κάπινγκ λοιπόν σε επίπεδο ευρωπαϊκό, ταυτόχρονα όμω λαμβανομένης υπόψη και τη κατάσταση στην απασχόληση στο καθε κράτο, κράτος, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν κράτη-μέλη, ιδιαίτερα αυτά τα οποία έχουν ε, βγει από το παλαιό κομμουνιστικό καθιστώς, έχουν κάποιε δομέ μεγάλε σε μέγεθο, αλλά που απαρτίζονται από πολλέ μικρότερε οικογενειακές εκμεταλλευσει που συνεργάζονται μεταξύ του. Αυτές τις δομές οπωσδήποτε δεν θέλουμε να τις περιορίσουμε ή να τις πλήξουμε. Άρα λοιπόν θέλουμε ένα κάπινγκ να λαμβάνει υπόψη και τον αριθμό των απασχολουμένων, ώστε να μην οδηγήσει σε ε, μετακύληση εισοδήματος από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, σε αναδιανομή δηλαδή, μεταξύ κρατών μελών. Πρέπει αυτό, αυτή η αναδιανομή να γίνεται μέσα στο ίδιο κράτο μέλο και από το ένα κράτο μέλο στο άλλο. Για την ε, δομή, την αρχιτεκτονική αυτού του συστήματο. Ε, νομίζω όντω ότι δεν έχει φέρει οικολογικοποίηση τα αποτελέσματα που περιμέναμε. Θα χρειαστεί μια νέα διαμόρφωση λοιπόν, ένα νέο σχεδιασμό τη οικολογικοποίηση. Αυτό σημαίνει σαφή αιρεσιμότητα για τον πρώτο πυλώνα, προστασία των πότσιμων υδάτων, ε, της ποιότητας ε, του ατμοσφαιρικού αέρα, προστασία από την κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά είναι καθήκοντα κοινά που πρέπει να καλυφθούν από τον πρώτο πυλώνα. Και οπωσδήποτε στον πρώτο, στα, στα κράτη-μέλη, στο σύνολο των κρατών μελών, πρέπει να υπάρξει ε, και η λειτουργία ε, με καλά αποτελέσματα και του δεύτερου πυλώνα. Μεγάλη πρόκληση επίσης για μένα είναι η εναλλαγή των γενναιών. Εδώ θα χρειαστεί μια στρατηγική των κρατών μελών η οποία θα ξεπερνάει και την κοινή γεωργική πολιτική, γιατί υπάρχουν πολλές αποφάσεις που μπορούν να ληφθούν σε επίπεδο κράτους μέλους σχετικές με την ενίσχυση της παρουσίας των νέων και τη δυνατότητα για ανάληψη γεωργικής δραστηριότητας από νέους πολίτες. Λιγότερα πράγματα λέω στην έκθεσή μου για το δεύτερο πυλώνα, όντω διότι θεωρώ ότι ο δεύτερο πυλώνας με την ανάπτυξη τη υπαίθρου έχει γενικά δώσει καλά αποτελέσματα σε μεγάλο βαθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο δεν θα πρέπει να ε, συνεχιστεί η γραφειοκρατική επιβάρυνση που παρουσιάζει αυτός ο δεύτερος πυλώνας. Θα πρέπει να ελαφρυνθεί λοιπόν ο γραφειοκρατικός φόρτος του δεύτερου πυλώνα. Και κάτι ακόμη για τις ε, οργανώσεις αγοράς, για τα οποροκυπευτικά και το κρασί. Βλέπουμε κάποια καλά αποτελέσματα. Ε, ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να επιδιώξουμε και μια αναθεώρηση του κατά πόσο τα συστήματα αυτά ισχύουν ή μπορούν να ισχύσουν με την ίδια χρησιμότητα και σε άλλους τομείς. Στην ε, παραγωγή γάλακτο σε ορεινέ περιοχέ, παραδείγματι, θα πρέπει να εξετάσουν οι υπηρεσίε Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν κάτι τέτοιο μπορεί να υλοποιηθεί, αν χρειάζεται μια διαφορετική ενίσχυση των ε, φορέων που δραστηριοποιούνται στην αγορά. Ακόμα δύο σημεία. Ε, εξασφάλιση από τον κίνδυνο, από τη διακινδύνευση. Εδώ δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε πολλά. Ε, αναφέρθηκε ήδη ο κανονισμό Omnibus. Έχει διαμορφωθεί αυτό ως ένα κεντρικό μέσο και εργαλείο για να προστατέψει τον γεωργό από τον κίνδυνο κατά, την, κατά τη γεωργική δραστηριότητα και εδώ δεν χρειάζεται, θεωρώ, νέα μέσα. Χρονοδιάγραμμα. Στόχο μου, στόχο δικό μου και των σκιωδών εισηγητών εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να, κατατεθεί, ψηφιστεί στι 17 Μαΐου η, η έκθεση αυτή στη Γεωργική Επιτροπή, έτσι ώστε στα τέλη Μαΐου να περάσει από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να είμαστε και εμεί έτοιμοι να προσφέρουμε τη δική μα συμβολή στην ε, νομοθετική αυτή διαδικασία. Σα ευχαριστώ πολύ. Euh, Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Πλάνκ, το Γενικό Γραμματέα στο Αυστριακό Υπουργείο Βιωσιμότητας και Τουρισμού. Μια και η Αυστρία θα αναλάβει την επόμενη Προέδρια του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Καθόλου εύκολο έργο. Κύριε Πλάνκ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Προεδρεύον, αγαπητοί συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού αλλά και των Εθνικών Κοινοβουλίων, κυρίες και κύριοι, Χαίρομαι ιδιαίτερως για την πρόσκληση αυτή και τη δυνατότητα να συμμετάσχω στη σημερινή συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ακρόαση για το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής και τη σημασία της ανάπτυξης υπαίθρου που μας απασχολεί και βεβαίω ήθελα να παρουσιάσω και τα θέματα πλευρά τη Αυστρία. Είναι μια ιστορία επιτυχία η κυνηγιορική πολιτική. Αυτό βλέπω και από την προοπτική τη Αυστρία. Και πιστεύω ότι θα παραμείνει και στο μέλλον κεντρικό τομέα δραστηριότητα τη ευρωπαϊκή πολιτική. Πρόκειται λοιπόν για κοινού κανόνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πρόκειται για μια πολιτική την οποία η Ευρώπη ως σύνολο διαμορφώνει. Τώρα βεβαίως περνάει σε μια άλλη θεώρηση η Ευρώπη μέσα από την πολυμορφία της και είναι μεγάλη η πολυμορφία της Ευρώπης ε, θα διαμορφώνει αυτή την ε, κοινή πολιτική. Η κοινή γεωργική πολιτική έχει πάντα αποδείξει ότι είναι σε θέση να φέρνει πάντα καλά αποτελέσματα για την ε, γεωργική οικογένεια, για την οικογένεια, την ε, οικογενειακή εκμετάλλευση, αλλά και για την Ευρώπη και τον Ευρωπαίο γενικότερα. Γι' αυτό και είμαι αισιόδοξο ότι και εδώ θα, ε, και στη νέα πολιτική θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις προτάσεις της ε, διαμόρφωσε από πέρσι τα πρώτα βήματα. Τα κράτη-μέλη υιοθέτησαν πιστεύω με πολύ θετική ανταπόκριση στα συμπεράσματά τους ε, τις προτάσεις αυτές ε, λέγοντας ότι παραμένει η κοινή ορική πολιτική σημαντική κοινή πολιτική. Αυτή άλλωστε είναι και η προσέγγιση της Αυστρίας η κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να παραμείνει και στο μέλλον κοινή πολιτική. Εν όλο βεβαίως ε, πρόκειται για μια κατάσταση όπου αντιμετωπίζουμε αρκετές ε, προκλήσεις. Έχουμε να κάνουμε με την ανάγκη για μια σύγχρονη παραγωγική κοινή γεωργική πολιτική, η ε, ποικιλομορφία του χώρου της υπαίθρου πρέπει να διαφυλαχθεί και να ενισχυθεί. Πρέπει να ενισχυθεί η ψηφιοποίηση, να εξασφαλιστεί η παραμονή στην ύπεθρο ε, δραστηριότητα των ε, οικογενειών των γεωργών και των εκμεταλλεύσεών τους. Ξέρετε ότι για την Αυστρία αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και βέβαια στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής είναι και η προσφορά της γεωργίας στην επιστηστική ασφάλεια και στην παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας, υψηλής στρατηγικής αξίας. Έχει και αυτό πολύ μεγάλη σημασία και πιστεύω ότι και στο μέλλον θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Η Προεδρία λοιπόν της Αυστρίας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε και στο μέλλον ε, η γεωργική πολιτική να ε, είναι σε θέση να υλοποιήσει τους στόχους της ε, για τους γεωργούς, άντρες και γυναίκες, χωρίς τίποτε θα μπορούσε να γίνει, για τους καταναλωτές και πολίτες ευρύτερα, αλλά και για όλη την κοινωνία. Η συζήτηση για τις νομοθετικές προτάσεις ε, θα ε, συνεχιστεί, θα συνεχίσουμε εμείς λαμβάνοντας τη σκητάλη από τους βούλγαρους συναδέλφους και θα συνεχίσουμε την συζήτηση στο Συμβούλιο. Το Σεπτέμβριο έχουμε άτυπο Συμβούλιο, 23 και 24 ε, Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα, που θα αξιοποιήσουμε για μια εντατική ανταλλαγή απόψεων και σας διαβεβαιώ ήδη από τώρα πως η Προεδρία της Αυστρίας θα ε, επιδιώξει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και πρόοδο σε συνεργασία με όλους τους εταίρους για ε, τις διαπραγματεύσεις αυτές της κοινής γεωργικής πολιτικής. Σημείο ε, είναι αυτή η θετική κατάσταση που σας περιέγραψα με την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που ε, στρέφεται μεν προς το μέλλον χωρίς όμως να κάνει να διακόψει το μοντέλο το οποίο έχουμε. Η σημασία των άμεσων ενισχύσεων αναγνωρίζεται, η προσέγγιση με τους δύο πυλώνες συνεχίζεται. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει και να διατηρηθούν οι προϋποθέσεις εκείνες οι οποίες θα διευκολύνουν την ε, δραστηριοποίηση των ε, γεωργικών ε, οικογενειών, να γίνει πιο απλό δηλαδή το σύστημα, να έχει βεβαίως την προσέγγιση στο περιβάλλον, να έχει την, το στόχο της καταπολέμησης του κλίμα, της κλιματικής αλλαγής, μεγάλες προκλήσεις που πρέπει να υλοποιηθούν χωρίς να επιβαρυνθεί το σύστημα με περισσότερη γραφειοκρατία. Αυτό έχει κρίσιμη σημασία για την αποδοχή του νέου συστήματος ε, από τους πολίτες. Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι η γεωργία παράγει δημόσιο αγαθό. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να γίνει ένα βαρύ και δυσκίνητο ε, σύστημα. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα για την Αυστρία. Το σύστημα που εμεί θα προτιμούσαμε είναι ένα σύστημα με περισσότερη επικουρικότητα για τα κράτη-μέλη. Κατά βάση λοιπόν αυτό το κρίνουμε θετικά, γιατί έτσι μπορεί να γίνει σεβαστή η πολυμορφία, οι διαφορέ μεταξύ των κρατών μελών, βεβαίω, ναι. Είναι θετικό αυτό το σύστημα. Ταυτόχρονα όμω ε, παραμένει ανοιχτό το πώ θα διαμορφωθεί αυτό το σύστημα, γιατί δεν πρέπει να οδηγεί εν τέλει σε μία ε, διάρρηξη του κοινού ιστού, της κοινή γεωργικής πολιτικής δηλαδή. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε την έννοια της σκηνής στη γεωργική πολιτική. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ σημαντικό σημείο για τις ε, γεωργικές οικογένειες. Έχουμε την ιστορική θεώρηση όπως υπόθηκε ήδη. Μεγάλη σημασία έχει για την Αυστρία γιατί έχει στενή διασύνδεση με τις ε, δραστηριότητες, όχι μόνο τις ιωρικές, αλλά και τις τουριστικές δραστηριότητες σε όλη την ε, περιοχή της Αυστρίας και αυτές θα πρέπει να διαφυλαχθούν και στο μέλλον. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα κεντρική σημασία ε, καθήκον και βέβαια θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, άλλωστε χρόνια τώρα το επισημαίνουμε, να ενισχυθεί όχι μόνο ο πρώτο πυλώνας, αλλά και ο δεύτερος ε, πυλώνας να διατηρήσει τη σημασία του και για την προαγωγή των εθνικών συμφερόντων, την έννοια δηλαδή της προαγωγής του περιβάλλοντος, της υποστήριξης των μειονεκτουσών περιοχών και ούτω καθεξής. Η κοινή γεωρική πολιτική πρέπει να παραμείνει ένας ανοιχτός δρόμος για την περαιτέρω οικολογικοποίηση στο χώρο της γεωργίας προ όφελο τη κοινωνία ευρύτερα, προ όφελο του καταναλωτή που άλλωστε και το απαιτεί. Το Και νομίζω ότι μπορούν οι γεωργικέ εκμεταλλεύσει αυτό να το υλοποιήσουν. Σημαντικό για μα είναι στο δεύτερο πυλώνα να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα περιβαλλοντικά γεωργικά προγράμματα και αυτά να προβάλλονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό γιατί όπως είπα πρόκειται για ένα σημαντικό κομμάτι του, της υπαίθρου ο δεύτερος πυλώνας με την περιβαλλοντική του διάσταση στηρίζει ταυτόχρονα και την τουριστική δραστηριότητα και με τη σειρά της αυτή τουριστική δραστηριότητα στηρίζει την γεωργική δραστηριότητα που έτσι παραμένει ελκυστική και για τη νεότερη γενιά. Για να το εξασφαλίσουμε λοιπόν αυτό, και νομίζω ήδη αναφέρθηκε, πρέπει να δώσουμε έμφαση στο εξής, ότι χρειάζεται μια ανοιχτή, γερή και ε, προβλέψιμη διαδικασία στη γεωργική πολιτική. Δηλαδή πρέπει κανείς ξεκινώντας μια δραστηριότητα να γνωρίζει τι μπορεί να περιμένει. Ασφαλώς κάποιος ο οποίος ε, περιμένει ότι η προσφορά στην κοινωνία της γεωργίας μπορεί να αλληλοποιηθεί με λιγότερα κονδύλια, απατάται αυτό το έχουμε αντιληφθεί, χρειάζεται να εξασφαλιστεί το υφιστάμενο επίπεδο χρηματοδότησης. Πρέπει η γεωργία μας να διατηρήσει την πολυμορφία της, ναι, πρέπει να είναι και βιώσιμη και άρα πρέπει να βρούμε τους τρόπους να την υποστηρίξουμε. Έτσι λοιπόν, ο γεωργικός προϋπολογισμός πρέπει να διαφυλαχθεί Χωρίς όμως ταυτόχρονα και να λησμονούμε ότι τα σημεία τα οποία έχουν εντωμεταξύ ε, εισαχθεί στη συζήτηση διαφύλαξη και της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων, διαφύλαξη της ε, γεωργικής εκμετάλλευσης, θα πρέπει να ε, δίνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Και όλα αυτά με την προϋπόθεση της ισότιμης συμμετοχής σε μια ελεύθερη και ανοιχτή αγορά. Με μια γεωργία η οποία θα είναι διαρθρωμένη κατά τρόπο ισοδίκαιο και έναντι και του υπόλοιπου κόσμου. Η ύπεθρος λοιπόν, η γεωργία θα πρέπει να δώσουν το χώρο στην ε, γεωργική εκμετάλλευση με σταθερό ορίζοντα, με πολυμορφία χωρίς υπερβολική επιβάρυνση και πίεση για την ύπεθρο, χωρίς επιβάρυνση υπερβολική των ε, ανθρώπων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστούμε κύριε Πλάνκ. Θα περάσουμε στη συζήτηση. Θα παρακαλούσα τον πρόεδρο της Επιτροπής Άγκρη, τον κύριο Σεκιάσκη, να συντονίσει τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ κύριε Σιμό για την εισαγωγή που μας κάνατε σε αυτό το πρώτο πάνελ. Όπως ε, είχα αναγγείλει, θα ισχύσει η εξής διαδικασία. Οι ομιλίες θα είναι δίλεπτες φαίνεται λίγο, αλλά και παίρνει διπλάσιο από ό,τι συνήθω δικαιούνται οι ευρωβουλευτέ στη συζητήση του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ακούμε δύο βουλευτέ από Εθνικά Κοινοβούλια και κατόπιν ένα ευρωβουλευτή από την Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έτσι. Θα συνεχίσουμε και εγώ δέκα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του χρόνου θα σηκώνω το σφυράκι μου για να ξέρετε ότι πλησιάζει η ώρα. Ο κύριος Γέρικ από τη Γερμανία έχει το λόγο. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πάντα ε, δείχνω σεβασμό στο σφύρι του Πρόεδρου. Θα σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για την ε, οργάνωση για τις ε, ομιλίες, για τη δυνατότητα για συζήτηση αυτής της κοινή γεωργικής πολιτικής που όλοι βεβαίω θέλουμε να δούμε να συνεχίζεται. Εμείς στη Γερμανία, όπως και εσείς άλλωστε, και άλλωστε το έχουμε περιλάβει και στον κυβερνητικό, στη Συμφωνία Κυβερνητικού Συνασπισμού, θέλουμε να δώσουμε στο δυνατόν περισσότερα χρήματα στη Γεωργία. Η Γερμανία μάλιστα έχει δηλώσει διάθεση να προσθέσει και φρέσκο χρήμα στην ε, γεωργική πολιτική Αυτά βεβαίως θα οριστούν και με την κατανομή και τις ανάγκες όπως θα προκύψουν στην περαιτέρω συζήτηση. Η κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να έχει κονδύλια στη διάθεσή της, τα οποία θα στηρίζουν την οικογένεια, τη γεωργική, το είπανε πολλοί ομιλητές ε, ήδη τώρα. Είναι τεράστιες διαρθρωτικές εξελίξεις ε, στην Ήπεθρο σε όλη την Ευρώπη και πρέπει να αγωνιστούμε για ισότιμη στήριξη. Πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική αλλά και πιο ε, απλή η κοινή γεωργική πολιτική. Είναι θέση μου λοιπόν ε, αυτή, κυρίως αυτό θέλω να μεταδώσω, ότι δεν χρειάζεται μια υπερβολική γραφειοκρατία. Πρέπει να δώσουμε έμφαση στην απογραφειοκρατικοποίηση. Χρειάζεται προοπτική επίση για το μέλλον η δυνατότητα να ε, μπουν στο, στην γεωργική δραστηριότητα ε, και οι νέοι. Και να υπάρχει δυνατότητα να στηριχθούν από την κοινή γεωργική πολιτική. Θεωρώ ότι οι θεμελιώδεις ε, δομές με τις άμεσες ενισχύσεις θα πρέπει να παραμείνουν στα χέρια του εις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια στις συνδεδεμένες ε, ενισχύσεις πρέπει να γίνει μεγάλη συζήτηση γιατί εμείς από τη Γερμανία αντιμετωπίζουμε σοβαρές στρεβλώσεις ανταγωνισμού. Ευχαριστώ. μικρόφωνο ο Πρόεδρος. Ο κύριος Τέγκιάραν από την Ιρλανδία. Μικρόφωνο ο μιλητής δεν έχει ανοίξει. Sorry, sorry, sorry, Chairman. Thank you. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Τράτω με τις ευκαιρίες να απευθυνθώ σε αυτή τη διάσκεψη. Μιλούσε πριν ο Επίτροπος Χόγκεν και σωστά εστιάστηκε στον προπολογισμό και τις επιπτώσεις που θα έχει ο γενικός προπολογισμό σε σχέση με την ΚΑΠ. Και ξεκάθαρα είπε ότι χρειάζεται οι εθνικές κυβερνήσεις να λάβουν τις ευθύνες τους και να βρουν τα απαιτούμενα κονδύλια. Ως μέλος του Κοινοβουλίου της Ιρλανδίας, αυτό που εγώ θα ρωτώ είναι το εξή που ρωτώ εάν τα κράτη-μέλη συμφωνήσουν, οι κυβερνήσει συμφωνήσουν να καλύψουν το κενό του Brexit και χρηματοδοτήσουν αυτά τα 12 δισεκατομμύρια που λείπουν, λοιπόν μπορούμε να έχουμε διαβεβαιώσει ότι αυτά τα χρήματα θα πάνε στην κοινή αγροτική πολιτική, ότι θα προστατευτεί η ΚΑΠ, ότι δεν θα πάνε σε άλλε τομεί προτεραιότητε τη Επιτροπή. Έχουμε επίση και άλλε προκλήσει να αντιμετωπίσουμε, όπω για παράδειγμα τη συμφωνία με τι χώρε Μερκοσούρ, πέρα από το Brexit διαπιστώνουμε ότι σε αυτή τη συμφωνία κάναμε παραχωρήσει, οι οποίε θα βλάψουν την αγορά του βόλιου κρέατος, ε, τους παραγωγού. Και αυτό θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα δεδομένου του Brexit. Θα ενταθεί το πρόβλημα. Όμως όταν έχουμε μια, ένα τέτοιο περιβάλλον και με αυτά τα επιχειρήματα, ε, φαντάζομαι δεν αμφιβάλλει κανεί ότι πρέπει να προστατεύσουμε τα κονδύλια που θα είναι διαθέσιμα για την ΚΑΠ. Και το ερώτημά μου λοιπόν είναι, εάν βρουν αυτά τα επιπλέον χρήματα, αυτού του επιπλέον πόρου που χρειάζονται οι κυβερνήσει, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει την ΚΑΠ που της αξίζει, έτσι ώστε να έχουμε παραγωγή τροφίμων ε, υψηλότερου επίπεδου, όπως επιθυμούν οι καταναλωτές μας. Και για να προασπίσουμε τις ε, βελτιώσεις και τα επιτεύγματα της ΚΑΠ ανά τις τελευταίες δεκαετίες, το ερώτημα λοιπόν είναι, θα καταλήξουμε σε μια ΚΑΠ η οποία να επιτύχει τους στόχους που θέτουμε για την περιφέρεια, για την, ε, τους αγρότες στην Ευρώπη. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η προστασία ring fencing των κονδυλίων για την ΚΑΠ, εφόσον συμφωνήσουν οι κυβερνήσει στο συνολικό προπολογισμό, θα είναι απαραίτητη. Ευχαριστώ. Έχουμε στην αίθουσα και καλεσμένο τη κυρία Πετήρ από την Κροατία. Από την Ολλανδία, καλεσμένο τη κυρία Ράιερ και, από και καλεσμένο του κυρίου Τσούλο από την Ιταλία. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους επισκέπτες μας και να δώσω το λόγο στον κύριο Άλμπερ Τες. Ε, για τους ευρωβουλευτές θα είμαι ακόμη πιο αυστηρό στην τηρήση του χρόνου. Δύο λεπτά είπα και ούτε δευτερόλεπτα παραπάνω. Πρόεδρε, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχει αποχωρήσει ο Επίτροπος ε, Χόγκαν δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς έχει σχεδιάσει την πρόταση και πρέπει να πω ότι δεν με ενθουσιάζει αυτό το λίγο που γνωρίζω για την πρόταση. Δεν δίνει δηλαδή την εντύπωση ότι θα είναι λιγότερο γραφειοκρατικό το σύστημα. Απλώς η γραφειοκρατία από το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα περάσει στα κράτη-μέλη. Κάτι το οποίο δεν μπορούμε να, σκεφτούμε, να δεχθούμε. Επίσης ε, υπάρχει κίνδυνος να εμφανιστούν και διαφορετικές προσεγγίσεις στα κράτη-μέλη με αποτέλεσμα περισσότερες τρευλώσει του ανταγωνισμού. 50 χρόνια τώρα έχουμε μια κοινή γεωργική πολιτική. Τότε που ξεκίνησα και εγώ τη γεωργική μου δραστηριότητα, δηλαδή ξεκινούσε και η γεωργική πολιτική. Με αυτήν λοιπόν συνέχισα τη δραστηριότητά μου και μπορώ να πω ότι γνωρίζω τις διάφορες ε, προτάσεις και το ιστορικό τους ε, με ε, τις επιλογές που έγιναν τελευταία μεταρρύθμιση. Η γεωργική πολιτική έγινε όλη αυτή την πεντηκονταετία το εργαλείο και της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Δεν πρέπει λοιπόν να διαλυθεί. Νομίζω ότι πρέπει να καταθέσουν πλέον ε, τις προτάσεις τους για το περιβάλλον, τα κράτη-μέλη, να τα ε, εξετάσουμε, να τις περιλάβουμε σε ένα κατάλογο και από τον κατάλογο αυτό μέτρων για το περιβάλλον να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μια επιλογή τα κρατημέλη ανάλογα με τις διαφορετικές συνθήκες που ισχύουν στο καθένα. Χρειάζονται, χρειάζεται να διατηρηθούν οι δύο πυλώνες, έστω και με βελτιώσεις που είναι οπωσδήποτε απαραίτητες. Οι προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής βλέπω να μην αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της κατάστασης και βλέπω επίσης να προχωρούν με πολύ ράθιμους ε, ε, ρυθμούς. Δεν φαίνεται να είναι σε θέση δηλαδή να εγκριθούν πριν να λήξει η θητεία. Μέχρι το καλοκαίρι δεν αναμένονται συγκεκριμένε προτάσεις και μετά μας μένουν πολύ, λίγες, ε, πολύ λίγοι μήνες από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Απρίλιο για να εγκριθούν οι προτάσεις. Ελπίζω ο Επίτροπος να καταθέσει το χέτερο δυνατό καλές προτάσεις και να ε, είναι δυνατό να τις εγκρίνουμε εγκαίρως. Για τον προϋπολογισμό, 40% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού περνάει στη Γεωργία. 1% των δαπανών ε, του συνολικού ΑΕΠ για τους γεωργούς που ε, φροντίζουν με, καλή, με καλά τρόφιμα την επιστηστική ασφάλεια των 500 εκατομμυρίων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι αυτό το 1% είναι πολύ λίγο. Εγώ σας είπα ότι οι ευρωβουλευτές έχουν συνηθίσει σε σύντομες παρεμβάσεις. Ο κύριος Καυκαλιάς από την Κύπρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ και εσάς και την Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διοργάνωση της παρούσας συνάντησης. Ομολογουμένως, η μείωση της γραφειοκρατίας, η απλοποίηση των διαδικασιών, ώστε να γίνεται και πιο εύκολα κατανοητή από τους αγρότες, η στόχευση και ο εξυγχρονισμός της ε, ΚΑΠ και η αύξηση της συνεχτικότητάς της με άλλες πολιτικές της Ένωσης είναι ένα βασικό ζητούμενο. Παράλληλα, οι προσπάθειε των κρατών μελών για τήρηση των περιβαλλοντικών προτύπων στου τομεί τη γεωργία και των τροφίμων στη βάση των προνοιών τη Συμφωνία των Παρισίων και των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών πρέπει να συνεχιστούν απρόσκοπτα μέσω ενίσχυση τη παροχή κινήτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδιαίτερη έφαση πρέπει επίση να δοθεί στην αντιμετώπιση των αθέμητων εμπορικών πρακτικών με στόχο την επίτευξη μια πιο ισορροπημένη αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και την ενίσχυση τη θέση των γεωργών, όχι μόνο εντό τη αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, αλλά και ευρύτερα στη γεφύρωση του χάσματο ανάμεσα στο εισόδημα των αγροτών και των άλλων επαγγελματιών, όπω πολύ σωστά έχει σημειώσει και ο Ευρωπαίο Επίτροπο, ο κ. Χόκαν, στην αναφορά του. Περαιτέρω, θα ήθελα να υπογραμμίσω την ανάγκη παροχή στοχευμένων μέτρων και κινήτρων για αποτελεσματική αντιμετώπιση τη πρόκληση τη γύραση του αγροτικού πληθυσμού, ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα τη γεωργία. Υπογραμμίζω επίση την ανάγκη διατήρηση του επίπεδου χρηματοδότηση τη ΚΑΠ στο πλαίσιο του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου μετά την έξοδο τη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια αλλά και από τη διαφαινόμενη ιεράρχηση άλλων τομέων όπως η άμυνα και η ασφάλεια, πιο ψηλά στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την άλλη. Τέλος, θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη μία στην περίπτωση της Κύπρου, η οποία αποτελεί απομονωμένη αγορά μικρού μεγέθους χωρίς χερσαία διασυνδεσιμότητα. Η Κυπριακή Γεωργία αντιμετωπίζει σημαντικέ προκλήσει λόγω του αυξημένου κόστου άσκηση γεωργική δραστηριότητα. Η αγορά είναι απομακρυσμένη από τα διεθνή κέντρα και οι γεωργοί μα καλλιεργούν μικρά τεμάχια γη, γεγονό που μειώνει τη διαπραγματευτική του δύναμη. Παράλληλα, η Κύπρο βιώνει τι έντονε επιπτώσει των κλιματικών αλλαγών και του αρνητικού αντίκτυπου του φαινομένου τη αστυνοφιλία στι αγροτικέ περιοχέ. Οι ιδιαιτερότητε αυτέ συνεπάγονται αύξηση του κόστου παραγωγή και διάθεση των αγροτικών προϊόντων. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. για το μέλλον της ΚΑΠ και τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ ζητούμε από τους γεωργούς και κτηνοτρόφους να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων να συμβάλλουν δηλαδή στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Αλλά οι αγρότες μας ήδη αντιμετωπίζουν πολλές δημοσιονομικές και χρηματοοικονομικές δυσκολίες. Θα έχουν μεγάλες ζημιές λόγω του Brexit. Και δεν θα πρέπει να ξεχνούμε τους παραγωγούς που είναι βασική κρίκη της τροφικής αλυσίδας. Εμείς στην Ισπανία θεωρούμε τους γεωργούς και κτηνοτρόφους πρωταγωνιστές του μέλλοντος της κοινή γεωργικής πολιτικής. Γι' αυτό και έχουμε τις εξής σκέψεις. Τι θα γινόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση αν θα έπρεπε να εξαρτά την ποσότητα και την ποιότητα των τροφίμων της σε τρίτες χώρες. Πολλοί μας ανησυχεί και προβληματίζει η απόπειρα επανεθνικοποίησης της κοινή γεωργικής πολιτικής. Μας α, θορυβούν αυτές οι φήμες για συγχρηματοδότηση των άμεσων ενισχύσεων, μα οι άμεσες ενισχύσεις είναι το δίκτυο ασφαλείας για τους γεωργούς και κτηνοτρόφους μας. Και μην ξεχνάτε ότι οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι μας είναι οι θεματοφύλακες της συνοχής και οι πρωταγωνιστές της κοινή γεωργικής πολιτικής. Κάτι άλλο που μας ανησυχεί τα μάλα είναι το γεγονός ότι η διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών μπορεί να αποβεί βάρος της κοινή γεωρικής πολιτικής, που είναι το βασικό στοιχείο της συνοχής της μελλοντική μεταρρύθμισης της κοινή γεωρικής πολιτικής. Γι' αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, γίνεται πολλής λόγος για τις μελλοντικέ προκλήσεις και τις νέες προκλήσεις, αλλά μην ξεχνάτε ότι... Ε, θα πρέπει να διατηρηθεί το 30% των βασικών ενισχύσεων ε, ε, που είναι το 30% των συνολικών γεωργικών ε, δαπανών. Και θα πρέπει οι άμεσες ενισχύσεις να εξακολουθούν να χρηματοδοτούνται πλήρως από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σαντρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ λυπάμαι που χρειάστηκε να φύγει ο Επίτροπος, γιατί το πιο φλεγόν ζήτημα είναι το δημοσιονομικό. Την περασμένη ε, Τρίτη μας, μας μίλησε για μείωση 10 με 15% του προϋπολογισμού και την Πέμπτη το πρωί ο Επίτροπος Έτιγκερ ε, ανέφερε τη μείωση κατά 6%. Βέβαια θα δούμε την τελική πρόταση σε λίγες μέρες. Στις 2 Μαΐου θα υποβληθεί η πρόταση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πάντως το ζήτημα είναι σοβαρό και φλέγων. Άλλο θέμα, το χρονοδιάγραμμα. Και αυτό είναι προβληματικό. Και η διάρκεια του χρονοδιαγράμματος θα εξαρτηθεί από την ποιότητα της νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό που φοβόμαστε από τις φήμες που κυκλοφορούν ή κάτι που έχει διαρρεύσει είναι ότι ε, ίσως ε, ε, να μην είναι και πολύ λεπτομερή η νομοθετική πρόταση λόγω επικουρικότητας. Βέβαια, ε, το Συμβούλιο είπε ε, ότι έχει σαφή αντίληψη για το μέλλον της ΚΑΠ. Αυτό μας είπε ο Βούλγαρος υπουργό. Το, το, το Συμβούλιο το μόνο που έχει ε, σαφές όραμα για το μέλλον της ΚΑΠ, γιατί οι υπόλοιποι δεν έχουμε. Θα είναι σημαντική λοιπόν η ποιότητα της νομοθετικής πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα κρίνει και τη συνέχεια. Ε, σπέβδε βραδέως, ε, δεν θα πρέπει να βιαστούμε πολύ και θα πρέπει να έχουμε και εκτενείς διαβουλεύσεις. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της μεταρρυθμίσης, εκεί έχουμε σημαντικά στοιχεία. Σε ό,τι αφορά τα μέσα διαχείρισης της αγοράς, ο κύριος Δόρφμαν που είναι ο συντάκτης της έκθεσης πρωτοβουλίας, είπε ότι το όμνιμπου συνιστά πρόοδο. Ναι, σίγουρα είναι απαραίτητο, αλλά όχι ικανό... Ε, είναι απαραίτητο, αλλά όχι ικανή η πρόοδος που έχει, έχουμε επιτελέσει με το omnibus. Δεν αρκεί αυτή ε, η πρόοδος. Επίσης, το πρώτο επίπεδο είναι το, ο κοινό πυλώνα και θα πρέπει να ενισχύεται με την αρισιμότητα να μην ψησφορά τη βιολογική γεωργία. Αλλά θα πρέπει να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι. Να πάμε στην ε, επιλογή 1 που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή ένα μείγμα των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων και το οικολογικό σύστημα, το eco και πιστεύω ότι αυτά θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά για όλου του γεωργού τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην είναι προαιρετικά. Αυτό θα είναι σημαντικό στοιχείο τη μελλοντική μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική πολιτική. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ακούμε πολλά διαφορετικά ποσοστά, πολλά διαφορετικά νούμερα. Αλλά θα πρέπει να δούμε αν θα είναι πάγια πόσα αναφορούν συγκεκριμένο έτος, σε τι αναφέρονται γιατί θα πρέπει να δούμε και τις τάξεις μεγέθους και σε τι αναφέρονται. Ο κύριος Αρνανόφσκι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας επιτρέπετε να παρουσιάσουμε τη θέση και της Πολωνικής Βουλής. Πολλά δε μάλλον που με ειδικό ψήφισμα η Πολωνική Βουλή παρά τη διαφορά απόψεων, στήριξε την πολωνική κυβέρνηση στις προσπάθειες να διαμορφώσει τη μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική. Θα σταθώ σε μερικά σημεία που είναι σημαντικά για την Πολωνία. Πρώτα απ' όλα ήρθε η ώρα να ε, ολοκληρώσουμε την εξίσωση των, και τη σύγκληση των ε, ενισχύσεων του πρώτου πυλώνα. Ε, Στη, στο νέο πολιτή δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να έχουμε εξίσωση αυτών των ενισχύσεων. Γιατί είναι άδικα τα ιστορικά δικαιώματα και θα πρέπει να σταματήσουν να λαμβάνονται υπόψη. Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των θέσεων των μικρομεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Το είπα και πολύ προλαλήσαντες. Ε, ιδιαίτερα στις νέες λειτουργίες που επιτελεί η Γεωργία και η Γεωργή. Είμαστε ευγνώμων προ την Αυστριακή Μελλοντική Προεδρία για τη σημαντική πρόταση μεταρρύθμιση ε, που έκανε ο Φρανς Φίσλερ όταν ήταν Επίτροπος Γεωργίας σε ό,τι αφορά ε, τη στήριξη της τοπικής παραγωγής και των τοπικών κοινοτήτων και την ισορροπημένη εδαφική συνοχή. Επίσης, πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της κοινή γεωργικής πολιτικής και να γίνει πιο εξορροπημένη η διαχείριση της ε, ΚΑΠ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα επανεθνικοποιήσουμε την κοινή γεωρική πολιτική. Η πατρίδα μου, η Πολωνία, περιμένει μια κοινωνική κοινή γεωρική πολιτική, αλληλέγγυα γεωρική πολιτική προ όλε τι χώρε ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου και βρίσκονται, στην Ανατολική ή τη Δυτική Ευρώπη. Επίση, ε, τονίζουμε το σημαντικό ρόλο του δεύτερου πυλώνα, της ανάπτυξης της υπαίθρου δηλαδή, που είναι ιδιαίτερα σημαντικός πυλώνας για την Πολωνία. Και η πολιτική του δεύτερου πυλώνα θα πρέπει να στηριχθεί με κάποια κονδύλια του Ταμείου Συνοχής. Αυτό είναι ε, ιδιαίτερα σημαντικό για την Πολωνία. Και επαναλαμβάνω, η θέση της πολωνικής κυβέρνησης τη χάνει της πλήρους υποστήριξης της Πολωνικής Βουλής. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βέσλικ από τη Σουηδία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή είναι πολύ σημαντική. Και εμείς στη Σουηδία θεωρούμε ότι η κοινή αγροτική πολιτική είναι ένα ζήτημα εξαιρετικά σημαντικό και ε, ένα εργαλείο που θα πρέπει να αξιοποιήσουμε για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Κατά την άποψή μας θα πρέπει να μειωθούν οι άμεσες ενισχύσεις και να πάμε περισσότερο προς μέτρα τα οποία προστατεύουν το περιβάλλον, να ε, δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ε, οικολογικοποίηση, γιατί ε, μέχρι στιγμής η κάψη αυτούς τους τομείς δεν τα έχει καταφέρει και τόσο καλά. Για αυτόν τον λόγο λοιπόν θεωρούμε ότι τα μέτρα της ΚΑΠ θα πρέπει να έχουν άμεση σύνδεση με τους περιβαλλοντικούς στόχους. Οι ενισχύσεις δηλαδή, να είναι άμεσα συνδεδεμένες με τους περιβαλλοντικούς στόχους και με άλλους παρόμοιους στόχους όπως για παράδειγμα η καταπολέμηση της αυξημένης μικροβιακής αντοχής ή η ευζοία των ζώων. θεωρούμε από αυτά που ακούμε μέχρι στιγμής ότι η στρατηγική όσον αφορά την αγροτική πολιτική είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Δεν είναι πάντοτε βέβαιο ότι η αύξηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού θα οδηγήσει σε καλύτερη επίτευξη των ε, ε, στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελέγχθη ότι δεν θα πρέπει να πληρώσουν οι αγρότες το λογαριασμό του Brexit. Βέβαια υπάρχει το πρόβλημα ότι πολύ λίγοι θέλουν να πληρώσουν τελικά το λογαριασμό του Brexit. Ούτε καν στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θέλουν να πληρώσουν το λογαριασμό του Brexit. Και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα έχει επιπτώσεις για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Κούσμικ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι κάπου μετά το 2020 θα πρέπει όχι μόνο να διατηρηθεί αλλά και να ενισχυθεί και να λάβει υπόψη την επιστηστική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να την εξασφαλίζει επίσης, να είναι φιλική προς το περιβάλλον, να ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική κατάσταση της υπαίθρου, να μην συνιστά διακρίση βάρος ε, κάποιων κρατών μελών ή γεωργών κάποιων κρατών μελών και φυσικά θα πρέπει να απλοποιηθεί. Δεύτερον, η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να προβλέπει δίκαιη εξίσωση των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου θα πρέπει να στηρίξει ε, την διαφοροποίηση μεταξύ των αγροτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, τα κονδύλια της αγροτικής ανάπτυξης θα πρέπει να διαφυλαχθούν και σε μεγάλο βαθμό να ε, δίνονται άμεσα στους γεωργούς. Λαμβάνοντας υπόψη την ε, τα χαρακτηριστικά και την ανάπτυξη των γεωρικών εκμεταλλεύσεων. Επίσης, ε, θα πρέπει να στηρίξουμε την οικολογική, βιολογική παραγωγή και να ενισχύσουμε τις προδιαγραφές για την καλή διαβίωση των ζώων. Η στήριξη του αγροεπιστηστικού τομέα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την ανάγκη στήριξη της τοπικής παραγωγής. Θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στη βραχή αλυσίδα ε, εφοδιασμού και στις τοπικές αλυσίδες διανομής. Και σε ό,τι αφορά την έκκληση του Επιτρόπου Χόγκαν, που μας υπενθύμησε ότι θα πρέπει να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν σε αύξηση της, ε, θετικής, ε, της εθνικής τους ε, συνεισφοράς, η πολωνική κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να αυξήσει την εθνική της συνεισφορά άνω του 1,1% του ΕΠ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στανκίχας από τη Λιθουανία. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι. Το Εθνικό Κοινοβούλιο της Λιθουανίας εξέδωσε τη θέση του στην Εαρινή Σύνοδο του 2017. Θέσεις λοιπόν για την κοινή γεωργική πολιτική, στις οποίες υπογραμμίστηκε ένα ζήτημα, η ισοδίκαιη αντιμετώπιση. Την ανέφεραν και πολλοί από τους ομιλητές σήμερα. Όταν μιλάμε λοιπόν για πολιτική ενισχύσεων, πληρωμών, αυτή πρέπει να είναι δίκαιη, ισοδίκαιη, δεν πρέπει να υπάρξει, να προκύψει στρέβλωση ανταγωνισμού. Οι χώρες ε, της Βαλτικής είναι μεταξύ εκείνων που, έχουν, που λαμβάνουν τα μικρότερα ποσά πληρωμών. Πολλοί πολίτες μας εγκαταλείπουν τις χώρες μας. Γι' αυτό λοιπόν στις ε, στη νέα προγραμματική περίοδο πρέπει οι πλήρωμες να στηρίζονται στην αρχή της ισότητας της μεταχείρισης. Αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει η χρηματοδότηση του προϋπολογισμού γενικά να περιοριστεί. Θα περιοριστεί αναγκαστικά λόγω του Brexit. Θα είναι όμως πολύ δύσκολο να ε, διαφυλαχθεί αυτή η αρχή της ίσης μεταχείρισης και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μην περισταλεί ο προπολογισμό για τη γεωργία. Να μην περικοπεί. Πρέπει να διαφυτηρήσει τον ε, όγκο του αυτός ο προϋπολογισμός, τον όγκο του χρηματοδοτικό. Βεβαίω θα πρέπει να κοιτάξουμε τα πράγματα όλα εξ αρχή στην κυνηγιορική πολιτική. Δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μόνο σε ιστορικές αναφορές. Οι χώρες ε, της Βαλτικής, οι χώρες του Βίζεγκρατ. Σημειώνουμε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η δική τους κατάσταση με βάση τις αρχές της ίσης μεταχείρισης. Γιατί αυτή είναι και η βάση και η βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν μιλούμε για τον προπολογισμό, ας μην ξεχνούμε ότι ο προπολογισμό ε, και το ΠΔΠ ήταν κατά 11% λιγότερο, δηλαδή κατά 28 δις λιγότερο, σε σχέση με το προηγούμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Οπότε ήδη μιλούμε για χαμηλότερο προπολογισμό σε αυτό το Πολιτες δημοσιονομικό πλαίσιο σε σχέση με το προηγούμενο. Και μάλιστα σε σταθερές τιμέ αυτή η μείωση κατά 10%. Ο κύριος Βαλντίνεκ από την Τσεχία. Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η Τσεχία έχει υποστηρίξει ε, διαχρονικά την κοινή αγροτική πολιτική και εμείς είμαστε έτοιμοι να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση που χρειάζεται έτσι ώστε τελικά να μην υπάρξουν ουσιαστικές περικοπές στα χρήματα που φτάνουν στους αγρότες. Όμως, έχουμε μια σημαντική διαφωνία. Εμείς δεν συμφωνούμε με την προτινόμενη αρχή της του υποχρεωτικού ανώτατου ορίου, του υποχρεωτικού κάπινγκ. Αυτό δεν μας το έχει εξηγήσει ποτέ κανείς γιατί πρέπει να είναι υποχρεωτικό και τι βοηθάει. Έχουμε επιχειρήσεις ε, των οποίων η ιδιοκτησία είναι κατανεμημένη σε 150.000 γεωργούς ορισμένες περιπτώσεις. Ε, φανταστείτε γιατί γραφειοκρατικό άχθος μιλάμε. Ε, ακούμε αυτές τις προτάσεις από τον Επίτροπο Χόγκαν, από τον Υπουργό της Βουλγαρίας, οι οποίοι και εκείνοι αναγνωρίζουν ότι θα χρειαστεί ε, μεγαλύτερη ευελιξία, δηλαδή τα κράτη-μέλη να έχουν ε, μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια. Λέγεται επίσης ότι θα πρέπει να φροντίσουμε οι επιδοτήσεις να μην φτάνουν ποτέ στα χέρια ατόμων που δεν είναι ενεργοί αγρότε. Θέλουμε να φτάνουν οι επιδοτήσει μόνο στου ενεργού αγρότες, λέμε, και στου νέου αγρότε. Αν είναι έτσι όμω, γιατί να είναι υποχρεωτικό το κάπινγκ, γιατί να είναι υποχρεωτικό το ανώτατο όριο τη επιδότηση. Ο Υπουργό είπε ότι, ο επίτροπο μάλλον είπε ότι αυτό μπορεί να συμβεί, μπορεί να χρειάζεται, επειδή οι μεγάλε αγροτικέ εκμεταλλεύσει καταφέρνουν με οικονομίε κλίμακο να μειώσουν το κόστο του. Ευτυχώς μιλούμε για, το, για την κλίμακα απασχόλησης, ε, για το επίπεδο απασχόλησης και λέμε να αξιοποιήσουμε την κλίμακα της παραγωγής. Κυρία Μίλλερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η κοινή γεωργική πολιτική είναι ιστορία επιτυχίας, πρέπει να συνεχιστεί. Όλοι εδώ στηρίζουμε την παραγωγή καλών ποιοτικών τροφίμων, την επιστηστική ασφάλεια στην Ευρώπη. Ωστόσο, βέβαια, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ιδιαίτερες ανησυχίες μας ε, γεννούν οι διαφορετικές αντιλήψεις και διαφορετικές μέθοδοι υλοποίησης αυτών των ε, κανόνων της κοινής πολιτικής από τα κράτη-μέλη δεν μπορούσα να φανταστώ ότι η Γερμανία είναι η μόνη χώρα που έχει αποσυνδεδεμένες πληρωμές και ότι όλα τα άλλα κράτη-μέλη έχουν διατηρήσει τις συνδεδεμένες πρημοδοτήσεις. Και ότι μάλιστα δεν είναι καν διατεθειμένα στο μέλλον να τις αποσυνδέσουν. Επίσης, δύσκολο θα είναι και το ζήτημα της εισαγωγής του κοινωνικού παράγοντα, της ε, κοινωνικής ενιστώσας στα προγράμματα. Δηλαδή η διαφύλαξη του κοινωνικού ιστού χάρη στη γεωργία, στην Ήπεθρο συγκεκριμένα. Εδώ νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με συνιστώσεις που ε, θα διευκολύνουν την ε, πληρωμή των ε, γεωργικών ενισχύσεων. Και επίσης θα πρέπει να φροντίσουμε τα κριτήρια των ε, κρατών μελών αλλά και του λιανικού εμπορίου να είναι διατυπωμένα κατά τρόπον ώστε να μην οδηγούν σε στρεβλώσεις. Θα πρέπει να υπάρξει ένας κατάλογος αυτών των κριτηρίων παράλληλος βέβαια με την νομοθεσία και τους κανόνες που ισχύουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι δυνατότητες που θα επιτρέψουν και θα εξασφαλίσουν μια προοπτική στους νέους, στους νέους γεωργούς. Είμαι πεπισμένη ότι εμείς εδώ από το Κοινοβούλιο έχουμε όλη τη βούληση να εξασφαλίσουμε συνθήκες πλαισίου για τους νέους αυτούς γεωργούς. Θα πρέπει όμως και τα κρατη και οι εκπρόσωποι τους εδώ, οι να μεριμνήσουν ώστε να μην ενισχυθεί η γραφειοκρατία υπερβολικά στα εθνικά συστήματα. Όταν μιλούμε για τις ενισχύσεις σε σχέση με την παραγωγή, θα πρέπει να Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι μόνο 13 με 15% του προπολογισμού μπορεί να αφιερώνεται με βάση το τρέχον πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο από τον προπολογισμό, μόνο 13 με 15% στις ενισχύσεις της παραγωγής. Και μόνο για εκείνες τις παραγωγές για τις που υπάρχουν σε συγκεκριμένο παράρτημα. Γι' αυτό μιλάμε για συγκεκριμένα κλίμακες παραγωγής. Τώρα για την επιτυχία του ΚΑΠ, όταν ο γεωργός λαμβάνει 50% των ε, ε, δαπανών από άλλες ε, επαγγελματικές οργανώσεις, δεν νομίζω ότι είναι και μεγάλη επιτυχία. Θα πρέπει να, να έχουμε υπόψη και το επίπεδο του γεωργού όταν μιλούμε για την επιτυχία της ΚΑΠ. Ο κύριος Δίας από την Πορτογαλία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ και Εθνική Βουλευτέ. Όταν μιλούμε για την ΚΑΠ που έχει πολλές συνιστώσεις και πυλώνες, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε τον αντίκτυπό τη στη Γεωργιακή, ιδιαίτερα στην Πορτογαλική. 400.000 είναι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 90% ε, των γαλακτοκομικών ε, εκμεταλλεύσεων βρίσκονται στην υπηρετική Πορτογαλία, αλλά έχουμε μεγάλη αδικία στην κατανομή των άμεσων ενισχύσεων. Ένα μικρό ποσοστό λαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα των ενισχύσεων. Επίσης είχαμε τραγικές πυρκαγιές κάτι που κατέστρεψαν τρία, τρεις δεκαετίες ολοκλήρωσης της Πορτογαλικής Γεωργίας. η Γεωργία θα μπορούσε να, να αποτελεί σημαντική μόχλευση για την οικονομική άνθηση και ιδιαίτερα των μικρών εκμεταλλεύσεων, γιατί αυτές οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις ε, έχουν βιώσει με παραγωγή ποιοτικών τροφίμων, διαφυλάσσουν το περιβάλλον και κρατούν τη ζωή στην ύπεθρο ζωντανή. Αυτή την γεωργία θα πρέπει να στηρίξουμε και να αναπτύξουμε. Οπότε χρειάζονται κάποια μέτρα ελέγχου της αγοράς ε, που θα προωθούν τις παραγωγές σε όλες τις περιφέρειες και τις χώρες. Και θα πρέπει να έχουμε αντίστροφη εξισορρόπηση της αλυσίδα και να μην έχουν την απόλυτη εξουσία οι αλυσίδε διανομής, αλλά περισσότερο οι παραγωγές Και Γιώργη, είναι απαράδεκτο να ε, πληρώνουμε ενισχύσει σε γεωργούς που είναι ανενεργοί, που είναι μόνο στα χαρτιά, που δεν ε, παράγουν ένα γραμμάριο ε, τροφίμων. Θα πρέπει να ενισχύονται οι ενεργοί γεωργοί. Θέλουμε μια ζωντανή πεθρό και αυτό θα το καταφέρουμε να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες γεωργικές επιχειρήσεις και τις οικογενειακές γεωργικέ εκμεταλλεύσεις. Ευχαριστώ.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 Tervehdys Suomen parlamentista. Ruoantuotannon kannat... Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας μεταφέρω τον χαιρετισμό του Φιλανδικού Κοινοβουλίου. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι η, πώς θα κρατήσουμε τους νέους στην ε, γεωργία, πώς θα ε, αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες προς αυτό. Γνωρίζουμε ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον της γεωργικής οικονομίας έχει αλλάξει. Έχουμε νέες δομές πλέον και δεν μπορούν όλες οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε ε, τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις να τα καταφέρουν και στο παρόν και στο σύντομο χρονικό μέλλον. Από την πλευρά της Φινλανδίας, εγώ θα ήθελα να επισημάνω ότι ε, ασκείται κριτική στις άμεσες ενισχύσεις και το πώς αυτές συνδέονται με ιδιαιτερότητες τοπικές εθνικές. Η Φιλανδία γνωρίζεται ότι οι κλιματολογικές συνθήκες, οι συνθήκες ε, ειδικέ της περιοχής είναι πολύ δυσμενείς. Αλλά θέλουμε να συνεχίσουμε ε, την αγροτική παραγωγή στην Φιλανδία όπως συνέβαινε επί αιώνες και θέλουμε να, συνεχιστεί, να, να συνεχίσει να συμβαίνει και στο μέλλον. Ε, αυτή τη στιγμή ε, εξαιτία ακριβώς των δυσμενών εθνικών συνδικών που οδηγούν σε αυξημένες τιμέ. η υποστήριξη που δίνεται στην Φιλανδία είναι αυξημένη. Έτσι λοιπόν, οι όποιε νέε μέθοδοι θα πρέπει να ε, τα λαμβάνουν και αυτά υπόψη του. Τι διαφορέ δηλαδή που υπάρχουν από κράτο μέλος σε κράτο μέλος, και θα ήθελα, εάν μπορείτε, να μου δώσετε κάποιε περισσότερε πληροφορίε σε σχέση με το τι θα γίνει με τι άμεσε πληρωμέ για, για, για περιοχέ τη Ευρώπη οι οποίε αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα δυσμενεί συνθήκε. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω σε ποιον απευθύνεται την ερώτησή σα. Αν την απευθύνεται σε μένα, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συνθήκε ε, ε, οι αντίξωε συνθήκες ε, στη γεωρική εκμετάλλευση, ποιότητα του εδάφου, αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη γιατί είναι σημαντικοί παράγοντε που επηρεάζουν την παραγωγή και άρα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και στι άμεσε ενισχύσει. Κυρία Σένρα. Σα ευχαριστώ. Μιλούμε όλο το απόγευμα για αποδοτικότητα και για εγγύηση του γεωργικού εισοδήματο για του αγρότε και τις αγρότησέ μα. Αλλά παραλείψαμε δύο κομβικά θέματα που πιστεύω ότι θα πρέπει να επισημαθούν το θέμα των τιμών που καταβάλλονται στον παραγωγό και που θα πρέπει να είναι δίκαιες τιμές, να αμείβουν τον Γιώργο για τον κόπο του και το δεύτερο είναι η ρύθμιση της παραγωγής και των αγορών. Πιστεύω ότι αν δεν ε, επικεντρώσουμε την πολιτική συζήτηση σε αυτές τις δύο πτυχές, δύσκολα θα εξασφαλίσουμε την επιβίωση των αγροτών και των αγροτησών μας. Και αυτό φυσικά έχει μεγάλη σχέση και με την ηλικιακή ανανέωση στη Γεωργία. Ένα άλλο πρόβλημα που συνεχώς αναφέρουμε. Αν δεν δώσουμε εγγυήσει ε, για αξιοπρεπή βιοπορισμό από την Γεωργία, πώς θα προσελκύσουμε νέους στις γεωργικές δραστηριότητε. Επίσης, ε, θα ήθελα να επισημάνω και ένα άλλο στοιχείο που επίσης παραλείπεται ή αποσιωπάται σχεδόν πάντα. Τα δικαιώματα των γυναικών στην Ήπεθρο, των αγροτησών, γιατί είναι φανή η διάκριση της κάπη βάρος των ε, γυναικών στη Γεωργία. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε την, τη συνειδιοκτησία στις γεωργικέ εκμεταλλεύσεις μεταξύ των δύο συζύγων και να εξασφαλίσουμε ισότητα δικαιωμάτων στις γυναίκες που απασχολούνται στι γεωργικέ εκμεταλλεύσεις. Επίση, θα ήθελα να μιλήσω λίγο και για τι εμπορικέ συμφωνίε οι συνέπειες ε, των εμπορικών συμφωνιών στις ε, μικρομεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι αρνητικές ε, και είναι αρνητικές συνέπειες και για τους γεωργούς Ευρωπαϊκής Ένωσης, του μικρομεσαίους και για τους γεωργούς των τρίτων χωρών. Πρόσφατα πήγαμε στη Βραζιλία και είδαμε με τα μάτια μας τι μας περιμένει και τι περιμένει την κτηνοτροφία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα την ε, γελαδοτροφία μετά τη Συμφωνία του Μερκοσούρ. Και να μην ξεχνούμε και το περιβάλλον. Ε, η κυκλοφορία στον πλανήτη προϊόντων από την άλλη άκρη του κόσμου, ενώ θα μπορούσαμε να δώσουμε έμφαση στι τοπικέ αλυσίδε παραγωγής, ε, αυξάνουν το αποτύπωμα του άνθρακα και είναι πολύ επιζήμιες για το περιβάλλον. Αυτό να το βαλάβουμε υπόψη όταν μιλούμε για βιωσιμότητα. Να μιλήσουμε δηλαδή και για το μοντέλο παραγωγή και για το μοντέλο εμπορευματοποίηση των τροφίμων. Ευχαριστώ. Ναι, είχαμε κάποιες, κάποιο κανονισμό για τις, και τις γαλακτοκομικές ποσοστώσεις και παρόλα αυτά είχαμε κρίση στο γαλακτοκομικό τομέα, οπότε δεν τα λύνουμε όλα με τη ρύθμιση. Ο κύριος Βικρόπ από την Ολλανδία. Thank you, Mr. President. Uh, on behalf... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συνεχίσω στα Ολλανδικά. Μέρος λοιπόν της Επιτροπής Γεωργίας του Ολλανδικού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να εκφράσω μια ανησυχία που μας έχει γεννηθεί σε σχέση με την οκολαπτόμενη νέα ΚΑΠ. Είναι η εξής απορία. Πώς μπορούμε να εγγυηθούμε ότι σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι συμφωνίες που θα επιτευχθούν, οι κοινέ μας συμφωνίες που θα θέσουν τους κοινού μας στόχους, θα εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο. Και πώς θα εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν διπλά μέτρα και, ε, δύο μέτρα και δύο σταθμά σε, από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό μπορεί να το εξασφαλίσει. Ευχαριστώ. Κυρία Καφαντάρη από την Ελλάδα σημαντική η σημερινή πρωτοβουλία να συζητηθεί το θέμα της ΚΑΠ, της κοινή αγροτικής πολιτικής, εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Ε, θα έλεγα καταρχάς ότι η κοινή αγροτική πολιτική πρέπει να παραμείνει κοινή πολιτική ολοκληρωμένη που θα εγγυάται τη διασφάλιση αγροτικού εισοδήματος κοινωνική συνοχή περιφερειακή ανάπτυξη προστασία του περιβάλλοντος και προστασία των καταναλωτών. θα συμφωνήσω δε με αυτό που ο επίτροπος χόγκαν ανέφερε αρχικά ότι άλλο μοντέλο αγροτικής πολιτικής στο βορρά και άλλο στο νότο και ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά και τη χώρα μου την ελλάδα η οποία άλλο μοντέλο αγροτικής πολιτικής μπορεί να έχει σε σχέση με τη Φιλανδία όπως ανέφερε ενδεικτικά ο ίδιος. Διότι πραγματικά βασικοί τομείς οι οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι σε κάθε χώρα τα θέματα της νησιωτικότητας, τα θέματα των ορεινών περιοχών και οι άμεσες ενισχύσεις θα μπορούν να εστιάσουν σε μικρές μεσαίες εκμεταλλεύσεις, σε εκμεταλλεύσεις όπως είπα πριν μειονεκτικών νησιωτικών περιοχών, σε νέους που θέλουν να μπουν στον τομέα της αγροτικής οικονομίας και σε τομείς που το εισόδημα παραμένει χαμηλό και η διατήρησή του πρέπει να υπάρχει. Αυτό το οποίο όμως θέλω να πω είναι ότι πολλές είναι οι προκλήσεις οι οποίες αντιμετωπίζει το αγροτικό, η αγροτική οικονομία, να το πω συγκεκριμένα σήμερα. Μία από αυτές είναι και τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, που είναι σημαντικό με τους κινδύνους οι οποίοι υπάρχουν. Γι' αυτό χρειάζονται και νέα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου. Ε, ένα σοβαρό τομέα είναι ο τομέας του νερού, που πρέπει να διασφαλίσουμε μέσα από συγκεκριμένη πολιτική ε, και την ποιότητα αλλά και την ποσότητα λόγω και της κλιματικής αλλαγής που παίζει σημαντικό ρόλο. Έχει μεγάλη σημασία η χρήση των νέων τεχνολογιών, η ψηφιοποίηση καθώς και επενδύσεις στην καινοτομία. Κλείνοντας, θα έλεγα ότι για την ΚΑΠ εμείς ως Ελλάδα πιστεύουμε ότι πρέπει να διατηρηθεί στα επίπεδα που υπάρχουν η χρηματοδότηση, τουλάχιστον σε αυτά τα επίπεδα. Είμαστε υπέρ των δύο πυλώνων, άμεσες ενισχύσεις αγροτική ανάπτυξη και επειδή αναφέρθηκε κάτι για την εξωτερική σύγκληση άμεσων ενισχύσεων, πρέπει να το ξαναδούει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η αναεκτάριο ενίσχυση δεν μπορεί να αποτελεί τη μοναδική παράμετρο για μια συζήτηση για την εξωτερική σύγκληση των άμεσων ενισχύσεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μιλήσατε για την διαφοροποίηση, την πολυμορφία της ευρωπαϊκής γεωργίας και αναφέρετε τα παραδείγματα της Ελλάδας και της Φιλανδίας. Είναι πολύ διαφορετικές ε, οι γεωργίες γι' αυτό. Σε τέτοια πολυμορφία, όταν έχουμε κοινή γεωργική πολιτική, θα πρέπει να δούμε τι ε, μέτρα θα χρησιμοποιήσουμε και τι μηχανισμούς για να στηρίξουμε τόσο διαφορετικά είδη και το πρόβλημα του νερού είναι πολύ σημαντικό, αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι και το θέμα της ενέργειας. Κύριος Χόισλινγκ, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα για την ευκαιρία για αυτή τη συζήτηση. Χαίρομαι που ε, έρχεται εδώ ένας υπουργό Γεωργίας για να πει ότι πρέπει να μείνει ο προπολογισμό της Γεωργίας όπως έχει. Ίσως ήταν καλό και οι υπουργοί Γεωργίας να αρχίσουν να μιλούν με τους πρωθυπουργού τους για να λυθούν τα προβλήματά μας ε, ως προς τον προϋπολογισμό της Γεωργίας. Ε, πάντως μπορεί να είναι το εκτάριο ένα μέτρο υπολογισμού και να συνεχιστεί η ενίσχυση να καταβάλλεται με βάση το εκτάριο ή θα πρέπει να κοιτάξουμε αν προσφέρει τον αναμενόμενο, το αναμενόμενο δημόσιο αγαθό η γεωργία, προστασία του περιβάλλοντος, ε, ε, τη θάση της κλιματικής αλλαγής και ούτω καθεξής. Δεν μπορεί να πηγαίνει ένα ποσοστό μέχρι και 80% του προϋπολογισμού της γεωργίας μόνο σε μεγάλες επιχειρήσεις. Πρέπει να στηρίξουμε και τις μικρές. Και επίσης, κάτι που είχα επισημάνει ήδη με την ανακοίνωση της Επιτροπής στο περασμένο φθινόπωρο. Πρέπει συνολικά να δούμε το θέμα της γεωργίας και την προσφορά της. Δεν μπορώ να, μιλώ, να μιλώ για, ε, μια, για ένα άνοιγμα σε παραγωγή από όλο τον κόσμο τη αγορά μας και από την άλλη να μιλούμε για την ευρωπαϊκή παραγωγή σε μόνο ποιότητα. Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τις χώρες της Μερκοσούρ. Δεν μπορούμε να ανοίγουμε τι δηλαδή, τις αγορές μας με την απελευθέρωσή τους ε, σε ξένα προϊόντα και ταυτόχρονα προσπαθούμε να διαφυλάξουμε την ποιότητα των δικών μα ε, προϊόντων. Δεν στέκει αυτό. Περιθώριο για τα κράτη-μέλη. Δεύτερο, πρέπει να πω ότι αισθάνομαι μεγάλη δυσφορία ότι δεν υπάρχει κοινή γεωργική πολιτική ακόμα με ε, όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε πίσω μα ε, τη λειτουργία του συστήματο κοινή γεωργική πολιτική. Και τώρα ε, είναι σαν να μα λένε τα κράτη-μέλη α, κοιτάξτε, δεν γίνεται, δεν το εφαρμόζαμε μέχρι τώρα. Δεν θέλουμε άλλη κοινή γεωργική πολιτική όμω. Μα όχι, το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε αρκετή γεωργική πολιτική. Γιατί αν περάσουν αυτές οι αρμοδιότητες στα χέρια των κρατών μελών, μπορούμε να αποχαιρετήσουμε την κοινή γεωργική πολιτική. Θα την δινάξουμε στον αέρα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να έχουμε μια γνήσια κοινή γεωργική πολιτική και να μην αφήσουμε να διαλυθεί. Ίσως έχουμε κοινή γεωργική πολιτική, αλλά μια ελαστική ευέλικτη κοινή πολιτική που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών. Ο κύριος Μπεκχάους από τη Γερμανία. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την ε, πρόσκληση και την ευκαιρία για συμμετοχή στη συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, προέρχομαι από Ομόσπονδο Κρατήριο της ε, Γερμανίας και έχω τη δική μου θέση για το πώς θα πρέπει να εξελιχθεί η κοινή πολιτική. Να σα πω λοιπόν ποιοι είναι οι κύριοι πυλώνε αυτή τη ιδέα. Πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε ένα τετράγωνο που θα συνδυάζει οικονομία, οικολογία, κοινωνική υπευθυνότητα και ε, γεωργική πολιτική, πολιτική ε, της υπαίθρου. Και εδώ νομίζω ότι η κοινή γεωργική πολιτική έχει στεφθεί με επιτυχία στην Ευρώπη. Πρέπει να τη στηρίξουμε και με παραπάνω μέτρα Ξέρουμε ότι οι στόχοι περιβαλλοντικοί της Ευρώπης δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί. Η οδηγία για τα ύδατα, για τα νήτρικα και νήτρο, διάφοροι στόχοι που δεν έχουν υλοποιηθεί. Ενώ ξέρουμε ότι μπορεί με την υποστήριξη αυτών των επιπλέον στόχων να εξασφαλιστεί και πρόσθετο εισόδημα για τον Γεωργό και την Ήπεθρο. Έχουμε ένα μοντέλο λοιπόν εξασφαλίσει το οποίο μπορεί εν γέννη στην Ευρώπη να φέρει καλά αποτελέσματα. Έχει αποδειχθεί αυτό και στην πράξη αλλά και στη θεωρία και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό πρέπει να το, έπρεπε να το αναφέρω εδώ. Επίσης, γνωρίζουμε σήμερα ότι το γεωργικό εισόδημα, το εισόδημα γενικά στην Ήπεθρο παρουσιάζει μεγάλες δεκιμάνσεις. Χωρίς τη γεωργία όμως, χωρίς την Ήπεθρο, η Ευρώπη δεν μπορεί να έχει μέλλον. Πρέπει λοιπόν ιδιαίτερα να τη στηρίξουμε. Και αυτό σημαίνει υποστήριξη γενικότερα της κοινωνίας η Γεωργία και η Πέθρος πρέπει να είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε αυτή την πρόοδο. Πιστεύω επίσης ότι έχει καθοριστική σημασία και η ανάληψη πρωτοβουλειών για να ανοίξουμε τις δυνατότητες του μέλλοντος. Ψηφιοποίηση είναι το ένα. Επίσης προοπτικές για δραστηριοποίηση στον χώρο της υπαίθρου των νέων είναι το δεύτερο και σε αυτό νομίζω πρέπει να εξυγχρονιστεί περαιτέρω η πολιτική για τους νέους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να εξυγχρονιστεί, πρέπει να διαφυλάξει την υπαίθρο, πρέπει να φέρει τη γενοτομία στην Ευρώπη και την υπαίθρο και είναι πάρα πολύ σαφές για μένα ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι πρέπει από το χέρι μας για να θέσουμε πλέον ένα τέρμα στην υπερβολική γραφειοκρατία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλώ πρώτα απ' όλα ως αγρότης, αλλά επίσης και ως πρώην υπουργό. Συμμετείχα επί τέσσερα χρόνια στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πιστεύω ότι τα νέα είναι τα εξής. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε είναι η νέα κοινή αγροτική πολιτική να είναι πιο απλή, να έχει λιγότερη γραφειοκρατία. Δεν έχει νόημα να κάνουμε ακόμα μια μεταρρύθμιση τη αγροτική πολιτική, αν δεν τα καταφέρουμε να την απλοποιήσουμε. Γιατί οι αγρότε δεν έχουν καταφέρει ακόμα να συνηθίσουν τι τρέχουσε αλλαγέ, τη σημερινή ΚΑΠ. Ε, θα ήθελα να πω ότι για την Τσεχία είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα του ανώτατου ορίου έχουμε μικρές εκμεταλλεύσεις, ακόμα και η γυναίκα μου έχει 20 εκτάρια αρρώσιμης γης. Οι μικρές εκμεταλλεύσεις λοιπόν στην Τσεχία είναι πολύ άριθμες. Δεν αντιλαμβάνομαι λοιπόν γιατί ο Επίτροπος Χόγκεν ε, ε, ε, έρχεται και, και, κάνει αυτή την πρόταση, γιατί προσπαθεί να αλλάξει αυτή την παράμετρο. Εξάλλου είναι ένα ζήτημα όχι προπολογισμού, είναι ζήτημα γεωργία, είναι ένα ζήτημα αρμενότητα του κυρίου Χόγκαν. Βεβαίω να αντιληφθώ μια συζήτηση σε σχέση με το πώ αξιοποιείται η επιδότηση του. Μα ενδιαφέρει τι τα κάνει τα χρήματα που παίρνει ο αγρότη, πώ σέβεται το περιβάλλον. Όμως γνωρίζουμε ότι το 65% ε, των αποσχολουμένων στη χώρα μου εργάζονται στην αγροτική οικονομία, ότι έχουμε ποσοστά άνω του 80% από τις μικρές εκμεταλλεύσεις που παράγουν γάλα. Ε, και γνωρίζουμε επίση ότι υπάρχουν πολλέ και διαφορετικέ προσεγγίσεις που μπορεί να ακολουθήσει μια εκμετάλλευση όσον αφορά τη χρήση των σπόρων, όσον αφορά την κυριότητα του εδάφου, κτλ. Αφού λοιπόν μιλούμε για επικουρικότητα, α αφήσουμε τα κράτη-μέλη να επιλέξουν τι λειτουργεί καλύτερα για αυτά και ειδικά αυτό α ισχύσει για το κάπινγκ, για το ανώτατο όριο. Αυτά τα 25 εκτάρια που έχει η γυναίκα σα την κάνουν πλούσια ή φτωχή. Ο κύριος Άγνιο. Uh, Ευχαριστώ. Εμένα με ανησυχεί ο αντίκτυπος που έχει η φτωχη ο κύριο αγνιο ευχαριστω εμενα με ανησυχει ο αντικτυπος που εχει η νομοθεσια γιατί αυτό είναι το αντικείμενο των πολιτικών. Και με εντυπωσίασε το γεγονό ότι δεν ε, μάλλον με εντυπωσίασε το γεγονό ότι συζητήσαμε με τέτοιον τρόπο για τα να πολλέ φορέ χωρί λόγο. Η γλυφωσάτη αυτή τη στιγμή η χρήση της ε, κρέμεται από μια κλωστή. Εάν τελικά απαγορευτεί θα, ε, γυρίσουν, θα έχουμε τεράστιο γύρασμα για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα επανέλθει τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια της Βουλγαρικής Προεδρίας, το οποίο είναι το ερώτημα της χρήσης. Νέο νοικοτινοειδών σε ε, καλλιέργειες οι οποίες δεν πρόκειται να να, να, συλλεγούν. Ε, ε, όλες αυτά, όλα αυτά τα μέτρα προσπαθούν να μας πούν ότι πρέπει να σταματήσουμε τη χρήση των χημικών, λένε. Όμως έχουμε βιολογική γεωργία η οποία χρησιμοποιεί νόσεις του θείου ε, ε ως στελεπάσματα και αυτό είναι εξίσου επιβλαβές. Εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα. Δεν υπάρχει μια τεράστια λοιπόν αντίθεση, ε, αναντιστοιχεία στις πολιτικές μας. Το ίδιο πιστεύω ε, είναι ε, εξίσου σημαντικό πιστεύω ότι είναι το ζήτημα της καταπολέμησης της μικροβιακής αντοχής. Εδώ είναι κάτι το οποίο θα επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους. Πιστεύω λοιπόν ότι υπό τον πυλώνα 2 θα πρέπει να κρατήσουμε στην ακρικά πια χρήματα για την βοήθεια, την ενίσχυση των κτηνοτρόφων των πουλερικών σε τέτοιε περιπτώσει επιδημιών. Αυτό είναι, το, να έχουμε τέτοιου τύπου ε, μέτρα ενίσχυσης σε έκτακτε καταστάσει είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για την α, στρεματική αποζημίωση, για το, το, συγκεκριμένα μέτρα για τους νέους αγρότε. Εγώ σα μιλώ για ζητήματα τα οποία θα έχουν πολύ μεγαλύτερο και ευρύτερο αντίκτυπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Βιγκριέβα. Madame Vingrieva. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινούμε τη συζήτηση για μια νέα κοινή γεωργική πολιτική. θεμενή αξία της γεωργίας είναι μεταξύ άλλων η παραγωγή τροφής για τον πολίτη με καινοτόμες μεθόδους. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια πολιτική στραμμένη σε αποτελέσματα μέσα από τις μεθόδους που εξασφαλίζουν θεμενή αξία. Οι στόχοι της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής είναι σωστοί και τους υποστηρίζουμε. Στόχος είναι να καταστεί ανθεκτικός, καινοτόμος, ο γεωργικός τομέας, να διασφαλιστεί η γεωργική παραγωγή, να ενισχυθεί η κοινωνική και οικονομική ευρωστία των ε, περιοχών της υπαίθρου. Πρέπει να ετοιμάσουμε τη γεωργία μας για τις νέες προκλήσεις και αυτό απαιτεί απλούστευση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Εν των ε, διεθνών μας ε, ευθυνών πρέπει να έχουμε και φιλόδοξους στόχους για την προστασία του περιβάλλοντος. Πρέπει να ενισχύσουμε και να προωθήσουμε μια βιώσιμη γεωργική παραγωγή. Πολιτική για τη γεωργία, αποτελεσματική και χρήσιμη για όλους. Υποστηρίζουμε λοιπόν το στόχο της ανάπτυξης της βιοοικονομίας, της κυκλικής οικονομίας και κάθε δραστηριότητας που σχετίζονται με αυτές. έτσι ώστε να ε, καταστούν οι γεωργικές δραστηριότητες πιο ανθεκτικές στους διαφόρους ε, περιβαλλοντικούς ε, παράγοντες. Αυτό με γνώμονα τη διαφύλαξη της ασφάλειας των, προφήμων, των τροφίμων, των, του περιβάλλοντος και πιστεύω ότι θα πρέπει αυτοί οι παράγοντες να λαμβάνονται υπόψη στη Νέα Κουγουπού και έτσι να προωθηθεί και πιο σύντομη αλυσίδα επιστηστική αλλά και ποιότητα. Ο κύριος Καρμό από την Πορτογαλία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, στην Πορτογαλία υπάρχει μεγάλη εθνική συνένεση σε ό,τι αφορά τους δύο πυλώνες της ΚΑΠ. Η διαφύλαξη του γεωργικού προπολογισμού είναι, προφανή. είναι προφανής θα πρέπει να παραμείνει αλόβητο ο γεωργικό προπολογισμό και η κοινή γεωργική πολιτική που έχει θεμελιώδη σημασία για την ε, κοινωνική συνοχή και η οικονομική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, η ΚΑΠ θα πρέπει να έχει και περιβαλλοντικά κριτήρια στον συνυπολογισμό των άμεσων ενισχύσεων. Αυτό είναι κέριο και αυτό έχει σημασία και για την Ήπεθρο και ενώπιση των κλιματικών αλλαγών και η προσπάθεια Αναχέτηση της απερίμωσης αλλά και στήριξης του αγροτικού κόσμου, ιδιαίτερα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχει στη Μεσογειακή ζώνη. Αυτό είναι βασικός παράγοντας για την κλίδα κατανομής των κονδυλίων της κοινή γεωργικής πολιτικής. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σουλουαζό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, από τη συνάδελφη. Το πρόβλημα της ΣΚΑΠ ουσιαστικά είναι ότι δεν έχουμε μια επαρκή αποζημίωση της εργασίας των παραγωγών, των αγροτών. Αυτή τη στιγμή έχουμε ε, παραγωγούς οι οποίοι πολλούν κάτω τη τιμή του κόστους. Και πρέπει να δούμε πώς στεκόμαστε στην παγκόσμια αγορά. Θα σας αναφέρω ενδεικτικά ότι για την σκόνη γάλακτος η τιμές που πληρώνουν δε οι παραγωγοί ε, είναι κάτω ε, ε, δεν ανταποκρίνονται στα κόστη των παραγωγών. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας απαντάει ότι οποιοδήποτε παρέμβαση δεν μπορεί παρά να καθυστερήσει τρία χρόνια. Μπορούν όμως να το περιμένουν αυτό. Θα πρέπει να περιμένουμε ότι πολλοί από αυτούς τους παραγωγούς θα αντιμετωπίσουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ακόμα και χρεοκοπίες θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτέ οι πολιτικέ σε σχέση με τον ανταγωνισμό, σε σχέση με την παγκοσμιοποίηση είναι αυτέ που οδηγούν σε δραματικέ καταστάσει του παραγωγού. Τώρα, πιέζουμε με την ΚΑΠ τους παραγωγούς να αυξάνουν την παραγωγή τους και ταυτόχρονα τους ε, καταγγέλουμε και τους κατηγορούμε ότι ευθύνονται ε, για την μόλυνση. Αντιθέτως, οι παραγωγοί είναι αυτοί οι οποίοι φροντίζουν τη φύση, δεν είναι αυτοί που μολύνουν, που θα ε, ε πρέπει ε, να εξετάζουμε οποιαδήποτε απαγόρευση φυτοπροστατευτικών μέσων με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί οποιαδήποτε απότομη αλλαγή είναι ε, αδύνατο να την παρακολουθήσουν οι παραγωγοί. Θα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στον τομέα των χημικών και δυστυχώς διαπιστώνω ότι η πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έναντι της χημικής βιομηχανίας είναι σκανδαλώδης, είναι απαράδεκτη. Η ενθάρρυνση που της δείχνει, δίνει. Θα μπορούσα να πω πολλά, θα μπορούσα επίσης να μιλήσω για το διαχειριστικό κόστος, αλλά δεν έχω πολύ χρόνο. Δυστυχώς φοβάμαι ότι οι παραγωγοί έχουν πολλούς λόγους να φοβούνται για το μέλλον τους. Πολύ, σε, πολύ επίκαιρη στιγμή ε, πήρατε το λόγο, την ώρα που έφτανε ο Γενικός ε, Διευθυντής της, Επιτροπής, Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, ο κύριος Πλέτβα, που τον καλωσορίζω θερμά. Τώρα περνάμε στους εθνικούς βουλευτές, ο κύριος Μωρό από τη Γαλλία. Εδώ είμαι. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι. Η εισαγωγική τοποθέτηση του Επιτρόπου Χόγκαν μάλλον μα ε, ανησυχεί παρά μα καθησυχάζει και δεν εκφράζω την πλειοψηφία τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Εδώ βλέπουμε ένα κίνδυνο μεγαλύτερη επικράτηση των τεχνοκρατών στην κοινωνική πολιτική από ό,τι βλέπουμε στι διαπραγματεύσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κρατών μελών. Παρα... Μπαίνει στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου πράγμα παράδεκτο για μα. Υπάρχει βεβαίω ανάγκη για την επικουρικότητα, αλλά δεν θέλουμε διστρέβλωση ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών εκείνων που θα προστατεύουν προς το περιβάλλον, παραδείγματι από τα άλλα, ή ακόμη και εντό, εντός του ίδιου της ίδιας της επικράτειας των κρατών μελών μπορεί να προκύψει ανταγωνισμός, κάτι το οποίο θα ήταν απαράδεκτο. Χρειάζεται μια γνήσια κοινή γεωργική πολιτική, η πρώτη μελέτη συνεπειών της νέας ε, ΚΑΠ δείχνει μείωση κατά 30% στη χρηματοδότηση βοήου κρέατος και 10 με 15, με 20% στη, στα οποροκυπευτικά. Χαιρετίζω τη δουλειά του Κοινοβουλίου στον κανονισμό Omnibus, τις προσπάθειες για την καταπολέμηση των αθέμητων ε, μέτρων και πρέπει να σταματήσει πλέον αυτή η υπερβολική εισαγωγή τεχνοκρατία, ε, ε, Ελέγχω από τους τεχνοκράτες, αυτή η αποδιάρθρωση ουσιαστικά της ΚΑΠ. Εδώ έχουμε στην Γαλλία ένα σύστημα που επεξεργαζόμαστε για τη διαφύλαξη των τιμών. Χρειάζεται να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα διαφυλάξει από τους διάφορους ε, παράγοντες κινδύνου, είτε είναι αυτό το περιβάλλον, είτε είναι οι ξένες αγορές, την γεωργία μας και όχι ένα σύστημα à la carte. Ευχαριστώ από την Δανία, κύριο Πολ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ασφαλής χρήση των νίκο... νέων Νέο. Γνωρίζουμε ότι είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για την ποιότητα των εδαφών. Χρειαζόμαστε μια ουσιαστική ε, πολιτική με έναν κοινό κατάλογο με πλήρη τεκμηρίωση για την κάθε μια από τις ουσίες σε αυτόν τον κατάλογο και με κοινού δείκτε. Έτσι ώστε να μετρούμε τον αντίκτυπο. Και αναρωτιέμαι πώς, με ποιον τρόπο θα φτιάξουμε αυτούς τους ε, δείκτες, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα που μας δίνει η νέα κάποια να εισαγάγουμε αυτούς τους νέους δείκτες. Υπάρχει συμφωνία των Παρισίων ε, που μπορεί να μας βοηθήσει και ουσιαστικά πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση για το τι παράγουμε και τι καταναλώνουμε. Χρειάζεται να βρεθεί μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στις διαφορετικές μεθόδους παραγωγής. Κάτι που, εάν επιτευχθεί, θα οδηγήσει και σε μείωση της εκπομπής ε, διοξιδίου του άνθρακα και ε, του θερμοκηπίου. Ε, αυτά πρέπει να είναι στοιχεία που θα παραμείνουν στο επίκεντρο της συζήτησης για την πολιτική μας. Ευχαριστώ κύριε Ντελέ. Ε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια, η κοινή γεωργική πολιτική έχει μεγάλη σημασία, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε την πολυμορφία των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι γεωργοί σε σχέση με πριν από 60 χρόνια κατάσταση. Γι' αυτό έχουμε και την ιωστή μεταρρυθμίση της ΚΑΠ, αλλά προσοχή, όποιος βιάζεται σκοντάφτη. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη και το λίγο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι το πέρας ε, ανεπαρκές για μια εμπεριστατωμένη ρύθμιση. Ε, σε σχέση με αυτά που μας είπε ο κύριος Φιλχόγκα, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η Γεωργία είναι τμήμα της λύσης για τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Άλλωστε είναι δική μας ευθύνη να εξασφαλίσουμε την επιστηστική κυριαρχία και ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, η μελλοντική ΚΑΠ θα πρέπει να συμπαρίσταται στους γεωργούς στην προσπάθεια μετάβασής τους προς διπλές επιδόσεις οικονομικές και περιβαλλοντικές ε, και αυτό θα γίνει κρατώντας αλόβητο τον ισχύοντα γεωργικό προϋπολογισμό. Θα πρέπει το κάπα της κοινή γεωργικής πολιτικής να κρατήσει το νόημά του και στο μέλλον. Ναι, η αυτάρκεια δεν σημαίνει ε, κατάργηση ή έλλειψη των εμπορικών συναλλαγών. Γιατί παγκοσμιοποίηση σημαίνει εμπόριο, σημαίνει εμπορικές ε, συναλλαγές. Παρακαλώ το συντονιστή μας τον κύριο Σιμό να κάνει μια ανακεφαλαίωση για να μπορέσουμε σε λίγο να περάσουμε στο δεύτερο πάνελ. Oh, Συγγνώμη, κύριε Ντόρφμαν, θέλετε και εσείς το λόγο για να σχολιάσετε αυτά που είπαν ε, οι συνάδελφοι, ίσως αργότερα. Πρώτα να ακούσουμε τη σύναψη του κυρίου Σιμών. Voilà. Bon, je vais pas essayer d'apporter une conclusion. Δεν θα προσπαθήσω να διατυπώσω εγώ οριστικά. Συμπεράσματα είναι πολλά τα ερωτήματα που ετέθησαν. Διότι πρώτον θέλω να επιτρέψω ξεκινώντας από τον κύριο Ντόρφμαν, ο οποίος μας σε τέσσερα λεπτά θα πρέπει να επιχειρήσει να δώσει απαντήσεις στις ε, πολυάριθμες ερωτήσεις. Σύντομα, βέβαια, κύριε Ντόρφμαν. Ναι και ευχαριστώ. Δεν τα χρειάζομαι όμως τα τέσσερα λεπτά. Δεν νομίζω ότι ήταν ε, στόχος της σημερινής συνάντησης τίποτα άλλο από το να ακούσουμε τις ανησυχίες των συναδέλφων από τα Εθνικά Κοινοβούλια, πράγμα το οποίο και πράξαμε. Με χαρά σημειώνω ότι πολλοί συνάδελφοι επισημαίνουν πως δεν επιδιώκουν την επανεθνικοποίηση της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής και ότι πρέπει να παραμείνει κοινή η γεωργική πολιτική. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει την κόκκινη γραμμή των συζητήσεων, στις, ε, ή μάλλον το μύτο της Αριάδνης των συζητήσεων στις επόμενους μήνες και εδώ στο Κοινοβούλιο. Δεν αλλάζει δηλαδή η βασική προσέγγιση. Η κοινή γεωργική πολιτική με ό,τι λαγές της επιφέρουμε θα πρέπει να παραμείνει κοινή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αναφέρθηκαν συχνά οι μειονεκτούσες ε, περιοχές. Βεβαίως και συμφωνώ, είναι ένα σημαντικό κομμάτι η πολιτική για τις ε, περιοχές αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να παραμείνει σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να διατηρηθούν στη ζωή Ακόμα και στις περιοχές που δεν έχουν τόσο ευνοϊκές συνθήκες να προσφέρουν. Ε, επίσης, ισότιμη ή ισοδίκαιη μεταχείριση είναι ένας όρος που ακούστηκε πολλές, ακούστηκε πολλές φορές. Βεβαίως, αντιλαμβάνομαι ότι κάποια κράτη-μέλη μπορεί να τον ερμηνεύουν διαφορετικά από κάποια άλλα είναι κάτι το οποίο οπωσδήποτε και εδώ στη συζήτηση του κοινοβουλίου, στο Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προκύψει και θα αναλυθεί περισσότερο. Αλλά πάντως νομίζω ότι πρέπει να μιλούμε περισσότερο για εξωτερική σύγκληση και άρα να αναπτύξουμε κριτήρια τα οποία θα επιτρέψουν μια εισοδική κατανομή των κονδυλίων. Έγινε επανειλημμένος επίσης λόγος για ένα ε, έντιμο εισόδημα, έντιμη αποζημίωση για τον κόπο στη γεωργική πολιτική. Βεβαίως ε, δεν κάνουμε πολιτική εισοδηματική, ε, ούτε είμαστε μια ένωση ευρωπαϊκή η οποία ζει μόνο μέσα σε κλειστά σύνορα. Είμαστε μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, είμαστε μεγάλη εξαγωγική δύναμη στον υπόλοιπο κόσμο και άρα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να μην στρεβλώνεται και ο ανταγωνισμός από τις δικές μας ε, επιλογές. Δεν πρέπει να γυρίσουμε σε μια πολιτική της αγοράς που θα έχει ε, ελεγχόμενες ή προστατευόμενες τιμές. Δεν είναι αυτό το μέλλον της κοινής πολιτικής. Για να ολοκληρώσω, δεν ε, είχα σκοπό να ε, δώσω απαντήσει σε όλε τι παρατηρήσει. Απλώ ε, θα επισημάνω για άλλη μια φορά ότι άκουσα με προσοχή όλε τι παρατηρήσει των συναδέλφων από το Εθνικά Κοινοβούλιο. Ο κύριο Πλάνκ έχει το λόγο τώρα. Θέλω και εγώ πολύ στο να δώσω μια συνοπτική, ένα συνοπτικό συμπέρασμα. Διαπιστώνω ότι η κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να συνεχίσει αυτή η λειτουργία που έχει τη υποστήριξη του εισοδήματο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αλλά ότι ταυτόχρονα έχουν πολύ μεγάλη σημασία και άλλοι τομεί. ο ρόλος του γεωργού στην ε, παραγωγή προσθέμενης αξίας, στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, ε, η παρουσία των νέων στη γεωργική δραστηριότητα, αλλά και γενικότερα την ε, ύπεθρο ε, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτά σημειώνω και σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος ευχαριστώ και τώρα εγώ διατυπώνω τα τελικά συμπεράσματα ή σχόλια αν θέλετε. Έχω στη διάθεση μου πέντε λεπτά. Η σχολια αν θελετε εχω στη πεντε λεπτα η συζητηση λοιπον ε, δείχνει κάποιε αποκλήσει που έχουμε διαπιστώσει και σε επίπεδο κυβερνήσεων, δια, ε, σχέση με τη διαφύλαξη του προϋπολογισμού της ε, Κουγουπού, με μια μικρή εξαίρεση σε σχέση με κάποιες χώρες του Βορρά. Ε, σύγκληση επίσης σε σχέση με την ιστορική και εξωτερική σύγκληση στις ενισχύσεις. Στην οικολογικοποίηση πάλι υπάρχουν κάποιε διαφοροποιήσει, δεν είναι αρκετή, είναι αρκετή παρά είναι μεγάλη. Άμεσες, ενισχύσει, ναι ή όχι, ε, περισσότερη ανάπτυξη της υπαίθρου με περισσότερες ενισχύσεις ναι ή όχι. Αυτέ ήταν οι αποκλήσει. Ωστόσο, διαπιστώνουμε ταυτόχρονα ότι όλοι συμφωνούν πω πρέπει να προχωρήσουμε στην απογραφειοκρατικοποίηση, Σαρδάμ, και ε, την ανάγκη για την χρήση του εργαλείου, γιατί αυτό είναι το νέο στοιχείο στις προτάσεις της Επιτροπής, της επικουρικότητας. Διερωτώμεθα λοιπόν αυτό θα μειώσει όντω την γραφειοκρατία ε, ή θα ε, την μετατοπίσει μόνο στις εθνικές αρχές ή μήπως αυτό οδηγεί τελικά ακόμα και σε στρεβλώσεις ανταγωνισμού. Εν όλο, διαπιστώνω ότι οι ομιλητές εδώ τάσσονται στο πλευρό της, του γεωργικού κόσμου, στηρίζουν την Κούγου που εν όλο, ίσως με μία μόνο εξαίρεση, Όλοι πιστεύουν ότι πρέπει να μην επιτραπεί να εξαρτηθεί ή να πέσει θύμα της υποχρεωματικής και ίσως και αναπόφευκτης διεθνοποίηση των συναλλαγών η γεωργική πολιτική, μάλιστα κατά μια χρονική στιγμή όπου η Ευρώπη προχωρεί σε σύναψη συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών. Τώρα που συζητούμε εμεί, μάλιστα, αυτή τη στιγμή που συζητούμε, ξεκινά ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Μερκοσούρ για τα λεγόμενα ευαίσθητα προϊόντα. Ένα ε, θέμα, ένα τομέα που όπως λέει και το όνομά του είναι ευαίσθητος ιδιαίτερα. Βεβαίως αυτό που μας ενώνει με όλες τις αποκλήσεις της θέσης μας είναι ότι θέλουμε μια ΚΑΠ για το μέλλον με τη διαφύλαξη του κοινωνικού ιστού και, ε, των ζωνών, και στις ζώνες της υπαίθρου και τη βελτίωση των συνθήκων ζωής αυτού του κοινωνικού ιστού. Αυτό ασφαλώς μας ενώνει οπωσδήποτε. Άλλο ένα σημείο που διαπιστώνω μας ενώνει είναι αυτό το εισοδήματος. Εισόδημα, δίκαιο εισόδημα το οποίο προσφέρει στον ε, γεωργό τη δυνατότητα να εξακολουθεί να παράγει μέσα στην αλυσίδα την επισητιστική καλά προϊόντα και που βεβαίως αφορά και εμάς, τους καταναλωτές, γιατί θέλουμε προϊόντα όχι μόνο απολύτως ασφαλή επισητιστικά, αλλά εμείς ως καταναλωτές απαιτούμε να είναι όλο και πιο ποιοτικά τα προϊόντα που καταναλώνουμε. Τα βιολογικά, παραδείγματι, που είναι στη μόδα. Αλλά θέλουμε και τη γεωργία ακριβίας, η οποία δεν θα ε, εισάγει στοιχείο ίχνο στοιχείο ή ουσία παρα, άλλη παρά μόνο από αυτές που χρειάζονται στην παραγωγή. Γι' αυτό λοιπόν ιδιαίτερα ο, η ποιότητα, η διαχείριση του κινδύνου, ο περιορισμός του κινδύνου είναι η προσέγγιση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βλέπουμε να γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια σε σχέση με τα εθνικά στρατηγικά σχέδια, γιατί περί αυτών πρόκειται τελικά και φαντάζομαι το αντιλαμβάνονται οι πάντε εδώ, θα έχουν κυρίαρχο ρόλο τα εθνικά κοινοβούλια, γιατί θα υπάρξει μεγάλη εκχώρηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων στα κράτη-μέλη. Δεν μπορούμε παρά να σας ευχηθούμε καλή δύναμη, σιδηροκέφαλη. Και μια σας βλέπω εδώ μπροστά μου, σας εύχομαι σιδηροκέφαλος και, και σε εσά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστούμε για τις ευχές σας. Και ευχαριστούμε για, τις, για την ανακεφαλαίωση. Ευχαριστώ τον κύριο Σιμών γιατί μας συντόνισε με ένα αντικειμενικό πνεύμα εξωτερικού παρατηρήτη τη συζήτηση και θα δώσω τώρα το λόγο στο δεύτερο δημοσιογράφο για γεωργικά θέματα που θα συντονίσει το δεύτερο πάνελ, αφού μας κάνει μια σύντομη εισαγωγή. Οπότε καλό τον κύριο Δημαύρο να καθίσει και μετά θα ακούσουμε το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης ε, Γεωργίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Γέζη Πλέβα, μετά την κυρία Γκυλέρα Γκαρσία, την πρόεδρο της Επιτροπής Άγκρη και στο τέλος τον κύριο Παντέρινγκ από την Ιρλανδική Βουλή. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε Σικέσκη. Μετά την εισαγωγή αυτή, να και αλλάζουμε πάνελ, όπως είπε ο Πρόεδρος, είναι σαν να περνάμε από το περιεχόμενο, από το τι, στο πώς, στη μέθοδο. Και στο επόμενο αυτό πάνελ θα μιλήσουμε για νέες δυνατότητες συνεργασίας, νέους τρόπους συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών για πολυτομεακή και πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, για επικουρικότητα. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν, ξεκινώντας, να συζητήσουμε και το πού αναλόγως βεβαίως Εθνικού ή Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θέτει ο καθένας το όριο μεταξύ δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και δράσης των κρατών μελών. Δύσκολο αυτό βέβαια να το πράξουμε χωρίς να έχουμε δει συγκεκριμένες προτάσεις επιτάπητος. Θα ήταν ενδιαφέρον όμω να ακούσουμε τις θέσεις σας. Εγώ ως δημοσιογράφος έχω μάθει να κάνω ερωτήσει και προτείνω λοιπόν τις ερωτήσεις μου και αν θέλετε μπορείτε να δώσετε απαντήσεις σε αυτά που θα σας ρωτήσω. Η πρόκληση λοιπόν βεβαίω, έχει να κάνει με την διαχείριση, με τη χρηστή διαχείριση και διοίκηση. Μία ΚΑΠ που καλείται όλο και περισσότερο να ικανοποιεί τα όλο και πιο πολυάριθμα και απαιτητικά, ε, τις πιο πολυάριθμες και απαιτητικές απαιτήσει των ε, πολιτών, θα πρέπει να δούμε το πώς μπορούν να υλοποιηθούν οι στόχοι για τους οποίους συζητήσαμε μέχρι τώρα. Αφενός μεν η επικουρικότητα επιτρέπει τη χρήση πιο ακριβών εργαλείων, πιο επακριβών εργαλείων για να φτάσουμε από το κοινοτικό επίπεδο σε επίπεδα που μέχρι τώρα ήταν πιο δυσπρόσιτα όπως οι παραδείγματι ζητήματα που έχουν να κάνουν με το έδαφος, το έδαφος που είναι πόρος μη ανανεώσιμος, ε, το έδαφος που δύσκολα μπορεί κανείς να το εντάξει σε μια κοινή προσέγγιση ή πολιτικές για την ε, υποστήριξη των νέων ή η εξέβρεση ενός κοινού ορισμού για το ποιος είναι ο ε, εν ενεργεία γεωργός που με δυσκολία εξευρέθη στην τελευταία μεταρρύθμιση και που ήδη τώρα πια ε, αποδεικνύεται πως δύσκολα είναι και εφαρμόσιμη, εφαρμόσιμος ο ορισμός αυτός. Ε, η επικουρικότητα πολλές φορές έχει αναφερθεί, ωστόσο είναι και ένας δρόμος γεμάτος στροφές και δυσκολίες και για την εσωτερική αγορά, γιατί είναι δύσκολο και να ε, ε, εισακουστούν οι θέσεις ε, των διαφόρων επιπέδων και βέβαια και των ευρωπαϊκών αρχών. Πώς λοιπόν θα γίνει αυτό και πού θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να εγγραφεί το όριο μεταξύ της κοινή προσέγγισης και της εθνικής προσέγγισης. Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι αυτή η επικουρικότητα, και αυτό αναφέρθηκε ήδη, Πώς λοιπόν αυτή η επικουρικότητα, αυτό νέο σύστημα εφαρμογής θα οδηγήσει σε πραγματική, σε γνήσια απλοποίηση για τη γεωργική εκμετάλλευση και επιχείρηση. Πώς μπορούμε να έχουμε μια αμοιβαία ωφέλεια και για τον γεωργό αλλά και για την κοινωνία. Γιατί δυστυχώς πολύ συχνά υπάρχει και ζήτημα ε, αμοιβαίας ε, συνεννόησης ή συναντήληψη, συναντήληψης πρόβλημα. Ζητάμε λοιπόν ε, με την νέα αυτή κοινή γεωργική πολιτική νέα πράγματα. Είναι περίπλοκη η κατάσταση εντωμεταξύ και στο διεθνές επίπεδο. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν χρησιμοποιήσει το μακροεπίπεδο με περιεχόμενο που ορίζεται σε ε, κοινό, ε, από κοινή απόφαση στο κοινό επίπεδο. Αλλά πώς αυτό θα υλοποιηθεί ε, στην κάθε περιοχή χωριστά, πώς θα συμβεί αυτό. Έχουμε τις ε, συμφωνίες της χιλι... του στόχους της χιλιετίας που μεταφράζονται σε συμφωνίες των Παρισιών. Στην υλοποίηση όμως τι θα γίνει. Και εδώ έχουμε να κάνουμε ως προς το περιβάλλον με μια ε, κίνηση από μηδενική βάση. Η κοινή γεωρική πολιτική όμως έχει παρελθόν, έχει 50 χρόνια ιστορία. Επομένως και ίσως να είναι αυτό το τελευταίο ερώτημα πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Το ερώτημα που θα πρέπει να θέσουμε λοιπόν αυτό το τελευταίο ερώτημα θα πρέπει να είναι από την ιστορία της ΠΑΚ, από το παρελθόν της ΠΑΚ, τι μπορούμε να φέρουμε και να διατηρήσουμε για το μέλλον. Και αντίθετα τι πρέπει να σβήσουμε και να αφήσουμε στο παρελθόν. Με τον Τζέσι Πλέβα που είναι ο Γενικός Γραμματέας ε, Διευθυντής ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την Γεωργία και Ανάπτυξη, με την κυρία Αγγιλέρα, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Πατ Ντιρίγκα, Πρόεδρο της κοινή Επιτροπής για τη Γεωργία, τα Τρόφιμα και την Αλία, Ντιρίγκ του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου θα γίνει αυτή η συζήτηση. Και ξεκινώντας, δίνω το λόγο στον Τζέρσι Πλέβα. Uh, <clears throat> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ και αξιότιμη βουλευτέ των Εθνικών Κοινοβουλίων, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Σικέρσκι για την οργάνωση αυτής της διακοινοβουλευτικής ε, συνάντησης και συζήτησης ε, για ένα τόσο σημαντικό θέμα και τόσο επίκαιρη στιγμή. Όπως είπε ο Επίτροπος Χόγκαν στην αρχική του μιλία, Θέλουμε φιλόδοξη και κοινή γεωργική πολιτική. Μια πολιτική που θα στηρίζεται η τρέχουσα πολιτική με βάση τους κανόνες και τη συμμόρφωση ε, το έχει παρατραβήξει και η ενιαία προσέγγιση για όλους έχει φτάσει στα όρια της ε, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη της απλοποίησης της πολιτικής και της ε, ενίσχυσης της αποτελεσματικότητάς και της αποδοτικότητάς της. Θα έχουμε καλύτερο έργο και καλύτερα αποτελέσματα για τους γεωργούς, το περιβάλλον και τους πολίτες μας, μόνο να αλλάξουμε τον τρόπο που οργανώνουμε την γεωργική μας πολιτική. Και χαιρετίζω την ευκαιρία που έχουμε να συζητήσουμε την οργάνωση και την εφαρμογή της ΚΑΠ σήμερα. Γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη της αλλαγής. Σήμερα η κοινή αγροτική πολιτική απορτίζεται από ένα μακροσκελή κατάλογο πολύ λεπτομεριακών κανόνων που θεσπίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η προσέγγιση όμως δεν λαμβάνει υπόψη την πολυμορφία της ε, Γεωργίας και τις κοινωνικο-οικονομικές ε, συνθήκες της Ευρωπαϊκής, ε, των διαφόρων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε, έχουμε μια μεγάλη περιπλοκή και όλο και αυξανόμενο όγκο εφαρμοστικών κανόνων, καταθυντηρίων γραμμών, εγγράφων και νομικών ερμηνεών που είναι απαραίτητες για να αντιμετωπιστεί η ανάγκη της απόλυτης ασφάλειας δικαίου σε ό,τι αφορά τον αριθμό των εξαιρέσεων που χρειάστηκαν για να ανταποκριθούμε στην μεγάλη πολυμορφία και διαφορετικότητα της γεωργίας και των κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων. Πώς θα αλλάξουμε λοιπόν την ΚΑΠ. Διαρωτηθήκαμε ποιος κάνει τι και με τον καλύτερο τρόπο. Ε, χάρη λοιπόν των γεωργών και των καταναλωτών μας και των πολιτών μας, πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την εφαρμογή της ΚΑΠ. Μπορούμε να ενισχύσουμε την επικουρικότητα και την αναλογικότητα στην κοινή γεωργική πολιτική. Πέρυσι, ε, είχαμε εκτενέστατες διαβουλεύσεις ε, με πάνω από 322 ε, προτάσεις πολιτών για το μέλλον της ΚΑΠ. Και αυτή η διαβούλευση ήταν η βάση για την ανακοίνωση που εκδώσαμε στα τέλη του προηγούμενου έτους. Θεωρούμε ότι ο νέος καταμερισμός των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών μεταξύ ευρωπαϊκού, εθνικού και περιφερειακού επίπεδου ήταν απαραίτητος. Ε, και έχουμε επινοήσει το νέο μοντέλο παράδοση, το νέο delivery model, όπω λέμε, στην εφαρμογή τη κοινή γεωργική πολιτική. Τι είστε όμω νέο μοντέλο παράδοση, νέο delivery model. Σημαίνει τα εξή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα θεσπίσει το πλαίσιο που χρειάζεται για να εξασφαλιστούν ε, τα κοινά επιτεύγματα και οι κανόνες που θα συμφωνηθούν μεταξύ Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσδιορίζουν τα εξή κοινού στόχου πρώτον. Κοινού στόχου όπως ε, την γεωρική συμβολή στο μετριασμό των κλιματικών αλλαγών, στην προσαρμογή στις αλλαγές ή στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας. Αυτή είναι μερική από τους κοινού στόχους. Δεύτερον, ε, ε, ευρύς μεταρρυθμίσεις που, παρεμβάσεις που θα ρυθμίζονται επίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή τι θα γίνεται με τα κονδύλια αποσυνδεδεμένη ε, εισοδηματική ενίσχυση, προαιρετική συνδεδεμένη ενίσχυση, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πληροφοριών. Τρίτον, και πάλι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βασικές προϋποθέσεις που θα θεσπίζονται καθώς και ένα πλαίσιο για τη διαχείριση των ταμείων, προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, τα, οι φορείς που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή της ε, ΚΑΠ, όπως οι φορείς πληρωμής ή το σύστημα Άγιαξ, οι συνθήκες ε, πληρωμής, κανόνες που εξασφαλίζουν τη συμβατότητα με τις συμφωνίες του ΠΟΕ για τη Γεωργία και ούτω καθεξής και γενικοί κανόνες για την αξιολόγηση των επιδόσεων, για παράδειγμα κοινοί δείκτες για τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο. Τώρα, τι θα χρειαστεί σε εθνικό επίπεδο. Τα κράτη-μέλη θα κάνουν τον επιμερισμό του πλαισίου και θα εξασφαλίσουν την εφαρμογή. Θα εκτιμήσουν ποιες είναι οι ανάγκες τους με βάση τους κοινού ε, στόχους, χρησιμοποιώντας, χρησιμοποιώντας κάποιες αναλύσεις ε, που ήδη κάνουν τα κράτη-μέλη στα πλαίσια των αναπτυξιακών τους προγραμμάτων και θα θεσπίσουν τα ειδικά μέτρα που χρειάζονται για την κατανομή των άμεσων ενισχύσεων, για παράδειγμα, για την υποστήριξη των νέων αγροτών. Επίσης, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προσδιορίζουν καταμετρήσιμους και αξιόπιστους στόχους για να εξασφαλίσουν αυτές τις επιδόσεις. Για παράδειγμα, μερίδιο γη σε σχέση με τα περιβαλλοντικά μέτρα ή μερίδιο της συμμετοχής των γεωργών σε οργανώσεις παραγωγών, για παράδειγμα. Επίσης, τα κράτη-μέλη θα προτείνουν σε ένα νέο στρατηγικό έγγραφο ε, και για τους δύο πυλώνες της ΚΑΠ με τίτλο «Το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ». Εκεί τα κράτη-μέλη θα εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουν στην εφαρμογή της ΚΑΠ. Και τώρα, έρχομαι στις κοινέ μας ευθύνες όλων των ενδιαφερομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ο νέος επιμερισμός των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων δίνει την ευκαιρία μεγαλύτερης συμμετοχής στον, στα εθνικά κοινοβούλια. Επίσης, δίνει ευκαιρία για τη λήψη μέτρων που θα ανταποκρίνονται στις τοπικές και περιφερειακές περιστάσεις. Μέσω διαβούλευσης με τους υφεροντούχου, για παράδειγμα, και για τους δύο πυλώνες της ΚΑΠ. Για τις επιτροπές παρακολούθησης, για παράδειγμα. Η πρόταση αυτή δίνει περισσότερες ευκαιρίες ώστε η εφαρμογή να είναι στόχοθετημένη αλλά και απλούστερη. Αλλά δίνει και περισσότερες δυνατότητες αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων που είναι ιδιαίτερα φλέγοντα σε πολλές περιφέρειες και περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη-μέλη και οι γεωργοί θα μπορούν να δρέψουν τους καρπούς της νέας προσέγγισης και του νέου μοντέλου. Θα έχουμε μια απλούστερη πολιτική ε, με λιγότερες λεπτομεριακές διατάξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με λιγότερες εξαιρέσεις. Και θα έχουμε μεγαλύτερη σαφήνεια σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Μια και οι κανόνες ε, και τα μέτρα, οι λεπτομεριακοί κανόνες και τα μέτρα θα θεσπίζονται σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Ένα άλλο πλεονέκτημα της νέας προσέγγισης είναι η μεγαλύτερη ελαστικότητα ε, για την εφαρμογή συνδυασμένων και στοχευμένων δράσεων που θα προσαρμόζονται στις τοπικές ιδιαιτερότητες και στις τοπικές ανάγκες και περιστάσεις. Αυτό θα δώσει μια επιπλέον ευκαιρία και δυνατότητα για καλύτερη στόχευση προς τα αποτελέσματα μέσω στρατηγικού προγραμματισμού, μέσω στοχευμένων δράσεων που θα υπόκειται σε καταμέτρηση των επιδόσεων. Τώρα, τι μηχανισμούς ε, και εργαλεία θα έχουμε στη διάθεσή μας για να διαφυλάξουμε τον κοινό χαρακτήρα της πολιτικής. Σίγουρα η διαφύλαξη του κοινού χαρακτήρα της αγροτικής πολιτικής ε, είναι σημαντική. Το συζητήσατε και σήμερα. Θα πρέπει να κρατήσουμε αυτό τον κοινό χαρακτήρα. Γι' αυτό και προτείνουμε κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες. Για παράδειγμα, το ενωσιακό πλαίσιο κανόνων που θα περιλαμβάνεται στη βασική πράξη. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει τα σχέδια, τα εθνικά σχέδια της ΚΑΠ. Τρίτον, θα έχουμε στενότερη παρακολούθηση της εφαρμογής των εθνικών σχεδίων με βάση τους κανόνες. Τέταρτον, διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση εντοπισμού σοβαρών προβλημάτων. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι δεν θα έχουμε λιγότερες δράσεις, αλλά απλώ θα δρούμε διαφορετικά και θα δαπανούμε τα κονδύλια πιο στοχευμένα προκειμένου να έχουμε αποτελέσματα, ιδιαίτερα για το μετοριασμό των κλιματικών αλλαγών και για την προστασία του περιβάλλοντος. Το μοντέλο αυτό του παράδοσης, το delivery model, δεν θα μας κάνει το βίο το πιο περιπλοκό, αλλά πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Πλέμπα. Η κυρία Αγγελέρα Γκαρσία, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης Πέθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ κύριε Δημάμπρο. Και ε, θα ήθελα να απευθύνω θερμό χαιρετισμό προς ε, όλους τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων και τους συναδέλφους. Και επιτρέψτε μου, πριν περάσω στο νέο μοντέλο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στην ΚΑΠ, θα ήθελα να πω, μια και είναι παρούσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι συνήθως οι διάφορες κυβερνήσεις των κρατών μελών ζητούν ενίσχυση της ΚΑΠ, διαφύλαξη του γεωργικού προϋπολογισμού. Γενικώ είναι πολύ θετικά τα κρατημέλη απέναντι στην ΚΑΠ. Γι' αυτό όμως χρειαζόμαστε ένα πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο που θα είναι αξιόπιστο και που θα ε, δίνει έμφαση στο μέλλον και αυτή τη πολιτική και των άλλων πολιτικών. Μερικέ κυβερνήσει ήδη έχουν αποφανθεί προ αυτή την κατεύθυνση, άλλε όχι. Δεν μπορούμε λοιπόν να ζητάμε από τα κράτη-μέλη να κρατήσουν αλόβητο τον προϋπολογισμό της ΚΑΠ όταν, η Ευρωπαϊκή όταν δεν είναι διατεθειμένα να ενισχύσουν τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το λέω τώρα γιατί καλό θα ήταν μέσω των Εθνικών Κοινοβουλίων να, να επεκταθούν τα κράτη-μέλη και σε αυτή τη συζήτηση. Γιατί θέλουμε να διαφυλάξουμε την ΚΑΠ, αλλά για να κρατήσουμε την ΚΑΠ και να διαφυλάξουμε το μέλλον της και τον κοινό της χαρακτήρα, θα πρέπει να αυξήσουμε και τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η σημερινή συζήτηση, αλλά σίγουρα η ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, οδήγησε σε αλλαγή του ρόλου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Δημιουργήθηκαν ε, μηχανισμοί συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων με στόχο την εξασφάλιση του πιο αποτελεσματικού δημοκρατικού ελέγχου της ενωσιακής νομοθεσίας και της εθνικής νομοθεσίας σε όλα τα επίπεδα. Οι διατάξεις της συνθήκης της Λισαβόνας ε, ενίσχυσαν αυτή την τάση. Αυτή η νέα μορφή συνεργασίας ε, μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα, ε, πραγματώνεται μέσω τέτοιου συνεδριάσεων σαν τη σημερινή. Βέβαια, τα Εθνικά Κοινοβούλια και στο παρελθόν είχαν συζητήσει ελάχιστα την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Και Πολλές φορές τα κοινοβούλια δεν γνωρίζουν, ή δεν γνωρίζουν ακόμη τι προτείνουν οι κυβερνήσεις τους στο Συμβούλιο. Λόγω της ε, έλλειψης διαφάνειας δημοκρατικής που ισχύει σε τέτοια θέματα. Γιατί είναι αδιανόητο οι εθνικοί βουλευτές ε, να μην γνωρίζουν τις προτάσεις που θα υποβάλει η κυβέρνησή του στο Συμβούλιο. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τη δημοκρατική διαφάνεια. Στη συζήτηση που έγινε για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας, κάτι που συζητήσαμε νωρίτερα, έφτασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έφτασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάποια έγγραφα με τις θέσεις της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Φιλανδίας, της Ιρλανδίας, της Λιθουανίας και της Σουηδίας και ένα κοινό έγγραφο τεσσάρων χωρών της Ιρλανδίας, Πολωνίας, Γαλλίας και Ιταλίας. Οι υπόλοιπε χώρε, ακόμη και η δική μου Ισπανία, η πατρίδα μου Ισπανία, δεν έχουν καταθέσει κανένα έγγραφο με τις εθνικές τους θέσεις. Από ό,τι λέει η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στόχος ε, της νέας ΚΑΠ είναι η απλοποίησή της. Και μάλιστα πολλοί συνάδελφοι νωρίτερα μίλησαν για την ανάγκη της απλοποίησης. Χρησιμοποιείται η ενισχυμένη επικουρικότητα μάλιστα για να ενισχυθεί αυτή η απλούστευση. Θα δούμε αν ε, θα ισχύσει όντω κάτι τέτοιο. Γιατί κάθε φορά που σχεδιάζουμε μεταρρύθμιση ζητούμε απλούστευση της ΚΑΠΑ. αλλά μέχρι τώρα δεν τα έχουμε καταφέρει να την απλουστεύσουμε. Για να δούμε αν αυτή τη φορά θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί και θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, γιατί οι στόχοι μας είναι ίδιοι, στα αποτελέσματα χωλένουμε. Πέραν της απλούστευσης μέσω ενισχυμένης επικουρικότητας, ε, θα πρέπει να βελτιώσουμε τις τοπικές συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους στα πλαίσια των κοινών στόχων που θα θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, με την συναπόφαση Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Ένα βασικό στοιχείο της ανακοίνωσης προβλέπει ότι η προσέγγιση του ενίου μοντέλου για όλους δεν θεωρείται πια κατάλληλη εν ώψη της πολυμορφίας των γεωργικών μοντέλων και της ε, πληθώρας ε, των συνθήκων άσκησης της γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε η μελλοντική ΚΑΠ θα έχει κοινούς στόχους ε, και μέτρα κατάλληλα, αλλά τα κράτη-μέλη θα αποφασίζουν ποια είναι τα κατάλληλα μέτρα που ανταποκρίνονται στι ιδιαιτερότητέ και στις ανάγκες τους Η ανακοίνωση έχει ένα στοιχείο που λέει 24 μέσα αναφοράς για τα κράτη-μέλη. Τα περισσότερα αναφέρονται στο ρόλο που θα διαδραματίσουν στην, κατά την εφαρμογή της ΚΑΠ. Το νέο μοντέλο της εφαρμογής ε, της ΚΑΠ, το delivery model που μας παρουσίασε ο κύριος Πλέβα, θα στηρίζεται στα αποτελέσματα που θα επιτυχάνονται μέσω των εθνικών στρατηγικών σχεδίων, όπως μας είπε ο κ. Πλέβα. Αυτό όμως είναι για μας προς το παρόν άγνωστο σχή. Πρόκειται για ένα νέο μοντέλο. Το delivery model είναι καινούριο. Όλα δείχνουν ότι αν εστιαστούμε περισσότερο στα αποτελέσματα θα βελτιώσουμε τα αποτελέσματα. Το μοντέλο όμως αυτό είναι καινούριο. Θα πρέπει να εμπιστευτούμε δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι ότου υποβάλει τις συγκεκριμένες προτάσεις μεταρρύθμισης στα τέλη του Μαΐου. Θα πρέπει λοιπόν να δείξουμε εμπιστοσύνη σε αυτό το καταμερισμό των αρμοδιοτήτων και να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα της νέας, ΚΑΠ, της νέας πρότασης για την ΚΑΠ. Ο φόβος μας είναι η πιθανή επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ και η πιθανότητα συγχρηματοδότησης των άμεσων ενισχύσεων, γιατί ίσως αυτή η δυνατότητα περιληφθεί στον πρώτο πυλώνα. Για, τον για το Ευρωπαϊκό όμως Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Γεωργίας, μια τέτοια πιθανότητα, δηλαδή συγχρηματοδότηση των άμεσων ενισχύσεων στον πρώτο πυλώνα, θα ήταν απαράδεκτη, γιατί είναι σαν να ανοίγουμε την πόρτα στην επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ. Η ενισχυμένη επικουρικότητα του νέου μοντέλου προβλέπει υπευθυνότητα αρμοδιότητα των κρατών μελών για το πώς και πότε θα επενδύουν τα κονδύλια της ΚΑΠ και πού. Και θα πρέπει επίσης να προσδιορίζουν τα κράτη-μέλη τους τελικούς δικαιούχους των ενισχύσεων. Πολύ συχνά μιλούμε για το μοντέλο και την προσέγγιση. Αναφέρονται τα ιστορικά δικαιώματα, αναφέρονται η ενεργεία αγρότες. Αλλά ποιος θα είναι ο τελικός δικαιούχος θα είναι η απόφαση του κράτους μέλους τελικά. Οπότε, ανάλογα με τους υποχρεωτικούς και προαιρετικούς στόχους, κάθε χώρα θα είναι ελεύθερη να αποφασίζει το μοντέλο για τους δικαιούχους των ενισχύσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια κρίσιμη απόφαση που λαμβάνουν πια τα κράτη-μέλη. Επίσης, κάθε κράτος θα πρέπει να θεσπίζει το εθνικό στρατηγικό σχέδιο με τις ε, παρεμβάσεις και των δύο πυλώνων. Για να δούμε πώς θα λύθει το πρόβλημα της, ε, του επιμερισμού αρμοδιοτήτων, γιατί χώρες όπως Ισπανία, Γερμανία ή Ιταλία ε, αναγνωρίζουν συνταγματικά περιφερειακές αρμοδιότητες για τη γεωργία. Οπότε, να δούμε πώς ενταχθούν αυτές οι περιφέρειες και οι αρμοδιότητες τους στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο. Επίσης, ο δεύτερος πυλώνας να δούμε πώς θα καθορίζεται με συμμετοχή των περιφερειών και πώς θα ενταχθεί η πρότασή τους στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο. Ίσως εδώ λοιπόν να ανακύψουν σημαντικά νομικά ζητήματα σύγκρουσης αρμοδιοτήτων μεταξύ περιφερειών και, και, κεντρικής κυβέρνησης. Επίσης, ε, τα κράτη-μέλη θα αποκτήσουν πιο πρωταγωνιστικό, πρωταγωνιστικό ρόλο στα πλαίσια του ελέγχου και της συμμόρφωσης στα πλαίσια της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Έτσι και τα Εθνικά Κοινοβούλια στο μέλλον θα αποκτήσουν πιο πρωταγωνιστικό ρόλο. Έτσι θα πρέπει να γίνει, γιατί αν ε, τα περισσότερα κριτήρια για την υλοποίηση των αποτελεσμάτων γίνονται σε εθνικό επίπεδο, τα εθνικά κοινοβούλια, δηλαδή η φωνή και η ψήφος των πολιτών, όπως απεικονίζεται στο Εθνικό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να εισακούγονται. Επίσης, ε, τα κοινοβούλια θα ενημερώνονται για τα αποτελέσματα των ε, γεωργικών συμβουλίων, αλλά θα δίνουν τη γνώμη τους και για τα εθνικά στρατηγικά σχέδια. Βέβαια, οι συνομιλητές θα είναι τα κράτη-μέλη και η Επιτροπή, όπως μέχρι σήμερα, αλλά από πολιτική άποψη είναι λογικό να σκεφτούμε ε, πώς θα αναθεωρούνται τα εθνικά στρατηγικά σχέδια ε, και πώς θα εξετάζονται και αυτός ο έλεγχος και η αναθεώρηση καλό θα είναι να γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Ναι μεν οι συνομιλητές θα είναι η κεντρική κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον καθορισμό του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου. Αλλά από πολιτική άποψη θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ανάμειξη και των εθνικών κοινοβουλίων στην αναθεώρηση, την, την εκτίμηση και την αξιολόγηση αυτών των εθνικών στρατηγικών σχεδίων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Αγγίλερα Καρσία. Πατ Ντίριγγ, πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Γεωργίας Τροφίμων Αλίας του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου. Δέκα λεπτά έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, εξότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Εθνικών Κοινοβουλίων. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, τη δυνατότητα που μας δίνεται να εξετάσουμε τη δυνατότητα συνέργειας στο πλαίσιο αυτής της πολυεπίπεδης κυβέρνησης. Στο πλαίσιο της επικουρικότητας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα εθνικά τα κράτη-μέλη ε, και τα εθνικά κοινοβούλια έχουν ξεχωριστού διακριτού ρόλου οι οποίοι θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι. Η στόχοι είναι κοινοί. Να έχουμε υψηλή ποιότητα τρόφιμα σε προσιτές τιμές, αλλά ταυτόχρονα να, να ε, προστατεύσουμε και το περιβάλλον. Να προσπίσουμε το εισόδημα των αγροτών και να υποστηρίξουμε μια οικονομική ε, δραστηριότητα η οποία είναι κρίσιμη σημασία για την περιφέρεια. Όπως γνωρίζετε, η επικουρικότητα είναι ε, το, η συζήτηση για το σε ποιο σημείο της διακυβέρνησης, ποιο είναι ο καλύτερο εκείνο που θα μπορεί να εφαρμόσει ένα συγκεκριμένο μέτρο. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν σε ποιο επίπεδο χρειάζεται να εφαρμόζεται μια πολιτική για να είναι πλέον αποτελεσματική. Θα πρέπει επίσης να είναι ξεκάθαρο ποιος το πράττει αυτό και με ποιον τρόπο διαπιστώνουμε ότι με τη νέα ΚΑΠ τα κράτη-μέλη θα έχουν μεγαλύτερη ευελιξία, μεταξύ μεγαλύτερε δυνατότητε. Αυτό είναι μια ευκαιρία και ένα κίνδυνο, γιατί θα πρέπει να φροντίσουμε η εφαρμογή τη ΚΑΠ να είναι ομοιόμορφη, να μην δημιουργηθούν προβλήματα κατακαιρματισμού που διαπιστώσαμε και επιλύσαμε στο παρελθόν, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και σεβασμό τη επικουρικότητα. Εμεί υποστηρίζουμε αυτόν τον διάλογο που ξεκινάει η Επιτροπή μα λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη αυτή τη νέα πρόταση που γίνεται για αυτή τη διαδικασία και για αυτή τη δομή. Θα υποβάλουμε τι ε, προτάσει μα, τι ε, παρατηρήσει μα. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει και μια ουσιαστική υποστήριξη και μια ουσιαστική εμπλοκή των Εθνικών Κοινοβουλίων στην ε, γενικότερη ευρωπαϊκή συζήτηση. Υπάρχουν διαφορετικέ προτεραιότητε σε κάθε κράτο μέλο. Και αυτό είναι ένα από του κύριου λόγου που υπάρχει η επικουρικότητα οι πολιτικέ αποφάσεις θα χρειαστεί να λεφθούν με ομοφωνία από 28 κράτη-μέλη, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στι διάφορε προτεραιότητες. Έχουμε δύο κύριους τομείς που, για τους οποίους μιλάει η ανακοίνωση του Νοεμβρίου. Ε, είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η τρόπος διαχείρισης της ΚΑΠ είναι κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ιρλανδία. Σε μέτρα Όπω, για παράδειγμα, πώ θα διασφαλίσουμε ότι οι επιδοτήσει θα φτάνουν σε πραγματικού αγρότε, πώ θα εξετάσουμε το ζήτημα του κάπινγκ, πώς, ε, ε, και, και άλλε ουσιαστικέ πολιτικέ αποφάσει. Αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να εξεταστούν σε, και σε, σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο. Πρέπει να δούμε λοιπόν με ποιον τρόπο μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις επιδοτήσεις έτσι ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ΚΑΠ για να περιορίσουμε την μεταβλητότητα των τιμών. Δεδομένη τη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωρίζουμε ποιε θα είναι οι επιπτώσει για την Ιρλανδία. Επομένω, είναι ακόμα πιο σημαντικό για εμά να ε, συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε η ε, διαχείριση τη ΚΑΠ να είναι αποτελεσματική περιοχές όπως η Ιρλανδία που, που, που ε, γειτονεύει, που έχει σύνορα με, την, ε, με το Ηνωμένο Βασίλειο, θα πληγεί περισσότερο. Ε, έχουμε επίσης μεγάλες ανησυχίες όσον αφορά τον τομέα της κτηνοτροφίας και των βοηδών που είναι ένα πολύ σημαντικό τομέα τη Ιρλανδική οικονομία. Και η συζήτηση που έγινε με τι χώρε με μα δίνει ένα ξεκάθαρο παράδειγμα. Πρέπει να βρίσκουμε έναν τρόπο με την ΚΑΠ να αντισταθμίζουμε τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργούνται σε κάποιου τομεί τη αγροτική οικονομία. Γνωρίζοντα ότι υπάρχουν διαφορέ ανάμεσα στι διάφορε περιοχέ και στου διάφορου τομεί τη αγροτική οικονομία. Εφαρμόζοντας όμως αυτά τα διαφορετικά μοντέλα, ε, δεν διαφωνεί κανείς, όλοι συμφωνούμε μάλλον, ότι έχουμε έναν κοινό στόχο και αυτός πρέπει να διασφαλιστεί. Έχουμε λοιπόν μια νέα κάρπη η οποία θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην εθνική συνεισφορά αλλά κρατώντας την ε, κοινή ε, προσέγγιση. Η... Τα μέτρα, για παράδειγμα, που συζητούνται για την ε, σύνδεση επιδοτήσεων για περιοχέ οι οποίε έχουν ιδιαίτερα αντίξωε συνθήκε, στι οποίε πρέπει να υπάρξει επιδότηση για την προστασία τη βιοποικιλότητα, είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Θα πρέπει να συζητήσουμε επίσης για τη θεσμική συνεργασία την πρόσφατα υιοθετήσαν διακήρυξη, η οποία αναφέρει ότι σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να εμπλέκεται η δημοσιοδίκηση στη διαχείριση της ΚΑΠ. Είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την επικορικότητα ο, το, ο τομέας του περιβάλλοντος είναι ένας τομέας στον οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε την επικουρικότητα ακόμα περισσότερο. Γιατί γνωρίζουμε ότι διαφορετικά κράτη-μέλη χρειάζονται διαφορετικά μέτρα για τη, να προσαρμοστούν στις τοπικές τους, ε, στις του τοπικού περιβάλλοντος. Την προηγούμενη εβδομάδα η Επιτροπή μας δημοσιοποίησε ένα έγγραφο με τον οποίο προσπαθεί να συνεισφέρει στον διάλογο που γίνεται για την κλιματική αλλαγή. Και πιστεύω ότι αυτή η κλιματική αλλαγή είναι η σημαντικότερη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μα τι τοπικέ ιδιαιτερότητε στον τομέα αυτό. Καλωσορίζουμε λοιπόν ότι η ανακοίνωση τη Επιτροπή αναφέρεται στην επικουρικότητα, στο κεφάλαιο που αναφέρεται στην κλιματική αλλαγή και τη σχέση τη με τον ΚΑΠ. Έχουμε την εμπειρία με την οικολογικοποίηση και διαπιστώσαμε μέσω αυτή ότι η προσέγγιση που προσπαθεί να εφαρμόσει το ίδιο μοντέλο παντού δεν λειτουργεί. Ε, θα πρέπει να βρούμε τι λύσει εκείνε οι οποίε είναι πιο πιθανό να οδηγήσουν σε λύσει σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Χωρί αυτό βέβαια να κατακαιρματίζει την, την ΚΑΠ και του κοινού μα στόχου ε, ο τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτό ή προτείνεται να γίνεται αυτό την Επιτροπή είναι τα στρατηγικά σχέδια δάση. Η Ιρλανδία, όπως γνωρίζετε, έχει μια πολύ σημαντική, στην Ιρλανδία έχει μια πολύ σημαντικό ρόλο η καινοτομία στον αγροτικό τομέα. Δεδομένου ότι δεν έχουμε βαριά βιομηχανία, είναι ο σημαντικότερο τομέα τη οικονομία μα. Γι' αυτό η συνεργασία και η καλή λειτουργία του τομέα αυτού έχει κεντρική σημασία για τη χώρα μα. Ποιο είναι ο ρόλο λοιπόν των Εθνικών Κοινοβουλίων. Γνωρίζουμε ότι θα έχουμε τα στρατηγικά σχέδια, θα πρέπει να τα παρακολουθούμε, να, να, να ελέγχουμε την εφαρμογή του. Πέραν από αυτό, δεδομένου ότι με βάση την επικουρικότητα θα λαμβάνονται και εθνικά μέτρα, τα εθνικά κοινοβούλια θα είναι εκείνα που θα ελέγχουν την θέσπιση αυτών. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι θα αυξηθεί ο ρόλο των κρατών μελών. Αυτό σημαίνει όμω ότι πρέπει να αυξηθεί ταυτόχρονα και η λογοδοσία και η ουσιαστική παρακολούθησή του. όπως για παράδειγμα στην, την, είχαμε μια πολύ καλή συμμετοχή της Ιρλανδίας στις συζητήσει για τις ποσοστώσεις στην Αλληλεία, κάτι αντίστοιχο φαντάζομαι ότι μπορεί να συμβεί και στην κατάρτιση των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΑΠ. Ε, εξάλλου, με βάση την Ιρλανδική νομοθεσία, η κυβέρνηση ενημερώνει πάντοτε το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο για οποιαδήποτε ε, ε, νομοθετική πρωτοβουλία στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητείται από το Κοινοβούλιο να υποβάλει ε, γνωμοδότηση. Μία από τις επιλογές είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβλέπει την ε, εφαρμογή των στρατηγικών ε, πλάνων από τα κράτη. Όμως, πέραν από αυτήν την παρακολούθηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι και τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να παρακολουθούν την υλοποίηση των στρατηγικών ε, σχεδίων, καθώς επίσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ανταλλάξουμε βέλτιστες πρακτικές μεταξύ μας γιατί με αυτόν τον τρόπο θα βελτιώσουμε και την εφαρμογή της ΚΑΠ και την εξέλιξη της στο μέλλον. Συμπερασματικά, διαπιστώνουμε ότι η νέα προτινόμενη ΚΑΠ θα δημιουργήσει μεγαλύτερη ευελιξία, μεγαλύτερη δυνατότητα να προσαρμόζουμε την πολιτική στις τοπικές συνθήκες. Για να λειτουργήσει το να λειτουργήσει αυτό είναι ακριβώς αυτό που όλοι επιδιώκουμε, που όλοι επιθυμούμε και ε, θα παρακολουθήσουμε με μεγάλη προσοχή αυτή την προσπάθεια. Eh, eh. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τζίρινγκ. Ξεκινούμε τη συζήτηση την οποία θα κατευθύνει ο πρόεδρος Σικέσκη. Πρόεδρε, ευχαρι... ο πρόεδρος ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Όφεντορφ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να εκπροσωπήσω στη συζήτηση τους βουλευτές από τη Γερμανία. Όντως ήταν ε, πολύ καλή αυτή η ιδέα, η ανακοίνωση. Έχουμε την ε, εντύπωση ότι ο Γιώργος δεν φοβάται τίποτε περισσότερο από το, την, ε, τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαίνεται να επανέρχονται αυτοί οι έλεγχοι. Σε λίγο καιρό ανοίγει πάλι η περίοδος και φοβούνται πάρα πολύ οι γεωργοί μας. Το ζώο εδώ και χρόνια αισθάνονται ότι είναι στο δόλιο του κατηγορουμένου πριν καν ανοίξουν το στόμα τους. Έτσι λοιπόν η κατάσταση. Τα κρατήδια <clears throat> κατακλείζονται από υπερβολικούς ελέγχους, υπερβολική ρύθμιση με κόστος σε κάθε ευρώ μέχρι και 87 λεπτά του ευρώ. Είναι δυνατόν να πούμε σήμερα ότι έχει νόημα να συνεχίζεται αυτή η επιβάρυνση η γραφειοκρατική. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Πρέπει να ξανασχεδιάσουμε τις λύσεις μας με τρόπο πιο αναλογικός προς τα αποτελέσματα. Και πάνω απ' όλα πρέπει να κερδίσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των γεωργών στη γεωργία και τη γεωργική πολιτική. Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι και η κοινωνία έχει όλο και μεγαλύτερη απόσταση από αυτό το οποίο αντιμετωπίζει ο Γιώργος πάλι πρόβλημα και η επικοινωνία και η κατανόηση, η αλληλοκατανόηση. Νομίζω ότι σε αυτό θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε να κατανοήσει ο ένας τον άλλον. Και η κοινωνία, το Γεωργό και ο Γεωργός στην κοινωνία. Η κυρία Φωνσέκα έχει το λόγο. Από την Πορτογαλία. Ευχαριστώ. Όντως, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με την επικουρικότητα. Γιατί αν παραενισχυθεί, ίσως οδηγήσει σε επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ. Αλλά αν υποβαθμιστεί υπερβολικά, ίσως οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Αναφέρθηκαν οι κλιματικές αλλαγές και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει επικορικότητα στη μετριασμό τους. Για τις χώρες του Νότου, όπως η Πορτογαλία, το νερό ε, έχει θεμελιώδη ρόλο. Θα πρέπει να είναι επιλέξιμες οι επενδύσεις ε, σε αρδεύσιμες καλλιέργειες, γιατί αν δεν είναι επιλέξιμες θα έχουμε τεράστια στρέβλωση ανταγωνισμού εις βάρος της Πορτογαλίας και εις βάρος των άλλων μεσογειακών χωρών. Επίσης, στα πλαίσια της επικουρικότητας, μετά ε, δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις κατεξουσιοδότηση πράξη της να ε, καταργεί τις προηγούμενες συμφωνίες για το τι είστε επιλέξιμο και τι όχι όπως αναφέρθηκε πολύ εύστοχα, η ΚΑΠ δεν περιορίζεται μόνο στη γεωργία. Θα πρέπει να προσέξουμε και την αγροτική ανάπτυξη και επενδύσεις στην Ήπεθρο, ε, ακόμη και γύρω τους γεωργούς, να χρηματοδοτούνται από την ΚΑΠ. Οι επενδύσεις όμως που δεν γίνονται από τη γεωργία για την Ήπεθρο, τα κράτη-μέλη να αποφασίζουν από ποια κονδύλια θα χρηματοδοτούνται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό κυρίως για τις χώρες που η χρηματοδότηση της ΚΑΠ ε, είναι ανεπαρκής για τις ανάγκες και τη δυναμικότητα των χωρών αυτών. Σε ό,τι αφορά την απομάκρυση του γενικού πληθυσμού από τη γεωργία και την εχθρότητα που επικρατεί μερικές φορές ε, απέναντι στους γεωργούς, θα πρέπει να αναδείξουμε το ρόλο της γεωργίας και των γεωργών, όχι μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για το, τα δημόσια αγαθά και για την ασφάλεια των τροφίμων θα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί το, το κοινό. Επίσης, ε, από τη δημόσια διαβούλευση είδαμε πολύ διαφορετικές απαντήσεις ε, ανάλογα από το αν κάποιος προερχόταν από τη γεωργική κοινότητα ή ήταν άσχετος με τη γεωργία. Γι' αυτό και θα πρέπει να κάνουμε μια εξτρατεία συνειδητοποίηση του Εβραίου κοινού για το ρόλο της και τις πολλαπλές λειτουργίες της γεωργίας. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Εράς Καρσία. Νομίζω ότι ένα σημαντικός ρόλος της ΚΑΠ είναι η ενίσχυση του γεωργικού κλάδου. Και φυσικά αυτό προϋποθέτει μια εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Θα πρέπει φυσικά να υλοποιηθούν και κάποιοι στόχοι, όπως μας είπε ο Επίτροπος θα πρέπει πρώτα απ' όλα να εξασφαλίσουμε την ηλικιακή ανανέωση στη Γεωργία και να καταστήσουμε προελκυστικό τον τομέα για τι νέε γενιέ. Αλλιώ θα μείνουμε χωρί Ευρωπαϊκή Γεωργία και κτηνοτροφία. Ήδη για την ενέργεια εξαρτώμαστε από τι αγωγές. Δεν θα πρέπει τέτοια εξάρτηση να επεκταθεί και στα τρόφιμα. Επίση, να βελτιωθεί η γραφειοκρατία, να μειωθεί η γραφειοκρατία και να γίνουν πιο εύκολε οι διατυπώσει για του γεωργού για την πρόσβαση στα κονδύλια τη ΚΑΠ. Επίση, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τη μελλοντική μεταρρύθμιση της ΚΑΠ για να ενισχύσουμε την κοινή γεωρική πολιτική και να την καταστήσουμε ομοιόμορφη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί καλό είναι με να έχουμε υπόψη από περιβαλλοντική άποψη της περιφέρειας και την κλιματολογική, τοπογραφική, περιβαλλοντική τους πραγματικότητα. Αλλά δεν έχουμε εδώ ε, μια πολιτική αλακάρτο που ο καθένας θα διαλέγει ότι τον βολεύει. Γιατί αυτό είναι ο κίνδυνος να αποδυναμωθεί η ΚΑΠ και ο καθένας να λέει ότι θα συγχρηματοδοτήσει ένα τμήμα μόνο. Λέμε όχι στην συγχρηματοδότηση, όχι στην επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ και λέμε ναι σε μια ισχυρή και ομοιόμορφη κοινή γεωργική πολιτική. Σίγουρα το Brexit ε, θα συνεπιφέρει μεγάλους ε, οικονομικούς κινδύνους και προκλήσεις. Χάρηκα όμως ε, για κάτι που είπε ο πρόσωπος τη πολωνική Βουλή και που το λέμε εδώ και χρόνια στην Ισπανία. Εδώ και χρόνια η Ισπανία ζητά αύξηση της εθνικής συνεισφοράς στον γεωργικό προπολογισμό. Το 1,10 είναι ε, καλό για να λύσουμε ένα πρόβλημα του χρηματοδοτικού κενού, αλλά θα ήθελα και τα υπόλοιπα κοινοβούλια να ζητήσουν από τι κυβερνήσει να κάνουν μια προσπάθεια για την αύξηση τη εθνική συνεισφορά αν θέλουμε χρηματοδότηση της ΚΑΠ θα πρέπει να βρούμε και πόρους και θα το κάνουμε βελτιώνοντας και ενισχύοντας, αυξάνοντας την εθνική συνεισφορά στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Έτσι πιστεύω ότι θα διατηρήσουμε μια ισχυρή και ομοιόμορφη ΚΑΠ αποφεύγοντας την επανεθνικοποίηση που αν υλοποιηθεί θα ε, καταργήσει σε λίγα χρόνια τη γεωργία από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Είναι σημαντικό να έχουμε μια αποφασιστική πολιτική ε, απέναντι στη μεταρρυθμίση αυτή. Μερικές ε, χώρες έχουν μεγαλύτερα προβλήματα γιατί όπω η δική μου θα πρέπει να συμφωνήσουν με τις ε, αυτόνομες περιφέρειες αλλά θα πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Ένα φλέγον ζήτημα για την Ισπανία είναι τα ιστορικά δικαιώματα, τα ιστορικά κριτήρια. αυτά τα θέματα όμως θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις και θα πρέπει να ληφθούν τώρα. ναι, κάποια χειροκροτήματα που ακούστηκαν μάλλον είναι ε, επιδοκιμασία τη λύση που προτείνατε για τα προβλήματα που επισημάνατε. Ο κύριο Πανέβιτς από την Κροατία. σα ευχαριστώ. Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ και αξιότιμη βουλευτέ από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Σας ευχαριστώ Ευχαριστούμε την Επιτροπή Γεωργίας για την οργάνωση αυτής της συνάντησης και χαιρετίζουμε αυτή την πρωτοβουλία για την διακοινοβουλευτική συζήτηση για τα θέματα της Γεωργίας. Θέλουμε η ΚΑΠ να γίνει ατμομηχανή περαιτέρω οικονομικής ανάπτυξης και να εστιάζεται σε αποτελέσματα με συγκεκριμένους στόχους και φυσικά με κατακόρυφη και οριζόντια ολοκλήρωση όλων των συνιστοσών. Και ποιο μπορεί να το κάνει καλύτερα αυτό, εμεί, οι εκπρόσωποι των, Εθνικ... των Εθνικών Κοινοβουλίων, οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί εμεί είμαστε ε, αυτοί που έχουν άμεση επαφή με του πολίτε και με του γεωργού. Εμεί μπορούμε να εκτιμήσουμε καλύτερα τα προβλήματα και να θεσπίσουμε τι κατάλληλε ευρωπαϊκέ πολιτικέ. Γι' αυτό και θα πρέπει να αναμειχθούν πιο ενεργά τα Εθνικά Κοινοβούλια στο διάλογο με την ευρωπαϊκή πολιτική. Με τέτοιε πρωτοβουλίε όπω η σημερινή και με τι δυνατότητε που δίνει η συνθήκη τη Λισαβόνα ε, με διακοινοβουλευτική συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και μάλιστα στα τέλη ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει την πρότασή της για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και την μελλοντική ΚΑΠ μετά το 2020. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω μια πρωτοβουλία της Κροατικής Βουλής που θα οργανώσει διάσκεψη για το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, στη διαμόρφωση της μελλοντική κοινή γεωργικής πολιτικής. Θα ήθελα να σας καλέσω λοιπόν σε αυτή τη διάσκεψη ε, της Κροατικής Βουλής όλου τους εκπροσώπου των ε, Επιτροπών Γεωργίας των Εθνικών Κοινοβουλίων και, της ε, και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στα τέλη Νοεμβρίου θα γίνει αυτή η διάσκεψη. Παρακαλώ λοιπόν και στις μελλοντικέ συνεδριάσεις να εμπλέκεται ενεργά τα Εθνικά Κοινοβούλια στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών γιατί από κοινού θα δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, οφείλει και δύναται ε, να βοηθήσει τους γεωργούς ε, στα σημερινά και στα αυριανά τους προβλήματος. Μπορούμε από κοινού να επιφέρουμε τις απαραίτητες αλλαγές, ε, γιατί είναι απαράδεκτο σε μερικές περιοχές της Ένωσης και κυρίως στις ανατολικές περιοχές της Ένωσης να έχουμε ε, γεωργούς που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή γεωργικές κοινότητες ε, που δεν ευημερούν. Ευχαριστώ τον πρόεδρο Σεκέσκη για τη διοργάνωση αυτής της συνάντησης και ελπίζω και στο μέλλον ε, να συνεργαστούμε και σας περιμένουμε στη διάσκεψη που θα οργανώσουμε στην Κροατική Βουλή για το μέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής και κυρίως το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής. Ευχαριστώ. Ναι, αλλά αν έρθουμε όλοι, αν ανταποκριθούμε όλοι στην πρόσκλησή σας, τότε θα έχετε μεγάλο πρόβλημα. Ο κύριος Μπόγκης από την ε, Λετωνία. γνωρίζουμε ότι οποιοδήποτε μοντέλο και αν επιλεγεί για την κοινή αγροτική πολιτική, χρειάζονται πόροι, χρειάζονται χρήματα. Εκπροσωπώ συχνά τους αγρότες. Προσπαθώ να περάσω τα προβλήματα των αγροτών στο κοινοβούλιο της χώρας μου, στη Λετωνία. Και γνωρίζω ότι τα προβλήματά τους είναι πολύ, πολύ άριθμα. Από το 2002 και μετά έχουν ξεκινήσει να αντιμετωπίζουν όλο και μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα. Εάν συνεχιστεί αυτή η τάση μέχρι το 2020, εκτιμάται ότι στη Λετωνία θα έχει μια απόδοση το εκτάριο 182 ευρώ, δηλαδή το 60% του μέσου όρου του ευρωπαϊκού οι άλλες χώρες της Βαλτική βρίσκονται σε, παρόμοια ε, μοίρα. Αυτά είναι στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα, προφανώ. Το 2009 έως το 2016 έχουν αυξηθεί οι αρρώσιμες γέες στη Λετωνία κατά 8% ε, μια αύξηση σημαντική για εμάς. Βέβαια, στο, στην Ευρώπη συνολικά, στο μέσο όρο είναι μείωση 3%. Ε, το, αυτή η εξέλιξη δεν είναι αποτέλεσμα από των δασών. Ε, συνεχίζουμε να έχουμε πολλά δάση στη Λετωνία, όμως τα τελευταία 17 χρόνια ε, αξιοποιήθηκαν γέες οι οποίες κατά το παρελθόν δεν αξιοποιούνται. Στο όνομα λοιπόν των λεπτονών αγροτών και του Κοινοβουλίου ζητώ να διατηρηθεί η χρηματοδότηση της κοινή αγροτικής πολιτικής και την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο, να αυξηθεί μάλιστα η χρηματοδότηση των αγροτών, έτσι ώστε να συγκλίνουμε και εμείς με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σλάιερ. Eh, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Απάντω σε αυτό που νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Γερμανικού Κοινοβουλίου. Να ξαναρχίσουμε, να κάνουμε μια νέα αρχή, να έχουμε εμπιστοσύνη, να δώσουμε ένα στο χέρι στον άλλον. Κατά βάση συμφωνούμε. Εγώ εκπροσωπώ εδώ γεωργούς επίσης, που θέλουν μια δίκαιη ανταμοιβή για τους κόπους τους, που θέλουν να συνεχίσουν τις γεωργικές τους δραστηριότητες. Πιστεύω ότι πρέπει να το στηρίξουμε. Στην Ολλανδία κάνουμε το άπαν για να φτάσουμε στους στόχους μας, αλλά δεν μας ακολουθούν τα άλλα κράτη. Και συμφωνώ με τον κύριο Πλέβα, ε, πρέπει να ακολουθήσουμε ένα άλλο σύστημα. Μπορούμε να εργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη και τους στόχους του κλίματος, της κλιματικής αλλαγής τον περιορισμό των ε, νητρικών που έχουν ήδη καταστεί πολιτική στη Γερμανία και της αμμονίας. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια, ένα μεγάλο πολιτικό και νομοθετικό έργο. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να διατηρήσουμε τη δυνατότητα της ευελιξίας έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στην κυκλική οικονομία και οι γεωργοί μας για να επιτυγχάνονται οι στόχοι. Ιδάλλως, ο καθένας θα κάνει στη γωνιά του το δικό του, οι κατοχώρες Φερρυπίν, αλλά τελικά δεν θα κάνει κανείς ε, κάτι κοινό. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα... Ο Χάικο. Ρόλος των ε, εθνικών κοινοβουλίων ε, ενισχύεται με το εις νέες προτάσεις, ακόμα και των τοπικών κοινοβουλίων. Στην Πολωνία έχουμε ομόφωνα εγκρίνει την ε, υποστήριξη της κυβέρνησης στην προσαρμογή των πληρωμών. Όντως, συχνά λέγεται ότι πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση στις πληρωμές, αλλά αυτό <clears throat> δεν μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες διαφορές και αποκλήσεις μεταξύ των κρατών μελών. Πού πήγε η αλληλεγγύη. Χρειαζόμαστε λοιπόν αλληλεγγύη στο εισόδημα που θα προσφέρουμε στους γεωργούς μας. ...2,5 εκατομμύρια γεωργούς έχουμε στην γεωργία Ήδη έχουν όμως εγκαταλειφθεί πάνω από 100.000 εκμεταλλεύσεις, τεράστια απώλεια για την Πολωνία. Έχουμε κοινή πολιτική, κοινέ προδιαγραφές, κοινή γεωργική πολιτική, αλλά μετά υπάρχει ευελιξία προς την εφαρμογή μεταξύ κρατών μελών. Υπάρχει ανταγωνισμός και κάποιοι απαιτούν όλοι να τηρούν τις ίδιες προδιαγραφές, χωρίς όμως ίδια υποστήριξη. Ξέρουμε ότι από την, τον προπολογισμό της γεωργίας θα πρέπει να στηρίζονται περισσότερο οι γεωργοί από τα νέα κράτη-μέλη γιατί έχουν να καλύψουν το έδαφος το χαμένο σε σχέση με τα πλούσια κράτη της Δυτικής Ευρώπης και αυτό σημαίνει αλληλεγγύη. Um... Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ εκ μέρους της Ιρλανδικής Αντιπροσωπείας. Χαίρομαι ιδιαίτερος. μας απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα της πτυτικότητας των ε, τιμών. Πρέπει να δώσουμε λύσεις μέσα από την κοινή ε, γεωργική πολιτική για την αντιμετώπιση της πτυτικότητας των τιμών. Είδαμε στο γάλα μεγάλη πτυτικότητα τιμών και αυτό πρέπει να ενσωματωθεί στο σύστημα. Πάνω απ' όλα μας απασχολεί όμως ο όγκος του προπολογισμού και εμεί, ω Ιρλανδοί εξαρτώμεθα σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική δραστηριότητα της γεωργίας, είναι μεγάλο κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητα της χώρας. Ο προπολογισμό της Κουγουπού έχει στηρίξει σε δύσκολες στιγμές την ε, υπεθρό τη Ιρλανδίας και χρειάζεται στην Ιρλανδία ολόκληρη πρέπει για την Ιρλανδία ολόκληρη και την υπεθρότη ειδικότερα να διαφυλαχθεί ο προπολογισμό της γεωργίας, και πρέπει να συνεχιστεί η γεωργική δραστηριότητα. Χρειάζεται να ε, περάσουν οι νέοι γεωργοί στην γεωργική δραστηριότητα. Έχουμε γεωργούς άνω των 85 ετών ηλικίας. Πρέπει να αλλάξουμε γενιές λοιπόν και πρέπει μέσα από την κουκουπού να δώσουμε λύσεις για τους νέους γεωργούς για να γίνει αυτή η πολύ σημαντική εναλλαγή μεταξύ γενεών. Η νέοι γεωργία είναι απαραίτητη για την γεωργική οικονομία τόσο στην Ιρλανδία όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Ιδιαίτερη έμφαση λοιπόν πρέπει να δοθεί από την κουκουπού στους νεαρούς για να εξασφαλιστεί αλλαγή γενεών στη γεωργία. Γιατί αν αυτό δεν συμβεί, δυστυχώς κινδυνεύει ολόκληρος ο τομέας της γεωργίας και της υπαίθρου, κύριος Φλάνακαν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σημείωσα τα όσα είπαν οι δύο μιλητές από το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο. Και αυτό που υπόθηκε νωρίτερα για το ποιο έχει την καλύτερη θέση, τι συνθήκες υπάρχουν στα κράτη-μέλη, οι διαφορές μεταξύ κρατών μελών για την αναλλαγή γενναιών. Τώρα το ποιο βρίσκεται σε καλύτερη θέση νομίζω το βλέπει ο καθένα διαφορετικά από τη σκοπιά του. Αλλιώς η Ιρλανδία, αλλιώς το Συμβούλιο, στην αναλλαγή γενναιών στις συζητήσεις για τον κανονισμό Omnibus στην αρχή είχε προταθεί από το Συμβούλιο να πληρώσουν ε, υπό το νέο σχέδιο για την στήριξη των νέων γεωργών που έμεναν πάνω από πέντε χρόνια στην εκμετάλλευση τα κράτη-μέλη την ε, ενίσχυση για να ενισχυθούν ε, οι ε, δυνατότητες αναλλαγής γενναίας. τώρα, ωστόσο όμως το Συμβούλιο παρενέβη η Ιρλανδική κυβέρνηση για να αλλάξει τον υποχρεωτικό όρο θα από τον δυνητικό δύναται. Και αυτό άλλαξε τα πάντα σε σχέση με τη δυνατότητα υποστήριξης των νεαρών γεωργών. Αυτό είναι που μπορείτε να κάνετε για την Κουγουπού. Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί ελήφθη αυτή η απόφαση. Ήταν καταστροφική για τους νεαρούς γεωργούς και αν σας ένοιαζε η εναλλαγή γελαιών δεν θα την είχαν λάβει την απόφαση αυτή και, και δεν αναμένω καμία απάντηση. Πολύ θα ήθελα να ακούσω τι έχετε να πείτε. Παρακαλώ. Από τη Σουηδία. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ινγκφια, που μου δίνετε την ε, δυνατότητα να παρέμβω σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Για, την, για τους Σουηδούς, από την πλευρά της Σουηδίας θεωρούμε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αποκέντρωσης είναι θετική. Θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε πιο ξεκάθαρα αποτελέσματα με την αγροτική πολιτική. Πολλοί από τους συναδέλφους όμως ανέφεραν ότι υπάρχει ο κίνδυνος επανεθνικοποίησης. Για να αποφευχθεί αυτό θα πρέπει να εστιάσουμε στην ανταγωνιστικότητά μας ο, άλλοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στις δυσκολίες που μπορεί να δημιουργηθούν στον τομέα της οικολογικοποίησης, που αυτό είναι δύσκολο, λέει, να, ε, να προσαρμόζεται ε, στα, στις τοπικές ιδιαιτερότητες. Αντιθέτως, εγώ θεωρώ και θεωρούμε στη Σουηδία ότι τα τοπικού χαρακτήρα μέτρα είναι αυτά που θα δώσουν μεγαλύτερη εξουσία, μεγαλύτερε δυνατότητε στα κράτη-μέλη, να προσαρμοστούν στις συνθήκες τους, συμπεριλαμβανομένων και, στον τομέα, και του τομέα της οικολογικοποίησης. Μιλούμε για τη σημασία που έχει η αγροτική οικονομία για την κοινωνία. Θεωρώ ότι υπό τον δεύτερο πυλώνα μπορούμε να ε, χρησιμοποιήσουμε μέτρα τα οποία θα γίνουν καλύτερα αποδεκτά από τους καταναλωτές. Ε, ε, Ενώ για παράδειγμα την ενίσχυση της έρευνας που μπορεί να βοηθήσει στο να γίνει η αγροτική μας παραγωγή πιο αποτελεσματική, πιο ανταγωνιστική. Επίσης χρειαζόμαστε καλύτερο συντονισμό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και ε, χαίρομαι που διαπιστώσω ότι πολλοί συνάδελφοι ανησυχούν για τους ε, νέους αγρότες, για το πώς θα μπει η νεολαία στην ε, Γεωργία, πώς θα προσελκύσουμε νέους στον τομέα αυτό της οικονομίας. Όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να το επιδιώξουν αυτό. Όλα τα κρατη θα πρέπει να δημιουργήσουν ε, συνθήκες ε, που να επιτρέπουν στους νέους να ασχοληθούν με τη γεωργία. Και τέλος, με κάθε ε, τρόπο, σε όλα αυτά θα πρέπει να καταπολεμούμε τη γραφειοκρατία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σμίτα από τη Γερμανία. Κυρία συγγνώμη. Αποσιάζει. Η κυρία Πετήρα από την Κροατία. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπρόσωπο τη Κροατία. Ευχαριστώ. μου υπόψη ε, το, το πλεονέκτημα, το τι κάνουν για, τη, για τα τρόφιμα, για την ε, περιβαλλοντική βιοπικιλότητα, για την αξία, για την διαφύλαξη του οικογενειακού πυρήνα. Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα της γεωργίας μας ε, οδηγούν στην ε, ανάγκη να διαφυλάξουμε αλόβητα τη, ε, την γεωργική πολιτική και το γεωργικό προϋπολογισμό. Βέβαια θα πρέπει να είναι πιο απλοποιημένη, να φροντίσει ιδιαίτερα τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και επίσης να στηρίζει τους νέους αγρότες και να εξασφαλίζει την ηλικιακή ανανέωση. Δυστυχώς ούτε μία χώρα μέλος προς το παρόν δεν μπόρεσε σε, στα πλαίσια του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης να αξιοποιήσει τις δυνατότητες και να δρομολογήσει πρόγραμμα για την παρουσία των γυναικών στην Ήπεθρο. Γι' αυτό θα ήθελα να απευθύνω έκκληση προς τα Εθνικά Κοινοβούλια να παροτρύνουν τις κυβερνήσεις τους ε, να περιλάβουν και τις γυναίκες ε, στα υποπρογράμματα της αγροτικής ανάπτυξης. Οι κρότες γεωργοί περιμένουν απλοποίηση της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής, αλλά ακούσαμε και την ανάγκη απλούστευσης και για τη διοίκηση, όχι μόνο για τους γεωργούς. Γιατί ε, δεν θέλουμε με το νέο μοντέλο απλώ η γραφειοκρατία να, μετατρε... να μετατοπιστεί από το ευρωπαϊκό στο εθνικό επίπεδο. Φυσικά είμαστε υπέρ τη επικουρικότητα και τη ευελιξία, αλλά θα θέλουμε να παραμείνει κοινή η γεωργική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα τη αγορά, επίση, θα πρέπει η αντίδραση στι ε, διαταράξει τη αγορά ή η αντιμετώπιση των κρίσεων να γίνεται πιο άμεσα και να δίνεται δυνατότητα σε όλα τα κρατημέλη να συμμετέχουν. Και επίση στηρίζω την πρωτοβουλία που έχω προτείνει πολλές φορές και ο Επίτροπος Φιλ Χόγκαν υποσχέθηκε ότι θα την κάνει δεκτή να έχουμε ιδιαίτερο αποθεματικό κρίσεων που θα βρίσκεται εκτός της, του προϋπολογισμού της ε, κοινής πολιτικής. Ευχαριστώ. Ματίας από την Πορτογαλία. Ο κύριος ε, Ματίας από την Πορτογαλία αποσιάζει. Η κυρία Ντάλη. Ντέιλι μάλλον. Από την Ιρλανδία. Ο κύριος Σάνι. Ευρωβουλευτής. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. εξεπλάγει θετικά από τις αναφορές στο ρόλο και την ιδιαιτερότητα της ε, κοινή γεωργική πολιτικής, τη σημασία, τους για, τη της για τους ε, γεωργούς αλλά και για την κοινωνία γενικότερα. Ε, πιστεύω ότι για να καλύψουμε τα ελλείμματα ανάπτυξη στην Υπεθρό πρέπει να, γίνει αυτή, να προχωρήσει αυτή η λύση και σε επίπεδο δύο οργανικό. Αυτό που ανέφερε ο Επίτροπος με την ε, ε, λύση των έξυπνων χωριών, παραδείγμα, είναι πολύ χρήσιμη, γιατί ορίζει ήδη για την προσεχή ε, προγραμματική περίοδο κοινού κανόνες με βάση και τα ταμεία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλείας, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κυρίως ε, στόχευση στην Ήπεθρο ιδιαίτερα. Άρα λοιπόν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο μπορεί να στηριχθεί από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και συγκεκριμένα ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ορίσει ως υποχρεωτικό ένα 5% του συνολικού προϋπολογισμού των ε, ταμείων που εμπλέκονται στο σύστημα αυτών των, νέων των έξυπνων χωριών, ακριβώς για την ανάπτυξη της Ήπεθρου. Ε, πρέπει μικροί οικισμοί να μην αποκλειστούν από το σχήμα αυτό, από το σύστημα αυτό. Πρέπει να διαδραματίσουμε και εμείς το ρόλο μας, ε, αλλά και οι κυβερνήσεις πρέπει να υποστηρίξουν σε επίπεδο συμβουλίου τις προτάσεις αυτές και επίσης πρέπει να ενσωματώσουν στα αντίστοιχα εθνικά του συστήματα και σχέδια τα έξυπνα χωριά. Ο κύριος Ευχαριστώ. Οι συνάδελφοί μου από την Πολωνική Βουλή επισήμαναν την ανάγκη εξίσωσης των αμεσών ενισχύσεων ε, και μίλησε για την κυβερνητική πρόταση που έχει δεκτεί από όλα τα πολιτικά κόμματα στην Πολωνία. Επίσης, θα πρέπει να διαφυλάξουμε και το ισχύον σύστημα που οδηγεί ε, σε μεγαλύτερη απλοποίηση και μπορεί να είναι και εναλλακτική, ελκυστική εναλλακτική λύση, ε, ιδιαίτερα για, τα, για τις χώρες που δεν έχουν ιστορικά δικαιώματα για τις άμεσες ενισχύσεις. Σε ό,τι αφορά το νέο μοντέλο για την ΚΑΠ, το delivery model που μας παρουσίασε ο κ. Πλέβα, τα εθνικά στρατηγικά σχέδια δίνουν την ευκαιρία στα κράτη-μέλη να προσαρμόσουν τα μέτρα τους στις εθνικές ιδιαιτερότητες και στις εθνικές περιστάσεις. Επίσης, αυξάνεται η αρμοδιότητα των κρατών μελών στο σχεδιασμό, στην εφαρμογή και την υλοποίηση των στόχων της ΚΑΠ. Αυτή είναι μια νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ελπίζω να έχει θετικά αποτελέσματα. Συμφωνούμε με την πρόταση, αρκεί το νέο μοντέλο να είναι όντως απλούστερο ε, και να να δώσει την ευκαιρία για καλύτερη λήψη υπόψη των τοπικών αναγκών και ιδιαιτεροτήτων και των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών απειλών στις επιμέρους περιοχές. Υπάρχουν όμως και κάποια κίνδυνα από το νέο delivery model. Για παράδειγμα, καθυστέρηση στην εφαρμόγη της κοινή πολιτικής σε περίπτωση παράτασης της διαδικασίας εκπόνησης των εθνικών στρατηγικών σχεδίων. Γι' αυτό είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει μια ενορμονισμένη προσέγγιση απέναντι στα εθνικά στρατηγικά σχέδια και το νέο delivery model να επιφέρει όντως απλούστευση και να μην οδηγήσει σε αύξηση της περιπλοκής στην αύξηση των επιβαρύνσεων των εθνικών διοικήσεων και των διατυπώσεων για τις εθνικές διοικήσεις. Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προϋποθέτει και περισσότερους πόρους για, την, το σχεδιασμό εθνικών στρατηγικών σχεδίων, για την αξιολόγηση των σχεδίων, για την εφαρμογή τους, για τον έλεγχο της ε, εφαρμογής και για την καταμέτρηση και την αξιολόγηση της υλοποίησης των στόχων. Για παράδειγμα, ε, ε, περίπου 1.300.000 θα είναι οι δικαιούχοι, αλλά από διοικητική άποψη θα είναι, θα είναι απλοποιημένο το σύστημα, θα εποφεληθούν όντω οι γεωργοί, γιατί πολύ συχνά χρησιμοποιούμε τον όρο απλοποίηση, αλλά τελικά το τελικό αποτέλεσμα είναι πολύ πιο περίπλοκο. Ευχαριστώ. Τώρα ένα λεπτό μόνο στους υπόλοιπους. Ο κύριος Σταρκεβίτσιους, ένα λεπτό. Δυστυχώς μόνο ένα λεπτό από εδώ και πέρα. Σα Σας ευχαριστώ. Άκουσα ένα ξεκάθαρο μήνυμα σήμερα ότι ο προϋπολογισμός για την ΚΑΠ θα μειωθεί κατά 10%. Θα πρέπει να σκεφτούμε. Μήπως έχουμε κάποιο αποθεματικό, κάποια χρήματα που έχουν περισσέψει, παραμείνει από την τρέχουσα κοινή αγροτική πολιτική, τα οποία να μπορούν να αξιοποιηθούν. Πιστεύω ότι αυτό μπορεί να γίνει. Ας εξετάσουμε επίσης άλλα έργα τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν όχι μόνο την κοινή αγροτική πολιτική, αλλά και άλλες ευκαιρίες χρηματοδότησης. Με... Επίσης, ε, ας δούμε αν θα μπορούσαμε να μειώσουμε ε, έξοδα για τη δημοσιότητα, για παράδειγμα, ή άλλα περιτά έξοδα. Επίσης, πιστεύω ότι η απλοποίηση θα οδηγήσει σε οικονομία πόρων. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Απευθύνομαι στους ε, βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, για τον προϋπολογισμό που λέτε, που λέτε ότι ναι θέλετε να τηρηθεί ο προϋπολογισμός για τους ε, γεωργούς αλλά δεν θέλετε περισσότερα χρήματα να δώσετε. Ε, αυτό δεν γίνεται. Ιδάλλως, ε, αν δεν θέλετε ούτε το ένα ούτε το άλλο υπάρχει η τρίτη λύση να επιτρέψετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τους ιδίους πόρους. είτε είναι φόρος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είτε είναι φόρος κυριοζήνης. Υπάρχουν λύσεις για την γραφειοκρατία και την απογραφειοκρατικοποίηση. Ε, δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο πράγμα το να έχουμε μια καλή κεντρική διαχείριση και πολλή γραφειοκρατία. Αλλά από την άλλη, το να έχουμε 27 κράτη-μέλη που κάνουν διαφορετικά στη γωνιά του ο καθένα πάλι μπορεί να οδηγήσουν και σε γραφειοκρατία και σε στρέβλο ανταγωνισμού. Γιατί αν βάλουμε τρεις χώρες γειτονικέ οι οποίες στην εκτροφή των χείρων ορίζουν διαφορετικά όρια ως προς το ε, σε ποιο σημείο ξεκινούν οι ενισχύσεις μπορούμε πολύ ωραία να δούμε στρεβλώσει του ανταγωνισμού. Για τις ε, περιβαλλοντικές προδιαγραφές και το περιβάλλον και το κλίμα μπορούν να διαφυλαχθούν με βάση ισοδύναμους κανόνες. Κυρία Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που είμαι σε αυτήν εδώ και τόσο ζωντανή συζήτηση. Ελπίζω να μπορέσω και εγώ να προσφέρω κάτι σε σχέση με ιδέες για την απογραφειοκρατικοποίηση που τόσο συχνά αναφέρεται και ο χώρο της γεωργίας. Οπωσδήποτε μπορούμε να έχουμε πολύ πιο απλούς ε, κανόνες. Είναι μεγάλες οι προκλήσεις για τους γεωργούς ε, που έχουν να αντιμετωπίσουν και τους κινδύνους από τη διεθνή αγορά και τους κινδύνους που οφείλονται στο κλίμα, και τις καιρικές συνθήκες νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην διαφύλαξη από τους κινδύνους. Οι νέες τεχνολογίες επίσης μπορούν να μας προσφέρουν τεράστιες ευκαιρίες. και να ικανοποιήσουν το αίτημα του καταναλωτή για πιο οικολογικά, πιο καθαρά προϊόντα, για πιο καλά προϊόντα. Μπορούν επίσης νέες τεχνολογίες ή θα ήταν καλό, πιστεύω, νέε τεχνολογίε να ληφθούν περισσότερο υπόψη. Ευχαριστώ τελείω. Αλμπουκέρκη από την Πορτογαλία. Απουσιάζει. Ο κύριος Μπούντα. Ένα λεπτό μόνο κύριε Μπούντα όμως. Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα, πρόεδρε χρειάζεται να έχουμε, συμφωνούμε όλοι πάνω ότι χρειάζομαστε μια χρηματοδότηση η οποία θα παραμείνει στο ίδιο επίπεδο. Αλλά α είμαστε ξεκάθαροι. Μετά τον Brexit έχουμε λιγότερα χρήματα. Επομένω, εάν θέλουμε να κρατήσουμε το ίδιο επίπεδο χρηματοδότηση, πρέπει να πείσουμε όλοι ο καθένα ξεχωριστά την εθνική μα κυβέρνηση να συνεισφέρει περισσότερο στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Ε, διαφορετικά, ούτε ο κύριο Χόγκαν, ούτε ο κύριο Πλέβαν, ούτε κανένα δεν μπορεί να σα βρει ένα μαγικό ραβδάκι που θα βρει τα χρήματα για τη χρηματοδότηση τη ΚΑΠ. Δεύτερον, σύγκληση. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, όλοι επιθυμούμε μια ουσιαστική σύγκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όλοι ε, δραστηριοποιούμαστε στην κοινή αγορά. Έχουμε ελεύθερη κυκλοφορία ε, προϊόντων υπηρεσιών, έχουμε πλέον μια κοινή αγορά και στις χώρες στην Ανατολή και στις δυτικές χώρες. Επομένως θα πρέπει να πετύχουμε την πραγματική σύγκληση και τα ε, εθνικά κοινοβούλια πρέπει να πέσουν τον ρόλο τους. Ε, ορίστηκαν κάποιοι στόχοι στην αρχή, γεωργία, κλίμα, κλιματική αλλαγή, αφενός ανταγωνιστικότητα αφετέρου, πολλά άλλα θα μπορούσαμε να πούμε και το περιβάλλον πιο γενικά. Αλλά το θέμα είναι στον ανταγωνισμό και την ανταγωνιστικότητα Πώ εντάσσονται όλα αυτά. Και όταν μιλούμε για ανταγωνιστικότητα εννοείται ανταγωνιστικότητα μέσα στην ιστορική αγορά ή εννοείται στην παγκόσμια αγορά ανταγωνιστικότητα όπω αντιλαμβάνομαι εγώ. Και εκεί θα θέσω το εξή ερώτημα. Τι είναι πιο σημαντικό. Είναι πιο σημαντικό να συνεχίσουμε με τη στρατηγική μας για την παγκόσμια αγορά ή να διαφυλάξουμε το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Βεβαίω και μπορούμε να είμαστε σημαντικοί παράγοντε στην αγορά και πρωταγωνιστέ. Αλλά ταυτόχρονα μπορούμε να θέσουμε όρου για τη γεωργία σημαντικού που θα επιτρέψουν και στο γεωργό και την γεωργό να κάνουν τη δουλειά του σωστά. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία όμω πρέπει προκαταβολικά να λύσουμε. Ο κύριος Ροπέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για αυτή τη σημαντική ευκαιρία που μας δίνετε σήμερα να συζητήσουμε αυτά τα σημαντικά θέματα με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Όλοι γνωρίζουμε τη σημασία ε, της ΚΑΠ και πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα πολύ γρήγορα, πολύ σύντομα. Γιατί τη χρειαζόμαστε την κοινή αγροτική πολιτική, για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Έτσι ώστε το ε, ε, εισόδημα των αγροτών να διασφαλιστεί. Όταν έχουμε τους αγρότες να κερδίζουν το 50% σε σχέση με το μέσο εισόδημα ανθρώπων σε άλλους τομείς της οικονομίας, κάπως πρέπει να τους προστατεύσουμε. Ε, επίσης υπάρχουν τεράστιες ανισότητες ανάμεσα στα κρατημέλη και πρέπει να τις γεφυρώσουμε. κάτω για να έχει νόημα πρέπει να φροντίσουμε να ξαναγίνει κοινή αγροτική πολιτική. Εάν δεν έχουμε ένα δίκαιο σύστημα για τις επιδοτήσεις, δεν θα έχουμε ένα δίκαιο, ε, έναν δίκαιο ανταγωνισμό. Ε, και, και πιο σωστά μάλλον δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στον ανταγωνισμό από τις τρίτες χώρες. Κύριε Et même, si je puis dire, redite. Κύριος Κολομπιέ, διέκοψε ο πρόεδρος. Θα πρέπει να δούμε τρία ερωτήματα με ρεαλισμό. Πρώτα απ' όλα, πιστεύετε ότι εάν αποφασίζει η πλειοψηφία των κρατών μελών να κρατήσουν τις άμεσες επιδοτήσεις και τον πρώτο πυλώνα ή εάν ε, θα επιδιώξουν μία ουσιαστική μείωση των άμεσων απαιτήσεων. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Μετά, θέλουμε τις ε, ε, τομεακές ε, επιδοτήσεις να τις κρατήσουμε ή όχι. Και τρίτον, πώς θα υπάρξει μια συνέργεια, μια, μια, συνεργασία μεταξύ των κρατών όλων και ταυτόχρονα προστατεύοντας την συνεισφορά των Εθνικών Κοινοβουλίων σε όλη την διαδικασία αυτή. Ευχαριστώ. ως Κάφη, η συζήτηση που έχουμε είναι πολύ σημαντική και καλωσορίζω και χαιρετίζω μάλλον το γεγονό ότι έχουμε εκπροσώπους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Έχουμε σοβαρού χρονικούς περιορισμού. όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι όταν λέμε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ε, συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων στη χάραξη της ΚΑΠ, αυτό σημαίνει ταυτόχρονα ότι θα πρέπει οι προτάσεις να είναι και πιο ξεκάθαρες. Με άλλα λόγια. Πολύ συχνά λέγεται στους αγρότες ότι μια απόφαση ελήφθη στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν έχει καμία δυνατότητα να την αλλάξει η Εθνική Κυβέρνηση του Εθνικού Κοινοβούλιο και μετά ακούν ακριβώς το αντίθετο από τις Βρυξέλλες. Επομένως θα πρέπει να βρούμε μια φόρμουλα συνεργασίας με τους βουλευτές των κρατών μας έτσι ώστε αυτό που θα λέμε στους αγρότες να είναι ξεκάθαρο σε σχέση με το ποιο έχει αρμοδιότητα γιατί. Ευχαριστώ. Κυρία Χάζεκαμπ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα να ενισχύσουμε την επικουρικότητα, ιδιαίτερα για τις κατοχώρες. Συμφωνούμε με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις κατοχώρες η ποιότητα του νερού δεν είναι και πολύ καλή, εν μέρει και λόγω των λοιπασμάτων που χρησιμοποιούνται και έχουμε απανοτές εξαιρέσεις για την πατρίδα μου στον τομέα αυτό. Επίσης, δεν έχουμε σεβαστεί ούτε τους ευρωπαϊκούς κανόνες που θεσπίστηκαν για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Πώς ε, θα κάνει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν κανόνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί μερικοί δεν το κάνουν. Κυρία Κάντενμπαχ, ήθελα επί τη ευκαιρία να αναφερθώ ε, μια και είναι εδώ η εκπρόσωπη των Εθνικών Κοινοβουλίων σε μια σπουδαία ψηφοφορία που είχαμε σήμερα με τον συνελφό Μακάρθη για, για τη μικροβιακή αντίσταση και τους οργανισμούς εδώ λοιπόν συμφωνήσαμε και στο πώς θα πρέπει να προχωρούν τα θέματα της αντιμετώπισης μικροβιακής αντίστασης και στη γεωργία με, το, με την ιδέα του One Health, ενιαία υγεία. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να προωθήσουμε και σας καλώ να το υποστηρίξετε κι εσείς. Ε, σας ευχαριστώ λοιπόν όλους για τη συζήτηση αυτή την τόσο ζωντανή. Και πλούσια σε τοποθετήσεις. Τώρα πια όμως δεν έχουμε και τόσο χρόνο. Και γι' αυτό θα ήθελα να δω τι μπορούσαμε να πούμε στην ε, Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμείς, από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Γι' αυτό και καλό τον κύριο Πλέβα να λάβει το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ για την τόσο γεμάτη ενδιαφέρον συζήτηση. που λαμβάνει η χώρα και την κατάλληλη στιγμή, γιατί βλέπουμε την ανακοίνωση χωρίς όμως ακόμα να έχει κατεθεί η πλήρης πρόταση. Ε, γενικές γραμμές μόνο, γενική προσέγγιση δίνει η ανακοίνωση, πολλά θέματα παραμένουν. Πάνω απ' όλα με πείθει η συζήτηση ότι το μοντέλο που προτείνει η Επιτροπή ως μοντέλο υλοποίησης είναι η κατάλληλη προσέγγιση και παραδείγματι θα σημειώσω την αποφυγή των υπερβολικών ρυθμίσεων, την αντίληψη μεταξύ νέων γεωργών, γεωργών και γενικότερα της κοινωνίας, ε, οικονομική και κοινωνική αλλά και περιβαλλοντική ανταγωνιστικότητα, οικολογικοποίηση που δεν φέρνει αποτελέσματα στον πρώτο πυλώνα, πώς πρέπει να βελτιωθεί καινοτομία, έρευνα, ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία που έχει και αυτή την αξία της, λιγότερο περίπλοκες διαδικασίες, λιγότερη επιβάρυνση, ε, διοικητική αλλά και μετατόπιση από τις ευρωπαϊκές τις εθνικές αρμοδιότητες χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Όλα αυτά λοιπόν συμβάλλουν σημαντικά στη συζήτηση η τελική διαμόρφωση μιας πρότασης που θα είναι πολύ πιο λεπτομερής ασφαλώς. Και πιστεύω ότι θα δείτε με ικανοποίηση το τελικό κείμενο, το νομικό κείμενο που θα είναι έτοιμο στα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Θα είναι έτοιμο πριν τις νέες προτάσεις για το πολιτισμό νομικό πλαίσιο. Αλλά σχόλια για το πολιτισμό οικονομικό πλαίσιο δεν σκοπεύω να κάνω, όμως ήταν απόλυτα σαφής ο Επίτροπος για το θέμα αυτό. Θα είναι δύσκολο τώρα βέβαια να εκθέσω όλα τα σημεία στα οποία διατυπώνεται συνένεση σε κάθε τους λεπτομέρεια. Αλλά πάντως γενικά νομίζω μπορούμε να πούμε πως ένα νέο μοντέλο προστερές ε, ευθύνες και ευελιξία για τα κράτα ή μέλη και τις εθνικές αρχές υπό τον έλεγχο της Επιτροπής. Ένα μοντέλο δηλαδή το οποίο πιστεύω θα ικανοποιήσει και τον όρο της συνένεσης που αναφέρατε. Σταματώ εδώ διαβεβαιώνοντάς σας ότι σας ακούσαμε προσεκτικά, καταγράψαμε τις θέσεις σας Και βεβαίως θα δείτε τη συνέχεια στο, όταν κατατεθεί το κείμενο της πρότασης. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πλήβο. Η κυρία Αγγιλέρα για τις τελικές ε, παρατηρήσεις και τις συμπεράσματά της. Ευχαριστώ. Εγώ τηρώ ευλαβικά το χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Τρία σύντομα σχόλια γιατί ήταν εκτενέστατη συζήτηση. Και η συζήτηση μας έδειξε τη διαφορετικά σκοπιά, τη διαφορετική σκοπιά που υιοθετούν τα κράτη ανάλογα με το που βρίσκονται στο βορρά, στο νότο, στην Ανατολή, στη Δύση. Διαφορετικές οι θεωρήσεις, διαφορετικά τα μέτρα, διαφορετικά τα μοντέλα. Και σε αυτή την περιπλοκότητα και την ποικιλομορφία θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια κοινή αγροτική πολιτική και για το μέλλον. Το θέμα των νεαρών αγροτών ακούστηκε επανειλημμένο στη συζήτηση και λέμε είναι από τα σημεία που μας προβληματίζουν περισσότερο λόγω της ηλικιακή ανανέωσης. Είμαστε όμως έτοιμοι όλοι, τα Εθνικά Κοινοβούλια, Εθνικές Κυβερνήσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκήσουμε πραγματικά πολιτικές που θα εσωματώνουν και τους νέους γιατί ε, οι πολιτικέ ε, αυτές για, για τη συμπερίληψη των νέων δεν θα πρέπει να λαμβάνονται μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό. Και δεν γίνεται κάτι τέτοιο σε εθνικό επίπεδο. Και για να προκαλέσω περαιτέρω τη συζήτηση, είμαστε ε, διατεθειμένοι να μην ε, δίνουμε γεωργικές ενισχύσει από την ΚΑΠ σε ε, αγρότε που έχουν συνταξιοδοτηθεί. Είναι αυτά ιδέες για τη συζήτηση, για να δούμε αν όντως ε, ε, είμαστε σοβαροί ως προς την ανάγκη της ηλικιακή ανανέωσης και της ε, ενσωμάτωσης και των νέων στη Γεωργία. Κάποιος, νομίζω από τη Γερμανία, είπε ότι οι Γεωργοί φοβούνται πολύ τους ελέγχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Α, τώρα θα αρχίσουν να φοβούνται τους εθνικούς ελέγχους. Ε, γιατί οι έλεγχοι πια θα γίνονται στο εθνικό, σε εθνικό επίπεδο με βάση τα εθνικά στρατηγικά σχέδια. Και ο Παντήρινγκ έχει δύο λεπτά για να απαντήσει, να σχολιάσει. Θα είμαι σύντομο, κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω πρώτα απ' όλα ότι η συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα και με έπεισε προσωπικά ότι πραγματικά η επικουρικότητα μα δείχνει το δρόμο. Πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την αρχή. Γενικότερα, επίση, πρέπει να δούμε το ζήτημα τη ανανέωση των γενεών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κατά την άποψή μου και κατά την άποψη όλων μα στην Ιρλανδία, ένα από του σημαντικότερου τομείς, ε, μια από τις σημαντικότερες προσπάθειες πρέπει να γίνει είναι να προσελκύσουμε και νέους αγρότες και για να συμβεί αυτό πρέπει να έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Έτσι θα γίνει πιο ελκυστική η δουλειά για τους νέους και αυτό δεν ισχύει αυτή τη στιγμή. Γιατί υπάρχουν μια σειρά από προϋποθέσεις γραφειοκρατικές διαδικασίες που πρέπει να τις απαλείψουμε για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Ε, αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας στην ε, νέα αναθεωρημένη ΚΑΠ πρέπει, όπως σωστά αναφέρθηκε, να την κρατήσουμε κοινή την αγροτική πολιτική στο μέλλον. Τέλος, ε, κύριε Πρόεδρε, το ζήτημα των, πόρων. Κατά την ταπεινή μου άποψη. ο Πρωθυπουργό της Ιρλανδίας το ανέφερε τον Ιανουάριο ε, ότι και σας το αναφέρω ότι θα πρέπει οι δαπάνες οι ευρωπαϊκές να είναι ε, ε, στοχευμένες σε εκείνα τα προγράμματα τα οποία προχωρούν προς τα μπρος τα ευρωπαϊκά ιδεώδη. Με αυτό το γνώμο να πρέπει πιστεύω να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Σειρά μου τώρα, τρία λεπτά μου λέει ο πρόεδρος, αλλά θα είμαι και πιο σύντομος. Από τι παρατηρήσει που ακούστηκαν πιο συχνά, περισσότερο ρόλο για τα εθνικά κοινοβούλια, μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκών Αρχών και Εθνικών Κοινοβουλίων, περισσότερε ευθύνε για τα εθνικά κοινοβούλια. Έφτασε κάποιο μάλιστα να πει ότι με την υιοθέτηση και την έγκριση των προσεχών εθνικών σχεδίων προσεχή, στην προσεχή Κουγουπού, αλλά αυτό νομίζω έχει να κάνει με ευρωβουλευτέ εναντί εθνικών βουλευτών. Ακούστηκε λοιπόν η έκκληση προ του εθνικού βουλευτέ να ασκήσουν περισσότερε πιέσει προ τι εθνικέ του κυβερνήσει. Από τον Επίτροπο Χόγκαν όλο ακούστηκε αυτό για να ενισχύσουν τη συμβολή του στον προπολογισμό ε, τη γεωργική πολιτική, γιατί χωρί πόρου δεν μπορεί η Κουγουπού να προχωρήσει. Τέταρτη παρατήρηση, υπερβολική συγκέντρωση, όπω ε, σημειώνουν όλοι αποκέντρωση που θεωρούν όλοι θετική, ε, αλλά βέβαια ο καθένα την ερμηνεύει στη συνέχεια κατά το δικό του τρόπο. Ε, τα έξυπνα χωριά επίσης μπορούν να αποτελέσουν ένα κύτταρο χωρίς μικρόφωνο. Ε, ένα κύτταρο λοιπόν, ένα πρώτο εγχείρημα, ένα μοντέλο. Τι άλλο, ανέ, ναι, τα εθνικά σχέδια επανέρχονται διαρκώ στη συζήτηση, βοήθεια για τους νέους, ενισχύσει για τους νέους, καινο, νέους, καινοτομία περιβάλλον. Εν γέννη έμφαση στις, στην ευθύνη που δεν μπορεί και να αποκοπεί από την ευελιξία. Πάνε μαζί αυτά δύο. Επίσης, πρέπει να ενισχυθούν ε, και να διευρυνθούν οι επαφές μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκών Αρχών, ε, πολιετές πλαίσιο και μετά τον επόμενο μήνα περιμένουμε τις ε, προτάσεις για την κυρία Πολιτική. Αυτά από τα δικά μου συμπεράσματα και αφήνω το λόγο στον πρόεδρο Σικέρσκη. Εγώ, α, έχετε ακόμη ένα λεπτό. Δεν εξαντλήσετε το τρίλεπτο. Μπράβο σας. Λοιπόν, κοινή γεωρική πολιτική. Η κοινή γεωρική πολιτική δεν είναι μόνο πολιτική για τους γεωργούς, είναι πολιτική και για τους καταναλωτές. Γιατί αυτό θα πρέπει να γνωρίζει ο Ευρωπαίος πολίτης. Χάρη στην κοινή γεωρική πολιτική έχουμε φθηνότερα τρόφιμα για τους καταναλωτές, δηλαδή για εμάς όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Αλλά έχουμε ταυτόχρονα και την περιβαλλοντική πολιτική, την πολιτική για το κλίμα. Θα πρέπει να διαφυλάξουμε τη βιοπικιλότητα. Έχει πολλές λειτουργίες η κοινή γεωργική πολιτική επίσης ε, προωθεί συγκεκριμένες αξίες. Ε, αυτό θα πρέπει να αντιληφθούν ε, οι φορολογούμενοι και να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής πολιτικής. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους καταναλωτές, αφορά και τους πολιτικούς, γιατί τις αποφάσεις δεν συμβαίνει μόνο η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πόσο σημαντική είναι η κοινή γεωργική πολιτική, γιατί θα πρέπει να την διατηρήσουμε, γιατί σήμερα τα γεωργικά εισοδήματα είναι στο 40% των μέσων εισοδημάτων άλλων κλάδων, τι θα γινόταν αν δεν είχαμε καν την κοινή πολιτική, τι γίνεται με τις εξωτερικές επιπτώσεις, τους εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν την κοινή πολιτική. Ε, μερικοί κλάδοι της παραγωγής επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις εξωτερικές συνθήκες. Ή το εμπόριο, για παράδειγμα, επηρεάζει τη γεωργία. Είναι πολυδιάστατο λοιπόν το φαινόμενο. Επίσης, την απόφαση τελική ανάλυση την παίρνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει για τον προπολογισμό, α μην γελιόμαστε. Αλλά πολλά εξαρτώνται και από τι επιτροπέ γεωργίας. Συζητήστε με του γεωργού σα, συζητήστε με τι κυβερνήσει σα. Γιατί μπορούμε πολλά να κάνουμε για τη γεωργία και για το καλό των γεωργών. Ε, νομίζω ότι είμαστε όλοι από επιτροπές γεωργίας. Έχουμε παρόμοιες απόψεις, ε, εστερνιζόμαστε κοινέ αξίες, ε, μέρημνά μας είναι το καλό των γεωργών και η διαφύλαξη της γεωργίας. Και πρέπει να είμαστε γνώμων ε, προς τους γεωργούς για τις πολλαπλές λειτουργίες της γεωργίας. Γιατί αν δεν έχουμε γεωργικά εισοδήματα, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στην Ήπεθρο, αν δεν έχουμε νέους γεωργούς, ενισχύσεις που συνδέονται με την παραγωγή χρειάζονται σε μεγάλο βαθμό. Γιατί αν δεν στηρίξουμε την παραγωγή θα αφανιστούν κλάδοι ολόκληρη της γεωργίας στην Ήπεθρο. Μέχρι 15% των πληρωμών, των ενισχύσεων να συνδέονται με την παραγωγή. Γιατί πολύ συχνά χρειάζονται τέτοιες ενισχύσεις. Επίσης υπάρχουν διαφορετικοί όροι και οι άμεσες ενισχύσεις θα πρέπει να εξαρτώνται και από, το, από την ποιότητα του εδάφους, γιατί η ποιότητα του εδάφους έχει αποφασιστική σημασία στην αποδοτικότητα της γεωργίας. Αναφέρθηκε και το θέμα της ανταγωνιστικότητας. Επίσης, τα μικρομεσαία γεωργή, ε, η σταθεροποίηση των τιμών, γιατί η αστάθεια των τιμών ε, ταλανίζει τους γεωργούς επίσης ε, χρηματοδότηση και επιδοτήσεις. Για όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να συζητήσουμε και στη συνέχεια. Ήταν πολύ χρήσιμη η σημερινή ε, συνάντηση. Να λάβουμε υπόψη τις κρίσεις, τις θεομηνίες, ε, τις διάφορες προκλήσεις και τους κινδύνους, τη διαχείριση κινδύνου στη Γεωργία ευρύ φάσμα θεμάτων. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ευχαριστώ θερμότατα τους βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβούλια, ευχαριστώ θερμά τους ευρωβουλευτές, τους συνεργάτες, τους οργανωτές, όλους όσοι συνέβαλα στην σημερινή διοργάνωση. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος. Α, 6 παρα 5. Σας κάνω και δώρο ένα πεντάλεπτο, γιατί μέχρι τις 6 κανονικά είχαμε χώρο. Είδατε, τι ωραίο δώρο, πέντε ολόκληρα λεπτά. Ευχαριστώ λοιπόν όλους σας και ελπίζω να κρατήσουμε ακόμα το ηθικό και να κρατήσουμε αυτό το σφρίγος και τον ενθουσιασμό και στις επόμενες συζητήσεις. Περιμένουμε πάντως την νομοθετική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως μας είπε ο κύριος Γιέζη Πλέμα, Γενικός Διευθυντής. Οπότε πριν το τέλος της κοινοβουλευτικής θα ξαναβρεθούμε κύριε Πλέβα για να συζητήσουμε τις προτάσεις